Καλησπέρα σε όλους. Καθίστε παρακαλώ έτσι ώστε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Our chairwoman, Linda. Η πρόεδρος, κυρία Μακάβαν, θα αργήσει λίγο να έρθει. Όμως εμείς θα ξεκινήσουμε στην ώρα μας. Είναι μεγάλη μερίσια διάταξη, έχουμε να αποφασίσουμε για αρκετά θέματα και να ακούσουμε αρκετές πληροφορίες. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν αμέσως. Καταρχάς, Έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Έχετε λάβει την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη με την προσθήκη του σημείου 9 για την ανθρωπιστική κατάσταση και ανταπόκριση μετά τον σεισμό και το τσουνάμι στο Σουλαβέζι της Ινδονησίας. Θα έρθει εκπρόσωπο της ΓΔΕΛΤΑ ΕΚΟ έτσι ώστε να μας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις. Δεν έχω να προτείνω κάποια τροποποίηση στην ημερήσια διάταξη. Σας ζητώ λοιπόν να την εγκρίνουμε ω έχει. Υπάρχουν σχόλια. Όχι, σας ευχαριστώ πολύ. Ανακοινώσεις της Προέδρου. Αλλαγή εισηγητών. Η ομάδα του ΕΛΚ μας έχει ενημερώσει για μια αλλαγή εισηγητών για, ένα, για μία από τις εκθέσεις τους. Πρόκειται για τον Φρανκ Έγγελ, ο οποίος έχει αποχωρήσει από τη θέση του εισηγητή της γνωμοδότησης της Επιτροπής Ανάπτυξης για την ενδιάμεση έκθεση τη Επιτροπή προπολογισμού πάνω στο επόμενο πολιτεύσιο δημοσιονομικό πλαίσιο, την οποία γνωμοδότηση θα ψηφίσουμε σήμερα, θα τον αντικαταστήσει η Ζέλιανα Ζόβκο. Παρομοίω και για τη γνωμοδότηση τη Επιτροπή μα την έκθεση τη Επιτροπή Προπολογισμού για την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που θεσπίζει το νέο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο από το 2021 ω το 2027. Έπειτα, έχουμε δημόσια συζήτηση με την European Think Tanks Group. Να σας υπενθυμίσω λοιπόν την δημόσια ανταλλαγή απόψεων που φιλοξενούμε την επόμενη Τετάρτη 17 Οκτωβρίου με την European Think Tanks Group από τις 2.30 έως τις 5.30 με τη συμμετοχή των Bill Gates και Φεντερίκα Μογκερίνη. Το θέμα της ε, συζήτησης είναι η καινοτομία στην ανάπτυξη, το μέλλον της διεθνούς συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε ήδη λάβει το πρόγραμμα και την πρόσκληση για αυτήν την συνάντηση. Θα σας το θυμίσουμε όλες μέσα στην εβδομάδα. Μετά, θα λάβει χώρα και μία έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ανάπτυξης στο Στρασβούργο στις 12 Νοεμβρίου ώστε να ψηφίσουμε τις γνωμοδοτήσεις για τα δύο ε, θέματα σχετικά με τον ορίζοντα, τον κανονισμό δηλαδή και την απόφαση, καθώς και για την γνωμοδότηση της Επιτροπής μας, την έκθεση της Επιτροπής ΙΝΤΑ για την προσχώρηση της Σαμόα στην ενδιάμεση συμφωνία εταιρική σχέσης με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η συνάντηση αυτή θα διεξαχθεί από τις 9 μέχρι τις 10. Ήταν η μόνη ώρα που μπορούσαμε να κλείσουμε, δυστυχώς. Θα λάβετε το σχέδιο της ημερήσιας διάταξης εμπρόθεσμα και θα συνεχίσουμε με τις ανακοινώσεις της Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάποιες ανακοινώσεις για μας. Σας δίνω το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, προς ενημέρωση, Θα θέλαμε λοιπόν να ενημερώσουμε την Επιτροπή σας πως ε, η ΓΔ θα δημοσιεύσει τρία έγγραφα που σας ενδιαφέρουν τον Οκτώβριο. Ελπίζουμε να προλάβουμε. Ολοκληρώνεται η διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα τρία έγγραφα λοιπόν είναι καταρχάς ένα έγγραφο εργασίας για το Action Plan για τα δύο φύλλα. Έχει να κάνει με την ε, εφαρμογή. Έπειτα άλλο ένα έγγραφο εργασίας για την διατροφή και επιστημιστική ασφάλεια. Έγγραφο αποκλειστικά της Επιτροπής και ένα κοινό έγγραφο για την επιστημιστική ασφάλεια το οποίο εκθέτει την πρόοδο της Επιτροπής και, τα και των κρατών μελών πάνω στο θέμα αυτό. Με μεγάλη μας χαρά λοιπόν θα έρθουμε στην Επιτροπή για να σας παρουσιάσουμε τα έγγραφα αυτά και να συζητήσουμε. Επίσης, να σας ενημερώσω ότι η Αυστριακή Προεδρία θέλει να καταλήξει σε συμπεράσματα του Συμβουλίου και στα τρία αυτά έγγραφα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 26 Νοεμβρίου. Αυτά από εμάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Θα ήθελε κάποιος να σχολιάσει ή να κάνει κάποια ερώτηση. Όχι. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ. Move. Περνάμε στο σημείο 4. Θα συζητήσουμε για τους ε, στόχους βιώσιμης ανάπτυξης σχετικά με την υγεία και την εφαρμογή αυτών. Έχει έρθει η ώρα να εξετάσουμε τις ε, πρώτες τάσεις και προκλήσεις που έχουν αναδεθεί την τελευταία φορά που συζητήσαμε θέματα υγείας στην Επιτροπή μας ε, ήταν τον Απρίλιο σε συνδυασμό με διάφορες αποστολές και επίσης είχαμε συζητήσει με το Γενικό Διευθυντή του ΠΟΗ το Μάρτιο. για την ενδυνάμωση των συστημάτων υγείας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης αφορούν 30 στόχους και 28 δείκτες. Ωστόσο, η υγεία αφορά και άλλους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης και στους άλλους στόχους επίσης υπάρχουν πτυχές που αφορούν την υγεία. Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε το, τη διαφορά ανάμεσα στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και την πρόοδο που έχει σημειωθεί, έχουμε καλέσει τον Πίτερ Sands, εκτελεστικό διευθυντή του Παγκόσμιου Ταμείου την καταπολέμηση του AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας. Ο Πίτερ Σάντς είναι εμπειρογνώμων σε θέματα δημόσιας υγείας παγκοσμίω και μετά από σταδιοδρομία στον τραπεζικό τομέα διορίστηκε εκτελεστικός διευθυντής το Νοέμβριο του 2017. Επίσης, προσκεκλημένη είναι η Φάνη Φότσφινκλερ, επικεφαλής του Γραφείου της Ένωσης στην Global Health Advocates. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Πίτερ Σάντς. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πολύ τα μέλη της Επιτροπής που μας έδωσαν τη δυνατότητα να έρθουμε και να μιλήσουμε σήμερα για το ρόλο της ε, του Παγκόσμιου Ταμείου για την καταπολέμηση του AIDS, της Ελληνοσίας και της φυματίωσης ως μέρος των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης 3. Είμαστε ο μεγαλύτερος ε, παγκοσμίος χορηγός ε, δανείων στον τομέα της υγείας και ένας από τους ε, πολύ συγκεκριμένους στόχους των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης 3 είναι η καταπολέμηση του AIDS, της φυματίωσης και της ελαιονοσίας. Τρεις δηλαδή από τις πιο θανατηφόρες μεταδοτικές ασθένειες σήμερα. Το Παγκόσμιο αυτό ταμείο διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση των τριών αυτών ασθενειών. Είμαστε μετά το διμερές πρόγραμμα των ΗΠΑ ο δεύτερος ε, μεγαλύτερος χορηγός ε, χρηματοδότηση αυτών τον τομέα και για την φυματίωση, η οποία είναι η πιο θανατηφόρα από τις τρεις αυτές ασθένειες που ανέφερα, όπου διαθέτουμε το, και το 57% της παγκόσμιας χρηματοδότησης ε, για την καταπολέμηση της ελαιονοσίας. Κάθε χρόνο Μάλλον το 2017 χορηγήσαμε δάνεια ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στόχος μας είναι όχι μόνο να καταπολεμήσουμε την ασθένεια, αλλά να δημιουργήσουμε παγκοσμίω ικανότητες και υποδομές. Το σύνολο, το μεγαλύτερο μάλλον μέρος των επενδύσεών μας ε, πηγαίνει σε χώ, στις χώρες που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Όπως θα δείτε, το 65% της χρηματοδότησής μας πηγαίνει στις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. Η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο παγκοσμίω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη είναι οι μεγαλύτεροι συνεισφέροντες με περίπου το ίμιση της χρηματοδότησης. Κατά την ε, πέμπτη περίοδο του Ταμείου χορηγήθηκαν 475 δισεκατομμύρια ευρώ. Μόλις το Μάρτιο ανέλαβα καθήκοντα, αλλά τα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου μαρτυρούν ότι έχουμε σώσει τη ζωή 27 εκατομμυρίων ανθρώπων. Αυτό είναι ενδεικτικό της κλίμακας ε, που, κινείται, που κινούνται αυτές οι ασθένειες. Έχουμε διανύμει αντιρετροϊκά φάρμακα, εκατομμύρια, 197 εκατομμύρια δίχτυα προστασίας από την ελαιονοσία. Είναι ενδεικτικά τα νούμερα αυτά. Ο αντίκτυπος των δραστηριοτήτων μας είναι πολύ σημαντικό. Οι θάνατοι από ελαιονοσία μειώθηκαν κατά 40% τόσο και από AIDS. Το ποσοστό για την ελληνοσία είναι λίγο λιγότερο, είναι περίπου 20%. Γι' αυτό προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε την πολιτική ηγεσία για να αυξήσουμε τη χρηματοδότηση. Πριν από μερικές εβδομάδες έγινε και η συνάντηση υψηλού επίπεδου με αυτό ακριβώς το θέμα. Ο στόχος μας είναι απλώς να δοθεί ένα τέλος στις επιδημίες αυτές του AIDS, της φυματίωσης και της αλλονοσίας. Είναι ένας στόχος μακροπρόθεσμος, όμως αντιμετωπίζουμε και προκλήσεις. Γι' αυτό πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο αντιμετώπισης και να κινητοποιήσουμε περισσότερους πόρους. Επίσης, η έμφαση δεν θα πρέπει να είναι μόνο στο να δοθεί ένα τέλος στις επιδημίες, αλλά σε βιώσιμους στόχους. Αυτό για να επιτευχθεί χρειάζεται ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας. Το 27% των επενδύσεων του Παγκόσμιου Ταμείου πηγαίνουν στην οικοδόμηση ανθεκτικών συστημάτων υγείας. Ε, ασχολούμαστε με όλους τους τομείς των υποδομών αυτών, κατάρτιση επαγγελματιών υγείας, ε, υποδομές, πολιτική, προμήθειες και παροχή υπηρεσιών. Επίσης, επενδύουμε περίπου ένα δισεκατομμύριο δολάρια το χρόνο για να βοηθήσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες να δημιουργήσουν και να χτίσουν συστήματα υγείας. Αυτή η βοήθεια που παρέχουμε είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλον ε, οργανισμό που δραστηριοποιείται στον τομέα αυτών. Επίσης, κινητοποίηση εγχώριων πόρων. Απότερο στόχος είναι να έχουν τη δυνατότητα οι ίδιες οι χώρες να χρηματοδοτούν τα συστήματα υγείας. Γι' αυτό και προσπαθούμε μέσω διαφόρων μηχανισμών συγχρηματοδότησης, για παράδειγμα, να επιτύχουμε το στόχο αυτό. Είδαμε πως ε, πέρυσι υπήρχε 41% αύξηση χρηματοδότησης στην δημόσια υγεία και στόχος μας είναι μία αύξηση ακόμα 40% από το 2018 στο 2020. Εδώ βλέπουμε πως αλλάζει το παγκόσμιο σκηνικό. Βλέπουμε πως ε, για πρώτη φορά οι χώρες ε, της ε, Αφρικής χρηματοδοτούν το, την καταπολέμηση του AIDS με περισσότερους πόρους από ότι οι τρίτες χώρες. Έπειτα, δραστηριότητες ως προς τα δύο φύλλα. Υπάρχουν στοιχεία για τις νέες μολύνσεις από τον ιό HIV στις ε, γυναίκες και τα κορίτσια. Τα δεδομένα αλλάζουν. Ε, φαίνεται πως οι γυναίκες και τα κορίτσια, ιδιαίτερα οι νέες γυναίκες και οι έφηβες, είναι εκείνες που προσβάλλονται συχνότερα από τον ιό. Οι λόγοι είναι πολλοί, υπάρχουν μειονεκτήματα και ε, σε σχέση με το φύλλο και σε σχέση με την παιδεία. Είναι μεγάλες οι προκλήσεις ε, που συναντάμε όταν προσπαθούμε να προστατεύσουμε ένα, μια 15χρονη κοπέλα από τη μόλυνση, από τον ιό. Γι' αυτό και για όλες τις προσπάθειές μας θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη στήριξη που μας έχουν δείξει από την αρχή, διότι μιλάμε για μεγάλα χρηματικά ποσά που προέρχονται από τους φορολογούμενους, αλλά και ο αντίκτυπος είναι εξίσου μεγάλος. Το έργο μας δεν έχει ολοκληρωθεί βέβαια. Εάν όμως θέλουμε μέχρι το 2030 να δώσουμε ένα τέλος στην επιδημία αυτή, θα πρέπει να συνεχίσουμε να διαθέτουμε σημαντικούς πόρους και να βελτιωνόμαστε. Η επόμενη χρονιά θα είναι κρίσιμη για το Παγκόσμιο Ταμείο διότι θα περάσουμε στον έκτο κύκλο ε, χρηματοδότησης. Ε, είναι τριετής η κύκλη και ο πρόεδρος ε, Μακρόν θα προεδρεύσει στην Λιόν όπου και θα διεξαχθεί το συνέδριο. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ κύριε. Να δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Βόιτς Βίνκλερ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εργάζομαι για τους Global Health Advocates που εξετάζουν ιδιαίτερα τις διάφορες πολιτικές ανάπτυξης, ευρωπαϊκές πολιτικές έρευνας κλπ. για να δούμε πώς εφαρμόζει τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα κάνουμε σε συνεργασίες, συμμαχίες, υποβάλλοντας συστάσεις και υποδείξεις που έχουμε αναπτύξει μαζί με άλλους μη κυβερνητικούς οργανισμούς. Λίγα λόγια πρώτα για την εφαρμογή των στόχων ε, βιώσιμης ανάπτυξης σε ολόκληρο το επίπεδο της Ένωσης. Δεν υπάρχει μια στρατηγική ανάπτυξη. Αναμένει λοιπόν η κοινωνία των πολιτών στην πρόταση πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου να προτείνει την υλοποίηση της στρατηγικής ή να βάλει την Ατζέντα 2030 ως υπόβαθρο. Όμως η ΜΚΟ σε όλο το φάσμα είμαστε πολύ απογοητευμένες, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο έγγραφο προβληματισμού της για τους SDG που θα εκδοθεί φέτος τον Δεκέμβριο, δηλαδή τρία χρόνια μετά από την έγκριση των ε, στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και ε, κάποιους μήνες μετά από την κατάθεση του ΠΙΔΕΛΤΑΠΗ. Ω γνωρίζετε επίση, τον προηγούμενο μήνα, στην ομιλία του State of the Union, ο πρόεδρο Juncker δεν μίλησε για του ε, στόχου βιώσιμη ανάπτυξη. Δύσκολο λοιπόν να μιλήσουμε για υλοποίηση των SDG όταν δεν μπαίνουν μέσα στο πολιτικό πλαίσιο αυτή τη προσπάθεια. Επίση, στι νέε προτάσει ε, οικονομική ανάπτυξη, ούτε η εξάλληψη της φτώχειας, ούτε οι SDG περιλαμβάνονται ρητά στα σχέδια κανονισμών. Δεν είμαστε οι μοναδικοί που θεωρούμε ότι το πολιτικό αφήγημα βασίζεται σε σενάρια, σε σενάρια συμφερόντων. Και θα πρέπει ωστόσο να αλλάξει αυτό, γιατί βρισκόμαστε ήδη σε αντίφαση με την αποτελεσματικότητα της βοήθειας που έχει συζητηθεί επί δεκαετίες για το πώς θα γίνει η βοήθεια αποτελεσματική. Όλοι όσοι εργαζόμαστε στην ανάπτυξη σε τρίτες χώρες γνωρίζουμε ότι πρέπει να είναι αποτελεσματική η βοήθεια και για να είναι αποτελεσματική και βιώσιμη πρέπει να παρακολουθείτε και να εφαρμόζετε από τις ίδιες τις κοινότητες τις οποίες ωφελεί. Σε ό,τι αφορά τώρα την δημοσιονομική πρόταση, το θεματικό πρόγραμμα αναλαμβάνει το μεγαλύτερο βάρος. Από την midterm review όμως του εξωτερικού ε, μηχανισμού χρηματοδότησης μας βοηθούν να συμβάλλουμε σε γενικούς συνολικούς στόχους κατά πολέμηση ασθενειών επιδημιών για να βοηθήσουμε να φτάσουμε δηλαδή τους SDG. Στην παρούσα πρόταση έχουν πάρει το ελάχιστο 8% του συνολικού προϋπολογισμού σε σύγκριση με το 21% του τρέχοντος του δημοσιονομικού πλαισίου. Αναγνωρίζουμε την πρόσθετη αξία των γεωγραφικών προγραμμάτων και την ανάγκη να ευθυγραμμιστούμε με προτεραιότητες των χωρών, αλλά μας απασχολεί η μείωση κατά 54% του φακέλου ε, παγκοσμίων προκλήσεων διότι από εκεί θα προέλθει η χρηματοδότηση για πρωτοβουλίες όπως το Global Fund και άλλα. Και όταν λέω ότι αυτό έχει αποδειχτεί, έχει αποδειχτεί και σε διάφορε αξιολογήσει, αλλά και σε εξωτερικέ αξιολογήσεις που έχει δημοσιεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει αποδειχτεί η αξία του μηχανισμού αυτού και κατ' επανάληψη μάλιστα. Όταν εξετάζουμε τα γεωγραφικά προγράμματα, βλέπουμε ότι αγνοούνται οι κοινωνικοί τομεί. Εκεί λοιπόν θα αποκατασταθεί μια ισορροπία με τα θεματικά προγράμματα. Στο τρέχον ΠΔΠ μόνο 10% των ε, εθνικών ενδεικτικών προγραμμάτων, μόνο 10% δαπανώνται εκεί στην παιδεία. Εκεί χρειάζεται λοιπόν μια ισορροπία. Άλλο σημαντικό κίνδυνο για τη χρηματοδότηση τη προστασία τη υγεία είναι οι νέε προτεραιότητε των δωρητών, που τώρα πια είναι η μετανάστευση και η ασφάλεια και αγνοούν κάπως τις βασικές, τις θεμελιώδεις κοινωνικές υπηρεσίες. Η συγχρηματοδότηση άλλωστε αποτελεί απέτηση για να αποκτήσει κανεί τη χρηματοδότηση. Ακόμα και το IMF λέει ότι σε πολλές χώρες, για παράδειγμα στον Ήγερα, βρήκαν ότι οι δαπάνες για την ε, υγεία και την παιδεία έχουν υποκατασταθεί τώρα από άλλες δαπάνες που πηγαίνουν στην ασφάλεια. Ακούσαμε ταυτόχρονα, ε, προηγουμένως από τον κύριο Σάντς, ότι η επένδυση στο Παγκόσμιο Ταμείο παρακινεί και τις άλλες χώρες να κινητοποιήσουν και αυτές με τη σειρά τους περισσότερους σπόρους, εθνικά δηλαδή. Τώρα, για να έρθουμε λίγο στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τις παγκόσμιες αυτές πρωτοβουλίες. Το τρέχον πι το συνολικό, η συνολική χρηματοδότηση για τον ΚΑΒΗ, Vaccine Alliance, είναι 175 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό χρηματοδοτήθηκε από δύο φακέλους παγκόσμια ε, αντιμετώπιση προκλήσεων, δύο φάκελοι έφταναν τα 7,5 εκατομμύρια. Τώρα για τη νέα προτινόμενη αντιμετώπιση προκλήσεων, Global Challenge Envelope, έχουμε 3 εκατομμύρια. Αν δηλαδή βάλουμε ένα όριο, κάτι το οποίο δεν είναι και υπερβολικά φιλόδοξο, βλέπουμε ότι είναι το μισό. Και αν δείτε τώρα και το παράρτημα, θα δείτε άλλους 12 θεματικούς τομείς που θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από τον ίδιο φάκελο. Αυτό που ζητούμε εμείς είναι δύο πράγματα. Αν θέλουμε λοιπόν να έχουμε τη φιλοδοξία να φτάσουμε να υλοποιήσουμε το SDG 3, θα πρέπει πρώτα το Κοινοβούλιο, το οποίο διαπραγματεύεται την πρόταση SCI, να εξασφαλίσει αύξηση του συνολικού χρηματοδοτικού φακέλου για τις παγκοσμίες προκλήσει κατά τουλάχιστον 5 εκατομμύρια και την, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από τις ευρωεκλογέ, διότι δεν ξέρουμε μετά από αυτό τι είδου επιτροπή θα έχουμε, τι είδου κομισιόν θα έχουμε, να Ε, να εξασφαλίσει και να δεσμεύσει 508 εκατομμύρια για την ε, ε, βοήθεια αυτή. Χρειαζόμαστε περισσότερε πρωτοβουλίε για τη χρηματοδότηση, διότι η χρηματοδότηση αυτών των προκλήσεων μα επιτρέπει να συμμετέχουμε στο Συμβούλιο των Πρωτοβουλίων αυτών. Να συνεχίσουμε δηλαδή να διατηρούμε τι ευρωπαϊκέ μα αξίε. Στο παρόν πλαίσιο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ιδίω αν δούμε πού πηγαίνει τώρα ο Οργανισμό Ενωμένων Ω κοινωνία των πολιτών το ίδιο ζητούμε. Ζητούμε περισσότερα χρήματα για αυτέ τι πρωτοβουλίε. Ταυτόχρονα όμω θέλουμε να βρισκόμαστε και στο Συμβούλιο για να φροντίζουμε να υποστηρίζουν διαρκώ τι πρωτοβουλίε αυτέ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, λέει η Πρόεδρο. Ήρθε η ώρα τώρα να λάβουν το λόγο τα μέλη μα να ερωτήσουν ή να κάνουν σχόλια. Πρώτο ο κύριο Σάρλ Γκέρεν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ του δύο προσκεκλημένου, έναν κύριο, μία κυρία και ε, έθεσαν μια ερώτηση που ζητεί απάντηση, δηλαδή σχετικά με την χρηματοδοτική ικανότητα για την υγεία για τα επόμενα χρόνια. Είμαι ένας από τους συνεισηγητές για το νέο μηχανισμό, ε, νέο ενιαίο μηχανισμό και είναι ένα ερώτημα λοιπόν αυτό το οποίο θέτω και εγώ ίδιο στον εαυτό μου. Χρειαζόμαστε περισσότερους πόρους. Έχουμε συνολικά περισσότερους πόρους από ό,τι είχαμε για το 2021-2027 Έχουμε, μάλλον θα έχουμε περισσότερο για το 2021-2027. Η ιδέα της Κομισιόν ασφαλώς δεν ήταν να περιπλέξει τα πράγματα, ωστόσο, όπως και εσείς, ενδιαφέρομαι να λάβω απάντηση από τους υπευθύνους της Κομισιόν σήμερα σχετικά με τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουν τη χρηματοδότηση, ανάγκη χρηματοδότηση του 2021-2027. Από όσο γνωρίζω και σε ό,τι αφορά τον τρέχοντα μηχανισμό υπήρξαν μικτές χρηματοδοτήσεις από πλείονες πηγές. Μηχανισμός για τη γειτονία, μηχανισμός DCI και Ευρωπαϊκό Ταμείο Αναπτύξεως. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι, μπορεί να βασιστεί κανείς στην προβλεπτικότητα της Κομισιόν. Εγώ δεν έχω απολύτως κανένα λόγο και καμία διάθεση να καταδικάσω την Επιτροπή, αλλά δεν θέλω να υπάρξουν παρεξηγήσεις ό,τι αφορά την ορατότητα των πόρων που θα τεθούν στη διάθεση του Παγκόσμιου Ταμείου και των χρηματοδοτικών δράσεων στον τομέα της υγείας γενικά. Ξεκινώντας από τις τρέχουσες προτάσεις, δηλαδή πώς προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει επαρκώς τη χρηματοδότηση. Και δεύτερο, αρκετοί εδώ στην παρούσα Επιτροπή θεωρούμε, επιθυμούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνει πρωτοπόρα στην διάθεση πόρων. Στο παρελθόν, άλλωστε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε πάντοτε μια σημαντική επίδραση στους άλλους εταίρους της διότι δεν έκανε ποτέ, δεν έκανε ποτέ οικονομίες, πάντοτε ανακοίνωνε περισσότερα χρήματα από ότι τώρα. Και εν ώψη όμως του χρηματοδοτικού, ε, προβλέψεων τώρα θα θέλαμε κάποιες απαντήσεις από την Κομισιόν. Η Πρόεδρος, ορίστε παρακαλώ, η κυρία Ζαμπόρσκα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. A preto ma zaujímajú niektoré otázky, ktoré... Με ενδιαφέρει, ε, κυρία Ζαμπόρσκα, για, με ενδιαφέρουν ορισμένα θέματα τα οποία προκύπτουν από τη σημερινή συζήτηση, ειδικά, ειδικότερα την αντιμετώπιση των ασθενειών. Γι' αυτό η πρώτη μου ερώτηση αναφέρεται στις ασθένειες που αναφέρατε προηγουμένως, δηλαδή AIDS, ελονοσία και μια στιγμή ξεχνώ την τρίτη, εννοεί την φυματίωση, να δούμε εάν μπορούμε να πούμε ε, πόσοι απειλούνται από τις ασθένειες αυτές, διότι Γνωρίζουμε ότι η ελονοσία, για παράδειγμα, σε ορισμένες χώρες της Αφρικής ήδη έχει απαλληφθεί. Στο Σουδάν, ας πούμε, έχει, έχουν μειωθεί σημαντικά οι αριθμοί των κρουσμάτων. Αυτό είναι, αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Δεύτερο, μπορεί να πει κανείς κατά αναλογία πόσα χρηματοδοτικά κονδύλια δίνονται για την υποδομή, για τις ιατρικές εγκαταστάσεις, για την εξασφάλιση πόσιμου νερού, πόσα χρήματα δίνονται για κατάρτιση και για περαιτέρω κατάρτιση του ιατρικού προσωπικού, διότι οφείλει να γνωρίζει κανείς ότι σε πολλούς από τους τομείς αυτούς που αναφέρεται, οι γιατροί Μπορεί να έχουν κατάρτιση βέβαια, αλλά δεν έχουν επαρκή ιατρικό εξοπλισμό. Δηλαδή ε, προσπαθούν οι άνθρωποι αυτοί να ε, εξετάσουν τον κόσμο με ένα στιθοσκόπιο. Δεν έχουν ούτε καν ε, μηχανήματα ακτινογραφιών. Ε, τρίτη μου ερώτηση, η θεραπεία. Η θεραπεία με αντιβιωτικά. Γνωρίζουμε ότι πολλές από τις νόσους, όπως για παράδειγμα η φυματίωση, έχουν πλέον γίνει ανθεκτικές στα αντιβιωτικά. Και ε, Αυτό, αυτό σημαίνει ότι πρέπει οι φαρμακευτικές εταιρείε να εγκύψουν, να ψάξουν να βρουν νέα φάρμακα, διότι αυτό θα καθορίσει και το μέλλον. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ τους ηγητές μας για τις δύο εισηγήσεις που είναι σημαντικές και για μας για να αρχίσουμε να βλέπουμε πώς εφαρμόζονται οι στόχοι σε αυτή τη τριετία. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε το ρόλο που διαδραματίζουν όλα αυτά στο εσωτερικό του προπολογισμού και των κονδυλίων και με ποια είναι τα κατάλληλα στοιχεία για να ενισχύσουμε ακριβώς τις χρηματοδοτήσεις και να ελέγξουμε ακριβώς και τις χρηματοδοτήσεις για αυτές τις τρεις παθήσεις. Πρώτη ερώτηση αφορά τα συστήματα υγείας. Ξέρουμε καταρχάς ότι θα πρέπει να ενισχυθούν και λαμβάνουν υπόψη τους τα συστήματα υγείας και άλλα στοιχεία όμως με, στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν τις παθήσεις αυτές. Δηλαδή υπάρχει σύγχρονη ιατρική και υπάρχει παραδοσιακή ιατρική. Πολλές φορές δύσκολα τα άτομα πάνε στα νοσοκομεία ή στα κέντρα υγείας επειδή αγνοούν ή δεν εμπιστεύονται αυτά τα συστήματα αλλά ξέρετε πόσο σημαντικό είναι ακριβώς να ενισχύσουμε αυτά τα δύο συστήματα ώστε να δώσουμε μια ισχυρή απάντηση και στους ασθενείς οι οποίοι δυστυχώς είναι μακριά α, λόγω νοοτροπίας από αυτά τα συστήματα υγείας. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Ένα δεύτερο ερώτημα είναι αυτό που υπογράμμισε η Φανή είπε ότι υπάρχουν όλο και λιγότερα κονδύλια όσον αφορά την ενίσχυση δηλαδή της κοινωνίας των πολιτών. Ρωτά την Κομισιόν αλλά και εσάς. Είδατε να υπάρχει διαφορά στην εργασία των ΜΚΟ και των άλλων οργανώσεων γιατί πολλές από αυτές τις οργανώσεις δέχτηκαν κατηγορίες. Αντί λοιπόν να έχουμε δημόσια κονδύλια οι προσφορές και τα άλλα κονδύλια φαίνεται να μην πηγαίνουν εκεί που πρέπει. Δεν θα πρέπει λοιπόν να θεωρώσουμε λιγάκι για την χρηματοδότηση ώστε να ενισχύσουμε περαιτέρω τα δημόσια ταμεία. Να μου πείτε αν υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά και εδώ όσον αφορά αυτά που διαδραματίζονται επί τόπου. Και κλείνω λέγοντα το εξή. Στη διαδικασία αυτή, πέραν της ενίσχυσης των δομών στι χώρε προέλευση, μήπω θα πρέπει να ισχύσουμε και τι δομέ στι χώρε διέλευση. Γιατί εντωμεταξύ οι μετανάστε είναι άτομα αδύναμα, ασθενή. Οπότε πολύ συχνά είναι θύματα μετάδοσης αυτών των ασθενειών. Οπότε θα πρέπει να ενισχύσουμε ακριβώς και τις δομές με πόρους και στις χώρες διέλευση. Ευχαριστώ. Then we give the floor to a commission. Ναι, Επιτροπή. Ο Γιάν Πάλερ. Γρήγορα μα. ε. Ναι, ευχαριστώ. Μακροχρόνιος υποστηρικτή τη Ένωσης από την απαρχή του, του Ταμείου του 2002 και η συμβολή μας στο Ταμείο είναι 1,9 δις από το 2002 και 475 εκατομμύρια την περίοδο 17-19. Συγχαίρουμε το Ταμείο για τα αποτελέσματά του και τον εκκληστικό διευθυντή Πίτερ Σάντς για αυτές τις τρεις παθήσεις που συνέβαλαν η δράση του τομείου στο να σωθούν εκατομμύρια ζωές. Και αυτό δεν αφορά μόνο το AIDS, αυτό που απασχολεί τους περισσότερους, αλλά και ελονοσία, και η φυματίωση, η πρόληψη και η θεραπεία τους. Και μάλιστα στην διάσκεψη της ΦΟΥΓΚΑ είχαμε μια υψηλό επίπεδο συνάντηση για την φυματίωση συγκεκριμένα. Παρά λοιπόν την ορατή πρόοδο σε πολλές χώρες εταίρους μας, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε και τις σημαντικές προκλήσεις και στις τρεις παθήσεις που παραμένουν. Δηλαδή για το AIDS, σε κύρια κομμάτια του πληθυσμού πρέπει να δοθεί προτεραιότητα γυναίκες και νέα κορίτσια, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε πολλές χώρες, αντίσταση στα φάρμακα στην θυματίωση και η εμφάνιση κουνουπιών τα οποία αντιστέκονται σε διάφορους τρόπους πρόληψης κάτι το οποίο μας ανησυχεί ιδιαίτερα και θα πρέπει η Ένωση να δώσει επίσης και ιδιαίτερη σημασία στο να φτάσει αυτή η βοήθεια σε αυτούς που χρειάζονται περισσότερο στις πιο μακρισμένε περιοχέ και στι ε, περιοχέ που βρίσκονται σε κατάσταση πολέμου. Στην περιοχή, α πούμε, του Σαχέλ. Εκεί θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά τα διαθέσιμα κονδύλια από το Παγκοσμίο Ταμείο. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι δράσει του Παγκοσμίου Ταμείου θα πρέπει να συντονιστούν με την ταυτόχρονη βοήθεια που δίδεται στον τομέα σε αυτό το χρόνο, ώστε να ενισχύσουμε τα εθνικά συστήματα υγεία Σε αυτό το πλαίσιο η Κομισιόν συνεργάζεται με το Παγκόσμιο Ταμείο για να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των δράσεών μα και των συνεργασιών μα. Νομίζω ότι η Ένωση του δίνει ιδιαίτερη σημασία στι προσπαθήσει και στι δραστηριότητε και των άλλων πρωτοβουλειών του Παγκοσμίου Ταμείου ε, για την παγκόσμια χρηματοδότηση κλπ. Και όπως αναφέρθηκε προηγουμένως από τον Επιτρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δεσμευμένη στο να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο με μια διάσκεψη στη Γαλλία το 19 ώστε να διασφαλίσουμε την ύπαρξη επαρκών πόρων για τις μονοδικές μας παρεμβάσεις. Και συγκεκριμένα για τη χρηματοδότηση είναι αλήθεια ότι τα στοιχεία που αναφέρθηκαν στο NDICI που πρότεινε η Κομισιόν στο Μηχανισμό δηλαδή Γειτονία Ανάπτυξη και Εθνού Εργασία, είναι αλήθεια ότι εδώ αυτό το όργανο συγκεντρώνει αυτό που χρηματοδοτούταν από το εργαλείο γειτονίας χωριστά. Έχουμε λοιπόν ένα νέο τρόπο προγραμματισμού, πιο εύκολο και πιο εύκολο να εποπτευθεί όσον αφορά τις πληρωμές. Και πράγματι μπορούμε να προτείνουμε να αυξηθούν τα κονδύλια για συγκεκριμένε βιογραφικές περιοχές, ώστε να έχουμε μια πιο συγκεκριμένη προσέγγιση αναχώρα και να ενισχύσουμε την, ε, το τομέα υγείας τους θα έπρεπε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε παγκόσμιες πρωτοβουλίε μέσω του Παγκόσμιου Ταμείου ανάλογα με τις διεθνείς προκλήσεις και τα γεωγραφικά προγράμματα που είναι παρόν το Παγκόσμιο Ταμείο, δηλαδή όλες αυτές τις χώρες οποίες ε, βοηθάμε στα πλαίσια διεθνούς μας συνεργασία. Επίσης υπάρχει μια πρόταση για ένα 20% των πόρων να αφορούν την ανθρώπινη ανάπτυξη, ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων ώστε να διασφαλίσουμε την συνέχιση στήριξης του ανθρωπίνου δυναμικού. Τώρα για συγκεκριμένα ερωτήματα, το πώς θα στηρίξουμε την εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού. Δεν μπορώ να σας δώσω κάποια γενικά στοιχεία, αλλά σε γενικές γραμμές η συμβολή της Ένωσης στα προγράμματα υγείας είναι 1,3 δις ευρώ για το τωρινό ΠΔΠ και τις πρωτοβουλίες ε, Γκάβη, ας πούμε, για τα εμβόλια, μετά οικογενικός προγραμματισμός, σε με το ΟΗΕ και ε, κύρια παρέμβαση σε χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Και τρία δις επίσης, σήμερα 1,3 δις επίσης, ε, προβλέπονται σε γεωγραφικές παρεμβάσεις σε 17 συγκεκριμένε χώρες που αφορούν ευρεία προγράμματα και τα συστήματα υγείας τους περιλαμβανομένης και της κατάρτισης του ιατρικού προσωπικού. Αυτά δεν αποκλίνει το ένα το άλλο, τα χρειαζόμαστε ταυτόχρονα. Δηλαδή τοπικέ παρεμβάσεις και παγκόσμιες παρεμβάσεις σε συνεργασία με τα θεσμικά όργανα και τους στόχους που έχουμε χαράξει. Τώρα, για τη χρηματοδότηση στο ΜΚΟ. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε παρεμβάσει στον τομέα της υγείας με τη συμμετοχή των αντιπροσωπείων της Ένωσης και έχουμε τις πρωτοβουλίες του Παγκοσμίου Ταμείου που περιλαμβάνουν μεγάλα ποσά που μεταφέρονται στην ε, κοινωνία των πολιτών και αποφέρουν συγκεκριμένα τα δικαιώματα, την υγεία, και τις, οι διάφορες άλλες ε, υπηρεσίες οι οποίες αφορούν με μειονεκτών της πληθυσμούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Σάντς για δύο λεπτά παρακαλώ. Θα είμαι πολύ σύντομος. Η κυρία Σαβόσκα ρώτησε για ποιο μιλάμε εδώ, ποιους αφορά οι τρει αυτέ ε, ασθένειες ε, δεν αφορούν τα ίδια κομμάτια πληθυσμού, αλλά το κοινό στοιχείο τους είναι ότι αυτοί που πλήττονται περισσότερο είναι πιο φτωχοί, πιο αδύναμοι και υπεριθωριοποιημένοι. Αυτοί είναι οι πληθυσμοί κλειδιά στις διάφορες κοινωνίες μας. Και αυτό τονίζει βέβαια τη σημασία αντιμετώπιση αυτών των ασθενειών. Όπως επίσης και τη σημασία της κοινωνίας των ε, πολιτών παγκοσμίω στα πλαίσια του Παγκοσμίου Ταμείου. Ρόλος που είναι τεράστιος ώστε να φτάσουμε και να εξυπηρετήσουμε αυτούς τους περιθωριοποιημένους πληθυσμούς. Το άλλο που θα ήθελα να σχολιάσω για τη φυματίωση και την αντίσταση στα φάρμακα. Αυτή η αντίσταση αποτελεί μια παγκόσμια απειλή και το 1 τρίτο των θανάτων αφορά αυτό ακριβώς την αντίσταση στα φάρμακα κατά της φυματίωσης. Το Ταμείο είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας κατά πολέμηση αυτού του φαινομένου και είμαστε πολύ ενεργοί σε συγκεκριμένες χώρες και στοχεύουμε τις παρεμβάσεις μας και τις επενδύσεις μας ακριβώς στην καταπολέμηση της ε, αντίστασης των φαρμάκων της φυματίωσης. Όμως να είμαστε ρεαλιστέ. Αν θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο, πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ίδια τη θυματίωση καταρχά. Γιατί εκεί βεβαίω που έχουμε φυματίωση έχουμε μεταλλάξει και τι παραλλαγέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Βίλαρ. Ευχαριστώ. Για να απαντήσω στην ερώτησή σας, δηλαδή διάκριση γεωγραφικών και θεματικών προγραμμάτων, διότι μας είπαν ότι μειώνονται τα θεματικά πρόγραμμα, προγράμματα και αυξάνονται τα γεωγραφικά. Και ότι θα χρηματοδοτηθούν οι παγκόσμιες πρωτοβουλίες μέσω των γεωγραφικών. Αυτά όμως είναι pool funding, δεν μπορούμε δηλαδή να διαθέσουμε ειδικά ταμεία σε, ειδικές, σε ε, ε, ορισμένα ταμεία σε ορισμένες χώρες. Η Κομισιόν ζητεί κονδύλια από τους φακέλους αυτούς, αλλά πώς μπορούμε να εγγυηθούμε ότι αυτά τα κονδύλια θα δαπανηθούν σε συγκεκριμένε χώρες. Είναι πολύ δύσκολο για λόγους προβλεψιμότητας, ε, λογιστική αποτίμηση, αλλά και αξιοπιστίας, όπως είπατε τώρα, για να συζητήσω τα δύο αυτά θέματα ταυτόχρονα, δηλαδή AIDS και ε, φυματίωση. Αυτά που γνωρίζω καλύτερα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, ε, αυτά κτυπούν, πλήττουν ευάλωτου πληθυσμού. Πρέπει λοιπόν να δει κανεί και το σύστημα υγείας αλλά και ένα ε, σύστημα οικονομικό το οποίο να αντιμετωπίζει την ανισότητα στην Ευρώπη. Είμαστε η μοναδική περιοχή του κόσμου όπου αυξάνονται οι αριθμοί των οροθετικών προσώπων. Αν εξετάσετε το πρόγραμμα NFF, για τον, ε, δηλαδή ΠΔΠ για τον τομέα της υγείας, εκεί προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μείωση και δεν ξέρουμε αν θα έχουμε καν χαρτοφυλάκιο επιτρόπου για θέματα υγείας μετά από τη Βρετανική έξοδο. Βλέπω ότι στο επόμενο θέμα σας θα συζητήσετε τον ορίζοντα Ευρώπη. Εκεί ε, προβλέπεται μεγάλη χρηματοδότηση για τους στόχους SDG3 και περισσότερη έρευνα για την υγεία, ειδικά για ε, AIDS και φυματίωση. Εκεί που θέλω να στοχεύσω τώρα είναι η ανάγκη της κοινωνιακής επέκτασης της έρευνας, θέλουμε επίδραση μάλλον της έρευνας, διότι για την ώρα βασίζουμε την έρευνα μόνο σε μια προσπάθεια αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Πρέπει η έρευνα να αποδείξουμε ότι έχει επίδραση και στην κοινωνία. Ευχαριστώ πολύ. Ένα σύντομο ερώτημα, κύριε Γκέρενς, έχετε ένα λεπτό. Πρόκειται για μια πρόταση, διότι εφόσον πρόκειται να συναντηθούμε με τους υπευθύνους του τομέα υγείας, αυτό θα γίνει για να δούμε τι μπορούμε να διαθέσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερο, να δούμε και ποια είναι η επίπτωση της χρηματοδότησης αυτής. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την ε, προσεχή περίοδο χρηματοδοτήσεως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον ενιαίο μηχανισμό χρηματοδότησης, θέλω να μάθω αν τα πράγματα θα είναι πιο απλά ή πιο περίπλοκα. Και για να είναι ξεκάθαρα, πριν από την έγκριση της εκθέσεως που θα γίνει τέλη του μηνό, θέλω να μάθω σε ποιο μέτρο οι νέες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν θετική ή αρνητική επίπτωση στον τρόπο που εργάζεται το Παγκόσμιο Ταμείο. Σημαίνει αυτό ότι θα αναγκαστεί το Παγκόσμιο Ταμείο να αλλάξει τρόπο διαχείρισης στην οποία περίπτωση θα πρέπει να διερωτηθούμε εάν οι τροποποιήσεις που κάνουμε είναι πραγματικά προς το συμφέρον μιας λύσης. Εγώ θέλω κάποια διαφώτιση. Δεν αφιβάλλω καθόλου για την καλή θέληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέναντι στο Παγκόσμιο Ταμείο. Θέλω όμως να με βοηθήσει να αντιληφθώ ω εισηγητής την προβλεψιμότητα των δαπανών για τον τομέα υγεία ό,τι αφορά τη χρηματοδότησή τους. Και αυτά, ε, ορίστε. Εάν μπορούν ε, να μου δώσουν κάποια διαφώτιση και μιλώ στο όνομα και των άλλων τριών συνεισηγητών για την πτυχή αυτή θα μου διευκολύνει το έργο. Δεχόμαστε πολλές ερωτήσεις. Και για να αποφευθούν οι παρανοήσεις πρέπει να υπάρξουν πλήρες διευκρινήσεις για να μην γίνονται τα πράγματα πιο δύσκολα και μέσα στην Επιτροπή μας και στο Κοινοβούλιο συνολικότερα. Πρόεδρος, ίσως μπορούμε να ακούσουμε την απάντηση αργότερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή θέλετε εσείς να πείτε κάτι κύριε Σάντς. Ναι, θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ για την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το ίδιο ευγνώμων είμαι και για την ερώτηση του κ. Γκέρενς, διότι νομίζω ότι η σαφήνεια εν προκειμένου είναι ουσιώδης για μας, για να έχουμε καθαρή εικόνα πώς μπορούμε να προγραμματίσουμε τις χρηματοδοτήσεις μας για την επίτευξη των στόχων SDG 3. Ευχαριστώ για την ε, παρουσία σας εδώ και για τη συμμετοχή σας στην συζήτηση. <clears throat> Ευχαριστώ, ε, ευχαριστούν οι δύο προσκεκλημένοι και από ε, Θα συνεχίσουμε, λέει η Πρόεδρος, με τις δύο προτάσεις, 5 και 6. Το νέο πλαίσιο για έρευνα και καινοτομία για την περίοδο 2021-2027 αποτελούνται από δύο ντοσιέ νομοθεσία που θα θεσπίσει κανόνες συμμετοχής και διάδοσης και αποφάσεις για συγκεκριμένα προγράμματα θα συζητήσουμε μαζί, από κοινού δηλαδή, τον προτινόμενο κανονισμό και την προτινόμενη πρόταση, το σχέδιο προτάσεω δηλαδή. Επαναλαμβάνω, πρόκειται για τα θέματα 5 και 6 της ημερήσια διάταξης. Με προτινόμενου προπολογισμού πάνω από 94 δισεκατομμύρια ευρώ για την ε, προγραμματική περίοδο το Horizon Ευρώπη προτείνει το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα έως τώρα για χρηματοδότηση έρευνας και καινοτομίας. Και ναι μεν πρόκειται για πρόγραμμα το οποίο ωφελεί καταρχήν την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, το πρόγραμμα ωστόσο προσφέρει και κάποιες ευκαιρίες για αναπτυσσόμενες χώρες και για περαιτέρω πρόθεση του θεματολογίου SDG, δηλαδή των ε, στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Η αρμόδια επιτουσίας επιτροπή που είναι η ΙΤΡΕ, παροιμήν, προωθεί μια πολύ φιλόδοξη ατζέντα και η ψηφοφορία προβλέπεται στην επιτροπή τους στις 21 ενδεκάτου. Η δε ψήφος ε, στην ε, Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προβλέπεται στην μήνυ περίοδο συνόδου του τέλου του Νοεμβρίου. Άρα το χρονοδιάγραμμα είναι πολύ σφιχτό και οδηγεί στην ανάγκη οργάνωσης έκτακτης συνάντησης της Επιτροπής μας στο Στρασβούργο στις 12 Νοεμβρίου, ώστε να μπορέσουμε να ψηφίσουμε τα δύο σχέδια γνωμοδοτήσεων. Ωραία λοιπόν, τώρα έχουμε την εισηγήτριά μας, κυρία Σάντσες Καλντεντέι, Ορίστε παρακαλώ, έχετε το λόγο κυρία Σάντσες Γκάλτεντέι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Προσπαθήσαμε το σχέδιο να απηχεί καινοτόμες ιδέες και ρεαλιστικές. Και προσπαθούμε να υπερβούμε τις ελλείψεις του ορίζοντα 2020. Εδώ πήραμε ως βάση τους SDG κάνουμε μια προσπάθεια να στοχεύσουμε σε ειδικού τομεί, έρευνα για την υγεία, πρόσβαση στα φάρμακα. Θέλουμε να έχουμε μια στέρεα οικονομική συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες, να αντιμετωπιστούν οι σημαντικότερες κοινωνικές προκλήσεις, η ανάπτυξη η ισότητα των φύλων, θέλουμε περισσότερη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην ε, λήψη αποφάσεων, θέλουμε να ιδρύσουμε μηχανισμούς που θα επιτρέψουν οι επενδύσεις να αποδίδουν υπέρ της κοινωνίας και θέλουμε να μπορούμε να συγκεντρώνουμε τα δεδομένα των ερευνών. Σε ό,τι αφορά την παγκόσμια υγεία και την πρόσβαση στα φάρμακα, εξετάζουμε με ανησυχία τις προτάσεις της Επιτροπής, διότι δεν επιτρέπουν επαρκή έρευνα προς το δημόσιο συμφέρον. Εξετάζουμε επίσης τους στόχους SDG3. Η πρόσβαση στο φάρμακο είναι μεγάλη πρόκληση για πολλές χώρες. Γι' αυτό χρειαζόμαστε το νέο πρόγραμμα πλαίσιο, όχι μόνο να αυξήσει τον προϋπολογισμό για θέματα υγείας, θέλουμε επίσης να μπορεί να γίνει και μεταφορά βιομετρικής, βιο, συγγνώμη, βιοιατρικής τεχνολογίας και να προσφέρει την ευκαιρία να υλοποιηθούν οι συστάσεις του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στον ε, τομέα αυτό, ιδίως όσον αφορά την θετική επίπτωση στην κοινωνία της βιοϊατρικής έρευνας. Θέλουμε επίσης να υπάρχουν στέρεα συστήματα υγείας, κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Και σε ό,τι αφορά τη διεθνή συνεργασία, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπέρ της διαμεθοριακής έρευνας. Είδαμε όμως τις τελευταίες δεκαετίες μια διαρκή, μια σταθερά μείωση των διαμεθοριακών ε, κονδυλίων. Μόνο 3% του επόμενου πιδελταπή είναι για διαμεθοριακά προγράμματα. Δεν έχουν δημιουργηθεί μηχανισμοί για την λεγόμενη επιστημονική διπλωματία ούτε επιτρέπουν επιστημονική ανάπτυξη σε χώρες μεσαίου ή χαμηλού εισοδήματος. Για να υλοποιηθούν όμως οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης, πρέπει να γίνει προσπάθεια σε στρατηγικούς τομείς για, τις, ε, για την ανάπτυξη οικονομίας των χώρων αυτών. Θέλουμε οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης να αποτελέσουν το θεμέλιο για την ανάπτυξη αυτή για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε και τι είδους πρόοδος γίνεται. Μας ανησυχεί πολύ η στόχευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην βιομηχανική ανταγωνιστικότητα. Θεωρούμε ότι μια ορθή δημόσια πολιτική θα πρέπει να αποδίδει κοινωνικά ωφέλη και απτή ωφέλεια για τις κοινωνίες. Πρέπει να διακρίνουμε ανάμεσα σε θέματα επιδίωξης κέρδους και κοινωνικά. Θέλουμε να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο. Να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στις κοινωνικές επιπτώσεις της υλοποίησης των προγραμμάτων, ιδίως των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και της Συμφωνίας του Παρισιού. Να πάψουμε να χρηματοδοτούμε έρευνα σε, μεγάλους, σε μεγάλες βιομηχανίες που ρηπαίνουν ή σε μεγάλες ε, πηγές ενέργειας που ρηπαίνουν. Να στοχεύσουμε περισσότερο στις ε, ανανεώσιμες ενέργειες και στην αποδοτική χρήση των ενεργειών. για να περάσουμε έτσι την οικολογική μετάβαση των κοινωνιών μας που με τη σειρά της θα οδηγήσει σε εκατομμύρια ε, βιώσιμων θέσεων απασχόλησης σε μια οικολογική οργάνωση της οικονομίας. Επίσης, είναι πολύ σημαντική η συμβολή της κοινωνίας των πολιτών στην ε, θέσπιση των προτεραιοτήτων. Θέλουμε το νέο πρόγραμμα να μην χρησιμοποιεί μονάχα διαβουλεύσεις επιγραμμικά για να έλθει σε επαφή με την κοινωνία των πολιτών. Τέλος, ο νέος ορίζον δεν περιλαμβάνει ρήτρες που να επιβάλλουν κοινωνική απόδοση, απόδοση πέρα κοινωνίας των επενδύσεων. Θέλουμε οι νέες τεχνολογίες να γίνουν βιώσιμες και προσβάσιμες από την κοινωνία. Για αυτές τις ιδέες αγωνιζόμαστε στη γνωμοδότησή μας. Ελπίζομαι μέχρι τις 24 να μπορέσουμε να περιλάβουμε και άλλες ιδέες ώστε η Επιτροπή μας να δώσει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στη Συναρμόδια Επιτροπή Ήτρε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει και η Πρόεδρος. Δεν έχουμε σκιώδεις συζητητές εδώ. Έχουμε όμως την κυρία Κένγκε. Έχετε το λόγο, κυρία μου. Λίγα λόγια για το σχέδιο γνωμοδότησης, ιδίως για το ορίζον Ευρώπη εξ ονόματος του κυρίου Φρουντζούριτσα, που είναι συνεισηγητής των Σοσιαλδημοκρατών και σήμερα κολλείεται να προσέλθει. Υποστηρίζουμε το πρόγραμμα Ορίζον Ευρώπη για να ενισχύσει τις επιστημονικές βάσεις της Ένωσης, για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις των καιρών μας και να υλοποιηθούν οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης. Δεχόμεθα ότι τα έργα που θα γίνουν στο, πρόγραμμα του, πλαίσιο του προγράμματος θα πρέπει να προωθούν την ισότητα μεταξύ των φύλων στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Χαιρόμαστε για το γεγονός ότι το προτινόμενο πλαίσιο ορίζων Ευρώπη προβλέπει διεθνείς συνεργασίες. Ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών που να είναι προς αμοιβέων Να μην λησμονούμε ότι ειδικώ για τι αναπτυσσόμενες χώρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αποτελεί ισχυρό παγκόσμιο εταίρο για την ενίσχυση τη έρευνα και τη καινοτομία και οι ομάδε τη διασποράς στην Ευρώπη αποτελούν σημαντικό συνδετικό κρίκο. Ιδίω για τι χώρε ΑΚΕ, Αφρική Καραϊβική Ειρηνικού, να ενισχυθούν οι πρωτοβουλίε αυτέ μέσω πρωτοβουλειών όπω Alliance Afrique, Europe, δηλαδή Συμμαχία Αφρική Ευρώπη και άλλα ε, βιώσιμα προγράμματα. Επίσης, να διατηρηθεί συνοχή με άλλους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς που υπάρχουν ήδη, όπως τα καταπισματικά ταμεία για την απόκτηση προσόντων και εκπαίδευση. Και ορίζον Ευρώπη να διευκολύνει τη χρηματοδότηση και υποστήριξη σχεδίων, προγραμμάτων, έργων. Αυτό είναι και μια κριτική των αναπτυσσόμενων χωρών, διότι η πρόσβαση στα, στις χρηματοδοτήσεις είναι πολύ δυσχερής και δαπανηρή. Πρέπει η Ευρώπη να ενισχύσει την καινοτομία και την έρευνα σε τομείς που είναι σημαντικοί για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτό έχει κρίσιμη σημασία αν θέλουμε να επιτύχουμε τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Για παράδειγμα, πιο σημαντική ενίσχυση στην έρευνα και καινοτομία για τις παραμελημένες νόσους, όπως έχουμε δει με την ανάπτυξη εμβολίου κατά του έμπολα. Δεύτερο, απαιτήσει για θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας δεν θα πρέπει να αποτελούν εμπόδιο για την πρόσβαση στα φάρμακα. Διότι τα φάρμακα πρέπει να προκύψουν και από νέες έρευνες και με θέσπιση νέων μηχανισμών για την ενθάρρυνση των ερευνών αυτών. Οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για μια ενδεχόμενη χρήση τους ιδίω στι αναπτυσσόμενε χώρε. Για παράδειγμα, αποτελεσματική γεωργία, ευφυή γεωργία, ενίσχυση σε περίπτωση θεομηνιών, ανθρωπιστική βοήθεια. Να, να ε, υπογραμμίσουμε επίσης ότι το νέο πρόγραμμα στοχεύει σε παράγοντε συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες και σε πιο δύσκολα θέματα, όπως η χαμηλή ευαισθησία του ορίζοντα 2020, ανισότητα στην πρόσβαση σε πληροφορίες, θέματα συνεργασίας, καθώς και δυσκολία εξέβρεσης Ευρωπαίων εταίρων από την πλευρά δηλαδή των αναπτυσσόμενων χωρών. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ και εγώ λέει η Πρόεδρος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχει κανείς που επιθυμεί να λάβει το λόγο. Η κυρία Νόρστετ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια, Λόλα Σάντσες, και τους ε, υπόλοιπους ευρωβουλευτές που σχολίασαν. Η συνεισφορά σας είναι πολύ σημαντική. Όπως ανέφερα, ο Horizon Ευρώπη είναι ένα αρκετά φιλόδοξο πρόγραμμα για την έρευνα και την καινοτομία και είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε επίσης, όπως άλλωστε τονίστηκε και πριν, ότι είναι μέρος άλλων ε, αντίστοιχων προγραμμάτων στον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό του πολιτισμού οικονομικού πλαισίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να τονίσω ότι ο Horizon Ευρώπη είναι ένα πρόγραμμα ανοιχτό στη συνεργασία για εταίρους από όλο τον κόσμο και αποτελεί μια νέα προσέγγιση στην πρόσβαση στα προγράμματα για όλες τις χώρες που έχουν ικανότητες έρευνας, επιστήμης και καινοτομία. Και η προσχώρηση των τρίτων χωρών θα είναι και απόδειξη τη ε, βούλησή του να κάνουν πολλά περισσότερα, ε, βασισμένη στην αρχή τη αμοιβαιότητα. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι τα περισσότερα προγράμματα του Horizon Ευρώπη και Horizon 2020 που τρέχουν αυτή τη στιγμή είναι προγράμματα συνεργατικά όπου καταργούνται τα γεωγραφικά σύνορα στην επιστημονική συνεργασία. Αυτό είναι έτσι προς προβληματισμό. Επίσης, σε ό,τι αφορά τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, βλέπετε και από τα προγράμματά μας ότι έχουμε δεσμευτεί να συνεισφέρουμε στην υλοποίησή του. Και η παρακολούθηση του προγράμματος είναι εξίσου σημαντική. Ακούσαμε μάλιστα πως ε, υπάρχει επιθυμία να εξετάσουμε τη συνεισφορά μας ε, στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που αφορούν την υγεία και τον ε, κύκλο καινοτομία στην ιατρική έρευνα. Αυτός ο κύκλος είναι αρκετά μεγάλος σε σύγκριση με άλλους τομείς, γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται περισσότερος χρόνος από ό,τι συνήθως, έτσι ώστε να μετρήσουμε τον αντίκτυπο κάποιου προγράμματος σε αντίθεση με την, ε, τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας, όπου τα πράγματα τρέχουν πολύ πιο γρήγορα και ο κύκλος της καινοτομίας είναι πολύ μικρότερο. Στην ιατρική μιλάμε για κύκλους 10-15 ετών. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε τρόπους μέτρησης. Επίσης υπάρχουν κάποια μοντέλα που είναι πολύ αποτελεσματικά σε ό,τι αφορά την ε, υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Για παράδειγμα ένα μέσο που εξετάζει τον αντίκτυπο και χρησιμοποιείται πιλωτικά σε προγράμματα επισητιστικής ασφάλειας, βιώσιμης γεωργίας, έρευνας και κοινοτομίας στο πλαίσιο του διαλόγου με την Αφρικανική Ένωση για τα θέματα αυτά. Θα μπορούσαμε λοιπόν να κοιτάξουμε και αυτά τα μέσα, να δούμε πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε κατάλληλα. Επίσης, ε, με χαρά μας ακούμε τα σχόλιά σας για την ισότητα των φύλων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλες τις κυβερνήσεις, αλλά και στο ερευνητικό πεδίο. Θεωρούμε λοιπόν πως είναι πολύ σημαντικό μέρος του προγράμματος. Επίσης, η πρόταση αυτή προβλέπει την ε, συμπερίληψη των διάφορων ε, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, της κοινωνίας των πολιτών, τη συμμετοχή όλων αυτών λοιπόν στην διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού και να αναφέρω επίσης ότι οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών είναι πάντα ευπρόσδεκτοι σε όλες τις δράσεις και τα έργα που χρηματοδοτούμε, στον τομέα της υγείας ιδιαίτερα η συνεργασία μας με την κοινωνία των πολιτών, με εκπροσώπους που μας στενών, πάντα άριστη. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση πρέπει να διευκρινιστεί πως ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέχουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να ερευνούμε ε, και να εξετάζουμε το πώς ε, χρησιμοποιείται η χρηματοδότηση από τους ερευνητές. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια ανοιχτή πρόσβαση για επιστήμονες σε διάφορα στατιστικά στοιχεία. Νομίζω πως ε, αυτά ήταν συνοπτικά ε, τα όσα ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Η συγγήτρια έχει κάποιο σχόλιο. Όχι, σας άρεσαν όλα. Πολύ ωραία. Προθεσμία υποβολής τροπολογιών 24 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ. Προχωράμε τώρα στο σημείο 7 για την προσχώρηση της ΣΑΜΟΑ στην ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών του Ειρηνικού. Η Σαμόα αποχώρησε από την κατηγορία των ελάχιστα αναπτυγμένων χωρών το 2014. Και ως αποτέλεσμα προάχθηκε λοιπόν και θα χάσει ε, τις, διάφορε, τις διάφορες, ε, διάφορα προνόμια που προκύπτουν από την θέση αυτή. Μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2018 θα ισχύει η συνηθισμένη μορφή του ε, γενικευμένου συστήματος προτιμήσεων το οποίο φυσικά είναι πολύ λιγότερο γενναιόδωρο από ότι το EBA, το Everything But Arms. Η Σαμόα θα πρέπει να προσχωρήσει στην ε, παρούσα συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Φίτζι και την ομάδα PNG μέχρι τον, την 1η Ιανουαρίου του 2019. Περισσότερα λοιπόν από τον εισηγητή Φλωρά Μαρσεγεζή και θα του δώσω αμέσω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Σήμερα είναι σημαντική μέρα γιατί είδαμε την έκθεση των εμπειρογνωμόνων των διεθνών για την κλιματική αλλαγή που μας θυμίζει ότι θα πρέπει να δράσουμε πιο φιλόδοξα και πιο γρήγορα αν θέλουμε να τηρήσουμε τους στόχους της φωνίας των, του Παρισιού για αύξηση της θερμοκρασίας κάτω από 1,5 βαθμό μέχρι το τελευταίο του αιώνα. Έχουμε λοιπόν εδώ το διεθνές εμπόριο σε αυτή την ε, διαρθρωμένη μορφή του που είναι υπεύθυνο για τον πέμπτο εκπομπές, υπεύθυνο, το, υπεύθυνο για τον πέμπτο εκπομπών. Πρέπει λοιπόν να τηρήσουμε την, στα πλαίσια της φωνίας του Παρισιού αυτά προβλέπονται και κατά συνέπεια ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται το εμπόριο δεν είναι πια βιώσιμο. Είχαμε λοιπόν και μια προφανή κριτική ότι δεν περιμέναμε, δεν ήταν στο ύψος των προσδοκιών η συμφωνία αυτή ενώπιον των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Και σε αυτή την περίπτωση, μάλιστα, ε, η Σαμόα δεν είναι και ο πιο καθαρός εταίρος που έχουμε. Για την κλιματική αλλαγή είχαμε πάντοτε δύο στοιχεία. Αφενός είχαμε τις χώρες που είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για την κλιματική αλλαγή όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, αφενός και αφετέρου, είχαμε κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις, νήσους νησίδες όπως η Σαμόα που ήταν από τους ε, κυρίους, από τα κυριότερα θύματα ε, της κλιματικής αλλαγής όπως τα νησιά Φίτσι, του Βαλού κτλ. Οπότε στα πλαίσια λοιπόν αυτού του διεθνούς εμπορίου πρέπει να προσέξουμε πολύ γιατί αυτό που κάνει είναι για άλλη μια φορά να μην θέσει στο επίκεντρο με τρόπο δεσμευτικό και υποχρεωτικό και νομικά εφαρμόσιμο το θέμα της βιώσιμη ανάπτυξη και τη συμφωνία του Παρισιού. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να αποτελεί ένα μπούσουλα για τις εμπορικές μα συμφωνίες. Νομίζω επίσης ότι εδώ το Κοινοβούλιο ήταν ξεκάθαρο στις στα πρόσφατα ψηφίσματά του για την ανάγκη σύνδεση, νομικής σύνδεση της βιώσιμης ανάπτυξης με τις ε, συμφωνίες τις εμπορικές. Και μάλιστα στο Κοινοβούλιο είχαμε μια πρόταση υπέρ της συμφωνίας για την δεσμευτικό χαρακτήρα της συμφωνίας του ΕΕ που αφορούν το, τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Είπαμε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με πολλές μορφές εμπορίου και επιθυμίζουμε ότι όλα τα κεφάλαια της βιώσιμης ανάπτυξης στις εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει τα κεφάλαια αυτά να είναι νομικά εφαρμόσιμα και υποχρεωτικά δεσμευτικά. και για άλλη μια φορά έχουμε μια συμφωνία, άλλη μια συμφωνία που δεν λαμβάνει υπόψη σε αυτό το στοιχείο αντίθετα λοιπόν από τις προσδοκίες μας. Ελπίζω λοιπόν να αλλάξει αυτό, ώστε πράγματι το κεφάλαιο της βιώσιμης ανάπτυξης να είναι και δεσμευτικό και νομικά εφαρμόσιμο. Δεύτερο ζήτημα, κέριο επίσης, είναι το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έβαλε στο μαύρο κατάλογο χωρών που δεν συνεργάζονται χώρες όπως τη Σαμόα Νομίζω ότι θα πρέπει για μια φορά η Ένωση να έχει μια πιο λογική πολιτική αυτές τις περιοχές που δεν συμμορφώνονται φορολογικά και θα πρέπει να επενθυμίσουμε ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αυτά τα θέματα όταν ας πούμε συζητάμε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και οικονομικές σχέσεις όπως εδώ. Και δεν φτάνει μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τα λύνει αυτά σε μια συνάντηση με τη ΣΑΜΟΑ αλλά να κάνει πράγματα αποτελεσματικά και απτά μέσω εμπορική συμφωνίας. Γιατί το Κοινοβούλιο σε δύο ψηφίσματα διαφορετικά υπενθύμησε ξεκάθαρα ότι και για πολύ σοβαρά ζητήματα όπως αυτά τα φορολογικά με μια χώρα, αυτό θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να ακυρώσουμε μια εμπορική συμφωνία. Οπότε εδώ έχουμε ένα μελανό σημείο το οποίο θα πρέπει να λύσουμε. Δεν θα επεκταθώ, γιατί νομίζω ότι αυτά τα ζητήματα είναι θέματα αρχής αυτή η συμφωνία δεν είναι τόσο σημαντική για τη ΣΑΜΟΑ για την Ένωση, αλλά είναι ε, εδώ ένα θέμα αρχή. Δηλαδή, οι εμπορικέ συμφωνίε θα πρέπει να είναι ένα εργαλείο, όχι ένα αυτό, σκοπό, ένα εργαλείο το οποίο θα πρέπει να μα επιτρέπει να κάνουμε δύο πράγματα. Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, δηλαδή, αφενός και αφετέρου, στόχοι τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αν δεν τηρούνται αυτοί οι δύο στόχοι θα πρέπει να αναθεωρούμε τι συμφωνίε αυτέ ώστε ακριβώ να περιληφθούν αυτά τα δύο στοιχεία. Συμφωνία Παρισιού και Κλιματική Αλλαγή. Και νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση η συμφωνία με τη ΣΑΜΟΑ δεν τηρεί αυτού του δύο στόχου, που είναι οι πιο σημαντικοί στόχοι και πολύ πιο σημαντικοί βέβαια από ένα απλό εργαλείο όπω η εμπορική συμφωνία που απλά και μόνο θα πρέπει να τηρεί κάποιου κανόνε και νόμους που έχουμε εδώ, ενώ εδώ στην ουσία πρόκειται για την διάσωση της ανθρωπότητας με σωστό τρόπο για αυτούς που υποφέρουν από την ε, κλιματική αλλαγή και στα πλαίσια των εμπορικών συμφωνιών, όπως και στη ΣΑΜΟ αλλά και στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. you. Thank you very much. And then... Ευχαριστώ πολύ, κυρία Σκέγγε. Ευχαριστώ πολύ. Όπως είπα πριν, ο κ. Φρουτζουλίκα είναι ο σκιώδης εισηγητής, ο οποίος δυστυχώς δεν μπορεί να έρθει σήμερα. Από ό,τι θα πω κάποια πράγματα εξ ονόματός του. Καταρχάς θα πρέπει να εξετάσουμε το συμφέρον της ΣΑΜΑ όσον αφορά την εταιρική σχέση, την οικονομική. Και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η ίδια η χώρα το ζήτησε αυτό ως χώρα που θα προσχωρήσει αυτήν τη συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν αποτελεί τον πέμπτο εμπορικό εταίρο της περιοχής του Ειρηνικού. Οποιαδήποτε διακοπή όσον αφορά την πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές θα έχει σημαντικό αντίκτυπο. Το δασμολογικό καθεστώς και οι αλλαγές του θα αφορούν θα πειράσουν το 67% των εξαγών της ΑΜΟΑ προς την Ευρωπαϊκή Ένωση με απώλεια η οποία θα είναι πολύ σημαντική. 79 μάλιστα. Τόσο πολύ. Και ιδιαίτερα πρέπει να πούμε ότι τα προϊόντα ελίας τα οποία προέρχονται από εκείνη την περιοχή είναι πολύ σημαντικά για αυτούς. Και μάλιστα λαμβάνοντας υπόψη το γεγονό ότι αυτός ο υποανάπτυξη Τομέα ε, προσφέρει ακόμα θέσει εργασία στις απασχόλησης στις γυναίκες. Γι' αυτό ακριβώς οποιαδήποτε απώλεια σε αυτήν την αγορά θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο μεγάλη μελέτης. Θα πρέπει λοιπόν να προβλέψουμε πιθανές εναλλακτικέ λύσεις αν θέλουμε πραγματικά να προσχωρήσει την ενδιάμεση συμφωνία η Σαμόα, χώρα η οποία θα ε, υποφέρει ε, τη στιγμή που Φίτζη, η Παπόα Γουινέα και άλλες χώρες θα συνεχίζουν να έχουν άλλο ρόλο στα πλαίσια αυτών των συμφωνιών και όλα αυτά εις βάρος της ΑΜΟΑ. Θα πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε ότι η ενδιάμεση συμφωνία δεν αποτελεί μια μακρόπνοη λύση. Θα πρέπει να προβλέψουμε και άλλες χώρες ως υποψήφιες προς προσχώρηση στη συμφωνία, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για να αναθεωρήσουμε τους φραγμούς, που ε, εμποδίζουν την ολοκλήρωση αυτής της συμφωνίας. Επίσης, η νέα συμφωνία δεν καλύπτει το σύνολο των διατάξεων που αφορούν τα εργασιακά δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, του περιβαλλοντικού κανονισμούς, τον κοινοβουλευτικό, έλεγχο, την κοινωνία των πολιτών, όλε τέλο πάντων τι ε, διατάξεις οι οποίε αφορούν τι πλήρε συμφωνίε. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Τέλος, η σύναψη μιας ε, συμφωνίας σχέσης ενδιάμεσης θα πρέπει να αποτελέσει ένα βήμα προς μια ολοκληρωμένη σχέση μεταξύ Ένωσης περιοχής χωρών, χωρών περιοχής ειρηνικού μέσω επικοδομητικού διαλόγου και πριν από το συνεργασία, λαμβάνοντα υπόψη ότι ο στόχο είναι η σύναψη μια συμφωνία που θα επιτρέψει τη βιώσιμη ανάπτυξη και θα προωθήσει την ολοκλήρωση, την οικονομική και την περιφερειακή. Πράγματι, αν οι χώρες που θα προσχωρήσουν στην διάμεση λύση, αν οι χώρες αυτές προσχωρήσουν στην διάμεση λύση, αυτό θα πρέπει να αποτελέσει μια όθηση εν ώψη μιας πλήρους συμφωνίας και όπου θέματα βιωσιμότητας όπως η αλία θα πρέπει να αναθεωρηθούν. Λαμβάνοντα υπόψη το τι ισχύει εκεί στον Ειρηνικό για την αλία, ώστε οι κανόνες τους να είναι συμβατοί με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον πρεσβευτή Λούτερη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, και επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω και τους δύο ομιλητές που συνέβαλαν στη συζήτηση αυτή για την ε, προσχώρηση της χώρας μου στην διάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης. Εμείς καλωσορίζουμε αυτή την συζήτηση Η συμφωνία αυτή βέβαια είναι σημαντική για τη χώρα μου για διάφορους λόγους που αναφέρθηκαν. Πιστεύουμε και είπαν και άλλοι ότι το εμπόριο είναι ένα από τα εργαλεία για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης και των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Όπως και των στόχων της Συμφωνίας των Παρισιών. Και θεωρούμε ότι πράγματι υπάρχουν ευκαιρίες για μας για να εμπορευτούμε με την Ευρώπη και η χώρα μου είναι μία από τις 37 χώρες που θεωρούνται ως μικρές νησιώτικες αναπτυσσόμενες χώρες στην αντίστοιχη ομάδα. Εσείς, λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν συγκυρίες και συνθήκες που μας θέτουν δυσκολίες αν δεν έχουμε εμπορικούς εταίρους. Όχι μόνο για να εμπορευτούμε, αλλά να εμπορευτούμε και ανταγωνιστικά, Πρόεδρε, μιας και είμαστε μικροί. Θα πρέπει λοιπόν να στοχεύσουμε σε συγκεκριμένες αγορές για τις εξαγωγές μας. Επειδή βεβαίως δεν έχουμε όσον αφορά την πλευρά της τροφοδοσία τα απαραίτητα για να ανταγωνιστούμε σε διεθνές επίπεδο. Οπότε, Πρόεδρε, κυρία μου, πρέπει να δουλέψουμε και να ανταγωνιστούμε σκληρά στις εξαγωγές μας. Αναφέρει και το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Να καταστήσω σαφές ότι η χώρα μου, μαζί με άλλε χώρες του ειρηνικού και αλλού βέβαια, και αλλού, ε, είναι στην πρωτοπορία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Εμείς δεν θέλουμε δραστηριότητες ή συναλλαγές με χώρα ή ομάδες χωρών που προσεγγίζουν την κλιματική αλλαγή ως κάτι το οποίο δεν τις αφορά, ενώ αφορά εμάς και την επιβίωσή μας. Μας επηρεάζει λοιπόν η κλιματική αλλαγή και βεβαίως εμείς δεν θέλουμε να συμμετάσχουμε σε οποιαδήποτε συμφωνία η οποία θα επιταχύνει τα πράγματα και θα χειροτρέψει την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε εμείς. Επίσης είμαστε μια κοινωνία που αναγνωρίζει τη συμβολή των διαφόρων φορέων και να υπογραμμίσω και μια ομάδα που είναι κέρια σημασία για την κοινωνία μας όσον αφορά την προώθηση και εφαρμογή δραστηριοτήτων. Εμείς ε, στα χωριά μας έχουμε τις Επιτροπές των Γυναικών. Οι Επιτροπές δηλαδή που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή δραστηριοτήτων και προγραμμάτων. Και είναι πραγματικά επίσης και στην πρωτοπορία κάποιων δραστηριοτήτων που αφορούν και το εμπόριο. Το ας πούμε. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα και οι διάφορες επιτροπές γυναικών εδώ είναι στην πρωτοπορία όσον αφορά όχι μόνο τη συμμετοχή τους σε επίπεδο γεωργίας, αλλά και σε επίπεδο μεταποίησης, Πρόεδρε. Όλα αυτά είναι λοιπόν πολύ σημαντικά, γιατί εμείς συζητάμε εδώ για ευπαθείς ομάδες, As other civil society organization, Uh, in our country uh, as well as uh, Δραστηριοποιούμαστε λοιπόν ε, σε διάφορους τομείς και ο ιδιωτικός τομέας <coughs> συνεισφέρει πάρα πολύ σημαντικά. Ε, επιτρέψτε μου επίσης να πω ότι η κυβέρνηση φυσικά και είναι υπεύθυνη σε τελική ανάλυση και αναλαμβάνει τις ευθύνες ε, των πράξεων και των αποφασεών της. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι διάφοροι διάφορες αυτές οργανώσεις δεν συμμετέχουν στην όλη διαδικασία. Υπάρχει ένας εθνικό φορέας που επιβλέπει όλες τις μη κυβερνητικέ οργανώσει τη ΑΜΟΑ. Και είναι άλλη μια συνεισφορά στην όλη διαδικασία. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ και σε κάτι άλλο που υπόθηκε και αφορά τους περιορισμούς. Να σας πω πως πριν έρθω εδώ, έλαβα μία επιστολή από την πρόεδρο, τον πρόεδρο της ομάδας δεοντολογίας στην οποία επιστολή ως απάντηση της δικής μου επιστολής πέρυσι αναγνωρίζεται η δέσμευσή μου για συνεργασία μαζί με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ανταλλαγή πληροφοριών και σε οποιαδήποτε άλλη αναγκαία δράση. Αυτή η επιστολή εστάλει αφού επισκέφθηκα όλους τους πρέσβεις των ε, κρατών μελών, έτσι ώστε να προσπαθήσω να βάλω το, το όνομα της χώρας μου στη λίστα και να δηλώσω ότι είμαστε δεσμευμένοι για να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία. Επίσης έδωσα την άδεια αυτή η επιστολή να ανέβει στην ιστοσελίδα της ομάδας. Και για μας δεν είναι μείζον θέμα. Φυσικά και είμαστε διατεθειμένοι να συμμορφωθούμε με την ε, διαδικασία. Και φυσικά είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ερωτήσεις που τυχόν έχουν οι ευρωβουλευτές. Και σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Έρια Άσκολα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, καλησπέρα σας. Με χαρά λαμβάνω το λόγο για να σας εξηγήσω κάποιες λεπτομέρειες της Συμφωνίας Οικονομικής Σχέσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη του Ειρηνικού. Η ΣΑΜΟ επιθυμεί να προσχωρήσει σε αυτήν την εταιρική σχέση. Η συμφωνία αυτή εγκρίθηκε το 2011 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για μας το ζήτημα δεν είναι αν η συμφωνία αυτή είναι καλή ή όχι. Το αίτημα έχει γίνει από μια νησιωτική χώρα, μικρή, αναπτυσσόμενη, όπως η Σαμόα, για να προσχωρήσει σε μια υφιστάμενη συμφωνία από την ε, οπτική γωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η πλατφόρμα αυτή μας ε, διευκολύνει και μας δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει διοργανικός και διακρατικός διάλογος. Η ΣΑΜΟΑ θα συμμετέχει ως παρατηρητής μαζί με την παππού Νέα Γουινέα και τα νησιά Φίτζι στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής APA στις Βρυξέλλες 24 Οκτωβρίου. Η ημερήσια διάταξη της ε, συνάντησης αυτής περιλαμβάνει και την βιώσιμη ανάπτυξη και θέματα για την εργασία, αλληλεία, γεωργία κτλ. Επίσης, στην ημερήσια διάταξη θα αναφερθούν οι φορολογικές δικαιοδοσίες που δεν συνεργάζονται. Μη συνεργάσουμε στις φορολογικές δικαιοδοσίες είναι καλύτερο να συζητηθεί αυτό παρά να το αποφύγουμε. Εάν αποκλείσουμε ένα μικρό κράτος όπως η Σαμόα από τη συμφωνία αυτή, θα μας αποτρέψει από το να έχουμε επιρροή στην περιοχή αυτή. περιοχή αυτή δέχεται επιρροές από την Κίνα, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Θα μας δώσει λοιπόν ε, την ευκαιρία να αναθερήσουμε τις ε, αξίες μας και το μηχανισμό λήψης αποφάσεων. Θα έλεγα πως η συμφωνία αυτή δεν αφορά μόνο το εμπόριο, αλλά και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι μια πραγματική εταιρική σχέση. Η συμφωνία αυτή έχει και μια ρήτρα μη εκτέλεσης. Στο άρθρο 73, παράγραφος 2. Αναφέρει ότι κατάλληλα νομικά δεσμευτικά μέτρα μπορούν να ληφθούν υπό τη συμφωνία του Κοτονού σε περίπτωση ε, παραβίασης των ε, στοιχειωδών μερών της συμφωνίας και η συμφωνία εξάλλου του Κοτονού περιέχει μια, έναν παρόμοιο διακανονισμό. Επίσης υπάρχει και μια ρήτρα αναθεώρησης έτσι ώστε να γίνουν τροποποιήσεις με τη λήξη της συμφωνίας του Κοτονού. Υπάρχουν λοιπόν αυστηρές προϋποθέσεις. Η Συμφωνία του Κοτονού παρέχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης των μηχανισμών αυτών, επιβολής κυρώσεων. Φυσικά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να ζυγίσουμε τα υπέρ και τα κατά πρωτού προβούμε σε κυρώσεις. Στο άρθρο 3 της ίδιας της ε, συμφωνίας αναφέρεται ότι τα συμβαλώμενα μέρη θα λαμβάνουν πλήρως υπόψη ε, τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ε, και ανάγκες των ε, συμμετεχόντων και θα προωθήσουν την συμμετοχή και το διάλογο. Ο κύριος πρέσβης, ο οποίος κατέχει και διδακτορικό στην οικονομική ανάπτυξη, ήδη αναφέρθηκε στα κίνητρα της χώρας του για προσχώρηση στη συμφωνία αυτή. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί πως πρέπει να δώσουμε την δυνατότητα στη ΣΑΜΟΑ να προσχωρήσει στη συμφωνία αυτή. Ο αποκλεισμό τη ε, θα απομονώσει ακόμα περισσότερο την οικονομία της από τον υπόλοιπο κόσμο και θα ε, απομακρύνει τη χώρα αυτή από τους ε, διάφορους μηχανισμούς διαλόγου που έχουμε για να προωθήσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ευχαριστώ κύριε Σκολά. Florence. Έχεις κανένα σχόλιο? Ναι. Πολύ γρήγορα. Ευχαριστώ για τις παρεμβάσει, Ευχαριστώ και τον Πρεσβευτή και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να καταστήσουμε κάτι σαφές. Δεν λέει κανείς εδώ ότι ο διάλογος δεν είναι κάτι το θετικό. Είναι θετικό. Αυτό όμως δεν αποκλείει και το άλλο κομμάτι, δηλαδή εργαλεία τα οποία είναι δεσμευτικά και εφαρμόσιμα νομικά. Αυτά πρέπει να συμβαδίζουν. Έτσι όπως έχει το πράγμα τώρα, δεν συμβαδίζουν. Ας πούμε, οι μηχανισμοί επίλυσης διαφορών. Και αυτό ακριβώς ζητάμε. Να υπάρχει διάλογος, ταυτόχρονα όμως να υπάρχει ένα δεσμευτικό κομμάτι πιο αναπτυγμένο, πιο σημαντικό. Εμείς θέλουμε μεγαλύτερη συνεργασία με τους φίλους της ΑΜΟΑ. Θέλουμε όμως η συμφωνία αυτή να τηρεί τους στόχους που έχουμε θέσει. Και αυτή τη στιγμή οι εμπορικέ αυτές συμφωνίες όπως έχουν σχεδιαστεί δεν ανταποκρίνονται στις αρχές που λέμε τώρα ότι συμβαδίζουν με τη Συμφωνία του Παρισιού και τη βιωσιμή ανάπτυξη. Δεν απορρίπτουμε δηλαδή την συμφωνία, αλλά τα κεφάλαια της βιώσιμης ανάπτυξης θα τα ξανανοίξουμε και θα τα κάνουμε δεσμευτικά. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Και έχουμε χρόνο, αλλά έχει έρθει η ώρα η Κομισιόν να δράσει ξεκάθαρα ώστε να αποτελέσουν όλα αυτά καλά προηγούμενα για τις μελλοντικές συμφωνίες. you, our Ευχαριστώ τον εισηγητή, τον κύριο Μαρσελεζή, τροπολογίες και προθεσμία 10 το πρωί 19 του Οκτώβρη η προθυμία για την κατάθεση τροπολογιών. Εντάξει. Okay, everybody. We... Ωραία. Προχωράμε τώρα. Στο σημείο 8 της ημερήσία η κατάσταση των Ροχίνγκια και η προστασία των γυναικών και των κοριτσιών. Την 5η 11 Οκτώβρη θα έχουμε τη Διεθνή Μέρα των Κοριτσιών κάτι το οποίο τονίζει την ανάγκη για αντιμετώπιση των αναγκών και προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα κορίτσια και την πρόθεσή τους ώστε να πετύχουν πλήρη ανθρώπινα δικαιώματα. Η υπόθεση στο Ροχίνγκια είναι δραματική και έχουμε και την διεθνή αποστολή για την ε, Μιανμάρ που αφορά παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σοβαρές παραβιάσεις διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Όλα αυτά αποτελούν σοβαρές παραβιάσεις διεθνούς δικαίου και κατέληξε το πόρισμα της αποστολής ότι η διερεύνηση των εγκλημάτων και η προστασία των στρατιωτικών και παραστρατιωτικών της Μιανμάρ αφορά τρεις κατηγορίες εγκλημάτων διεθνούς δικαίου. Γενοκτονίες, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου. Ιδιαίτερα απεχτής ήταν η χρήση σεξουαλικής βίας ως τρόπος άσκησης εκφοβισμού και τιμωρίας του πληθυσμού, του άμαχου πληθυσμού. Ως αποτέλεσμα αυτής της εκστρατείας, ένα εκατομμύριο άτομα διέφυγαν στα σύνορα με τον Μπαγκλαντές, όπου αυτή τη στιγμή ζουν σε κάποια από τα μεγαλύτερα στρατόπεδα προσφύγων παγκοσμίω. Η κατάσταση σε αυτά τα στρατόπεδα συγκεντρώσεων είναι πολύ κακή. Είδαμε εικόνες από τα στρατόπεδα αυτά να πλήττονται από τους μουσώνες. Και με υπάρχουν βασικής ανάγκης για φαγητό, νερό και προστασία. Πέραν αυτών των φυσικών αναγκών, η βία για στον άμαχο, επί του αμάχου πληθυσμού έχει προκαλέσει τραύματα στα θύματα που χρειάζονται μεγάλη ψυχολογική στήριξη. Για να συζητήσουμε λοιπόν την κατάσταση των Ροχίνγκια και την προστασία των γυναικών και των κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένων και συγκεκριμένων αναγκών, έχουμε εδώ τον Μάρκου Σκίνερ, σύμβουλο πολιτικής για τα θέματα κρίσεως των Ροχίνγκια από τη Διεθνή Επιτροπή Διάσωσης International Rescue Committee, IRC. Ο κύριος Κίνερ θα μας κάνει μια παρουσίαση η οποία θα συμπληρωθεί από τις υπηρεσίες της Κομισιόν και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Επιτρέψτε να κάνω κάποια τελευταία σχόλια πριν δώσω το λόγο στον κύριο Σκίνερ. Λόγω των σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μιαμάρ και στην ε, Καμπότζη, η Κομισιόν εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο άρσης εμπορικής βοήθειας προς την Μιανμάρ και την Καμπότζη. Η υποσυμφωνία τα πάντα εκτός των όπλων, το EBA δηλαδή, που διασφαλίζει μια πρόσβαση ατελώς στις ευρωπαϊκές αγορές για όλες τις εξαγωγές τους εκτός από τα όπλα και τα πολεμοφόδια. Θα δώσουμε τώρα λόγο στον Μάρκο Σκίνερ. Παρακαλώ κύριε Σκίνερ. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε σήμερα στην Επιτροπή σας για να μιλήσουμε για την ε, κρίση αυτή στο πλαίσιο της πολιτικής αντζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα θα μιλήσουμε για την πολιτική προστασία των ε, Ροχίνγκια που είναι κάτι που μας απασχολεί ιδιαίτερα τελευταία. Έχουν καταφύγει στο Μπαγκλαντές ε, πολλοί Ροχίνγκια και οι έρευνες μας έχουν δείξει ε, στοιχεία καταδίωξης, περιθωριοποίησης των Ροχίνγκια και περιπτώσεις ε, βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προτίθεται να δημιουργήσει ένα μηχανισμό αντιμετώπισης και από τις δηλώσεις των ε, Ροχίνγκια αλλά και από τις παρατηρήσεις μας παρατηρούμε ότι η λογοδοσία είναι απαραίτητη έτσι ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν οι Ροχίνγκια στη Μιανμάρ. Επίσης, η Συμβουλευτική Επιτροπή μία συμβουλευτική επιτροπή θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Η Ροχίνγκια και οι συνθήκες διαβίωσης τους εξαρτώνται πάρα πολύ από τις ε, συνθήκες στη χώρα υποδοχή, στην προκειμένη περίπτωση στο Μπαγκλαντές. Πήγα τον Ιούνιο στο Μπαγκλαντές πριν αρχίσουν οι βροχές και κατέστησα σαφές ότι οι μουσώνες μπορεί να έχουν τρομακτικές επιπτώσεις στις εγκαταστάσεις ε, αυτές. Η μουσόνος βέβαια δεν ήταν τόσο έντονη όσο φοβόμασταν, όμως θα μπορούσαν να έχουν δυνητικά άσχημες επιπτώσεις στα, ε, στους καταβλισμούς ε, συγκέντρωσης των Ροχίνγκια προσφύγων. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να έχουμε επίγνωση των κινδύνων που διατρέχουν οι γυναίκες και τα κορίτσια Ροχίνγκια. Είναι το 52% του πληθυσμού εξάλλου ε, οι πιο επικίνδυνε ομάδες είναι οι γυναίκες ή τα κορίτσια που ταξιδεύουν μόνα. Οι κίνδυνοι είναι πολλοί. Είναι, το... είναι η φυγή τους πρώτα απ' όλα. Είναι το καθεστώς του άπατρη. Είναι οι συνθήκες που τους επιφυλάσσει η χώρα υποδοχής, τον Μπαγκλαντές. Διότι παρά το γεγονός ότι στα στρατόπεδα αυτά υποδοχή στο Παγκλαντές ε, η κατάσταση είναι σχετικά ασφαλής. Υπάρχουν κίνδυνοι έμφυλης βίας, σεξουαλικής βίας και δεν έχουν πρόσβαση στο νομικό σύστημα του Μπαγκλαντές εξαιτία της ε, μη ιδιότητας του πρόσφυγα. Τα στρατόπεδα αυτά είναι υπερπλήρη, υπάρχουν προβλήματα με τον φωτισμό, με τις εγκαταστάσεις υγιεινής, με την ίδρευση που κάνουν τη ζωή των Ροχίνγκια στο Μπαγκλατές φυσικά άσχημη, αλλά η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τις γυναίκες και τα κορίτσια. Οι γυναίκες αυτές και τα κορίτσια είναι απομονωμένα, δεν έχουν πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες και πέφτουν θύματα έμφυλης βίας. Τέλος, βλέπουμε πως υπάρχει έλλειψη πρόσβασης στην εκπαίδευση, στην εργασία. Είναι κίνδυνοι που προστίθενται στους ήδη αυξημένους κινδύνους που διατρέχουν οι γυναίκες και τα κορίτσια ροχίνγκια. Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης, ε, διακίνησης, καταναγκαστικών γάμων. Είναι δύσκολη και περίπλοκη κατάσταση και αντιμετώπιση της θα πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να αναγνωρίσουμε την προσφορά του κράτους, του Μπαγκλαντές και της κοινωνίας εκεί, δεδομένης της έκτασης της μασικής εξόδου από τη Μιανμάρ. Υπάρχουν διεθνείς ε, οργανώσεις που δραστηριοποιούνται. Η δική μας, η Διεθνής Επιτροπή Διάσωσης είναι εκεί από τον Αύγουστο και προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και τα κορίτσια λόγω της ιδιαιτερότητάς τους. Επίσης, η εμπειρία μας δεν είναι κατά ανάγκη ενδεικτική της ε, ανθρωπιστικής ε, ανταπόκρισης στο, στην κατάσταση των προσφύγων στο mm-hmm. Μπαγκλαντές. Χρειάζεται αύξηση της ανταπόκρισης και κινητοποίηση διάφορων ε, εταίρων. Ορισμένοι από αυτούς βρίσκονται ήδη εκεί. Το Μπαγκλαντές έχει περιορισμένους πόρους και το νομικό του σύστημα με την ε, καταχώρηση προσφύγων ε, με την πρόσβαση σε νομικές υπηρεσίες είναι αρκετά περίπλοκο. Πολλές φορές οι συνήγοροι που υπερασπίζονται τους πρόσφυγες δεν έχουν πείρα σε περιστατικά έμφυλης βίας. Βλέπουμε ότι ένα χρόνο μετά συνεχίζουν να παρατηρούνται μεγάλες ελλείψεις σε πολλούς τομείς. Υπάρχει έλλειψη εμπειρογνωμοσύνης ε, σε πολλούς τομείς, όπως για παράδειγμα στην αντιμετώπιση των ε, παιδιών προσφύγων, ναι. στην αντιμετώπιση της έμφυλης βίας. Έπειτα βλέπουμε κάποιες ε, πρακτικές οι οποίες απέχουν πολύ από το να χαρακτηριστούν βέλτιστες. Βλέπουμε για παράδειγμα γυναίκες που υποφέρουν ε, από ασυτεία, τις εμποδίζουν οι άνδρες να έχουν πρόσβαση σε τροφή. Αυτό έχει να κάνει με έμφυλη βία και με την έκθεση των γυναικών αυτών σε διάφορα προβλήματα που επιδεινώνει περισσότερο την κατάστασή τους. Όλα αυτά σίγουρα αποτελούν πρόκληση. Θεωρούμε όμως πως ε, η πρόκληση αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί και πως η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο τόσο ως ε, δωρητής όσο και ως διαμεσολαβητής με την κυβέρνηση του Μπαγκλατές και μέσω της δέσμευσή της να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Για παράδειγμα, το σχέδιο δράσης για τα φύλλα προωθεί την ε, πρόσβαση των γυναικών σε υπηρεσίες υγείας, ε, στη δικαιοσύνη η Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της ε, θέσης της και του κύρους της μπορεί να κάνει συστάσεις έτσι ώστε να βελτιωθεί η ικανότητα ανταπόκρισης και τα ζητήματα ισότητας. Θα ήθελα τέλος να καταλήξω ε, αναφέροντας τρεις ε, συστάσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με μια πρωτοβουλία για τη βελτίωση των συνθήκων στα ε, στρατόπεδα αυτά εγκατάσταση των προσφύγων διότι παραμένουν οι κίνδυνοι για τα κορίτσια και τις γυναίκες. Έπειτα, δημιουργία μιας κοινή επιτροπή διαχείριση και δημιουργία ανάπτυξη ικανοτήτων τόσο από την Ευρωπαϊκή, με συμμετοχή τόσο τη Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και του Μπαγκλαντέ. Θα παρέχεται τεχνική υποστήριξη και εμπειρογνωμοσύνη και θα αυξηθεί η θετική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, μακροπρόθεσμες λύσεις, ανταπόκριση στην κρίση. Μέσω μακροπρόθεσμων λύσεων μπορούμε να αντιμετωπίσουμε διαρθρωτικά προβλήματα στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και τα κορίτσια πριν τη μαζική έξοδο των Ορχήν και τον Αύγουστο του 2017 δεν είχαμε απόλυτη εικόνα του πόσο θα επιβάρυνε η μαζική έξοδος αυτή τον πληθυσμό του Μπαγκλαντές. Βλέπουμε όμως ότι οι προκλήσεις είναι μεγάλες. Χρειάζεται λοιπόν να στηρίξουμε τους πρόσφυγες να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα έμφυλης βίας και ισότητας, αλλά και τις επιπτώσεις της κρίσης ε, στους φιλοξενούμενους, στην κοινότητα στον Μπαγκλαντές. Χρειάζεται επίσης ε, να αντλήσουμε βέλτιστες πρακτικές από χώρες που έχουν αντιμετωπίσει στο παρελθόν παρόμοιες κρίσεις, όπως η Ορδανία και ο Λίβανο, στη Μέση Ανατολή. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η δωρεάν ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά όλο το πακέτο. Χρειάζονται διάφορες εμπορικές παραχωρήσεις στην ε, Ιορδανία και τον Λίβανο. Οι εμπορικές παραχωρήσεις προς τις ε, δύο χώρες αυτές βοήθησαν να βελτιωθεί η υποδοχή των προσφύγων, οι υποδομές, η πρόσβασή τους σε εκπαίδευση, υπηρεσίες υγείας, στέγαση κτλ. Μέσω της στήριξή μας στις ε, χώρες που υποδέχονται τους πρόσφυγες ε, θα βοηθήσουμε τόσο τις χώρες αυτές όσο και τους ίδιους τους πρόσφυγες. Μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε ένα παρόμοιο μοντέλο εδώ που σε συνδυασμό με τη διπλωματία θα βελτιώσει την ε, ικανότητα ανταπόκριση στις ανάγκες των προσφύγων γενικότερα και των γυναικών και κοριτσιών ειδικότερα. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ. Όντως η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Ακούσαμε ορισμένα πράγματα από εσά και πρέπει να κάνουμε μεγάλη προσπάθεια για να καλύψουμε καλύτερα το θέμα. Η κυρία Ανδρούλα Καμινάρα τώρα. Έχετε το λόγο κυρία. Σας ευχαριστώ. Θα αποφύγω να επαναλάβω πολλά από αυτά που είπε ο κύριος Σκίνερ και όπου συμφωνώ. Θα ομιλήσω για την κατάσταση στο Μπαγκλαντές και την κατάσταση στην Μιανμάρ, αρχίζοντας από το Μπαγκλαντές. Είναι αληθές ότι πρόκειται για ε, ένα τεράστιο ε, καταβλισμό, μεγαλύτερο στον κόσμο και πράγματι ήμουν εκεί στην εποχή των μουσώνων. Είναι απίστευτη η τροτότητα των ανθρώπων αυτών ολόκληρη περιοχή που τους έχει δοθεί από την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές είναι σε μια περιοχή λόφων που ήταν κάποτε ε, δέντρο φυτευμένη, ήταν δασωμένη. Έκοψαν τώρα τα δέντρα για να βάλουν, να φτιάξουν εκεί τους οικίσκους και τώρα είναι μέχρι τα γόνατα στη λάσπη σε συνθήκες πραγματικά απαράδεκτες. Ήδη λοιπόν έχετε πολύ ευάλωτους ανθρώπους που μπαίνουν πλέον σε μια πολύ ευάλωτη κατάσταση λόγω του τόπου όπου έχουν πλέον βρει κατάλημα. Και αν δείτε την κατάσταση γυναικών και νεαρών κοριτσιών που ακούσαμε ήδη ότι είναι πάνω από το 50% του πληθυσμού αυτού στους καταβλισμούς αυτά λοιπόν τα πρόσωπα αυτές οι γυναίκες και κορίτσια είναι σε ακόμα χειρότερη κατάσταση πήγα και ε, είδα μερικούς από αυτούς τους gender friendly spaces όπου είχαν να μου πούν ε, τρομοκρατικές ιστορίες οι γυναίκες αυτές θα σας πούν ότι έχουν δει μωρά να τα πετάνε στο ποτάμι ή ε, να θανατώνονται συγγενείς τους ή σας μιλούν ακόμη οι ίδιες για το πώς ε, τις εβίασαν με ανέκφραστα πρόσωπα. Ε, μιλούν οι ίδιες με ανέκφραστα πρόσωπα γιατί έχουν βαρύτατους ψυχολογικούς τραυματισμούς. Τώρα υπάρχουν αυτοί οι χώροι που υποτίθεται είναι ασφαλεί για τι γυναίκες σε ορισμένου καταβλισμού, όχι σε όλους. Αυτό πρέπει να βελτιωθεί. Ε, λόγω του τρόπου με τον οποίο ε, διοικούνται αυτά τα camps οδηγούνται σε αύξηση της ε, γενετήσιας βίας από την πλευρά των Παγκλατεσιανών. Είναι χωρισμένοι, είναι χωρισμένοι οι καταβλισμοί σε τμήματα. Υπάρχουν οι μάτζι που είναι ορισμένοι από την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές και έχουν απόλυτο έλεγχο σε έναν αριθμό οικίσκων, ας πούμε, τόσο πάντων δομών όπου ε, ζουν οι Ροχίνγκια. Το βράδυ όμως δεν υπάρχουν πλέον εκπρόσωποι μη κρατικών οργανώσεων και άλλων στους καταβλισμούς. Ο απόλυτος έλεγχος ανήκει πλέον σε κάποιους από αυτούς τους μάτζι. Πρώτο λοιπόν, μια γυναίκα η οποία ε, μπορεί να βιαστεί, δεν πρόκειται να πάει σε έναν άντρα να του πει «Κοιτάξτε, με βιάσανε». Δεύτερο, ακούσαμε και ιστορίες ότι ορισμένοι από αυτούς τους ίδιους που υποτίθεται ότι είναι οι προστάτες των, ε, φυγά, των προσφύγων εμπλέκονται σε οτιδήποτε τέτοια ιστορία. Υπάρχει μια πίεση λοιπόν και μια όθηση για ασφαλείς τόπους. Μιλούμε ήδη με τα Ηνωμένα Έθνη για τον τρόπο αυτό, διότι πρέπει να αλλάξει οπωσδήποτε, οπωσδήποτε ο τρόπος διοίκησης των καταβλισμών. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Ωστόσο, ο συντονισμός μεταξύ ION και Ηνωμένων Εθνών έχει βελτιωθεί από την αρχή του χρόνου, αλλά υπάρχει ακόμα σημαντικός χώρος βελτίωσης. Είναι αλήθεια επίσης και συμφωνώ με τον κύριο Σκίνερ ότι ακούμε όλο και περισσότερο για βία μεταξύ ε, συζύγων ή εν πάση περιπτώσει συντρόφων. Κάτι το οποίο είναι απολύτω αδικαιολόγητο, αλλά κάτι που βλέπουμε όταν, άνθρωποι, όταν ζουν άνθρωποι σε πολύ ε, στενούς περιορισμούς και ε, άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι σε πάρα πολύ περιορισμένο χώρο που δεν τους επιτρέπεται η έξοδος, δεν τους επιτρέπεται να κάνουν τίποτα. Αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε. Partner violence αλλά δεν μιλούμε μόνο για partner violence. Υπάρχουν και κάποια θετικά αποτελέσματα, θετικά παραδείγματα. Ορισμένοι εκ των Ροχίνγκια μένουν σε σπίτια, σε κοινότητες εκτός καταβλισμών. Πήγα και είδα μερικούς από αυτούς όπου βοηθούμε, όχι μόνο τους Ροχίνγκια βέβαια, αλλά ολόκληρη την κοινότητα, ώστε να ζουν Ροχίνγκια με τους υπόλοιπους δίπλα-δίπλα, πόρτα-πόρτα. Και ήταν και εκπρόσωποι των καταβλισμών εντός εισαγωγικών και κάτι που με εντυπωσίασε ήταν ότι και ο εκπρόσωπος των Ροχίνγκια και ο εκπρόσωπος των Τόπιων μας ζητούσαν να προσφέρουμε κάποιο είδους εκπαίδευση στα νεαρά κορίτσια μεταξύ 12 και 18 ετών για διάφορους λόγους Αφενός για να μπορέσουν να, να ε, κερδίσουν κάποια χρήματα. Διότι μετά τα 12-13 συνήθως δεν τους επιτρέπεται να βγαίνουν από τα σπίτια τους. Επίσης, όπως μας είπαν, για να συγκεντρώσουν κάποια χρήματα για να μπορέσουν να παντρευτούν να φτάσουν στα 18. Ένα από τα θέματα που τους ενδιαφέρουν, τους απασχολούν πολύ. Πάντως, η πρόσβαση στην εκπαίδευση των νεαρών κοριτσιών είναι κάτι που και οι δύο κοινότητες μας το ζήτησαν. Η εκπαίδευση και, και πάλι συμφωνώ ότι είναι ένα από τα μείζωνα θέματα από τα λίγα που μπορούσαμε να προσφέρουμε στον χώρο της εκπαίδευσης, διότι υπάρχουν και περιορισμοί σχετικά με το τι είδους εκπαίδευση μπορεί να προσφερθεί στα παιδιά Ροχίνγκια. Από τα λίγα που μπορέσαμε να προσφέρουμε, είναι όμως όχι στη γλώσσα των Ροχίνγκια ούτε στα, στη γλώσσα Μπάνγκλα, που είναι η γλώσσα του τόπου όπου ζουν τώρα, πρέπει να είναι στη βιρμανική γλώσσα, που τα περισσότερα από τα παιδιά αυτά δεν έχουν ακούσει ποτέ. Έχουν λοιπόν μια γλώσσα την οποία μιλούν στο σπίτι, όπως μιλούν δηλαδή με τους γονείς τους, δεν μαθαίνουν ούτε τη γλώσσα της χώρας όπου ζουν τώρα και μαθαίνουν μια τρίτη γλώσσα που ενδεχόμενα να τους φανεί χρήσιμη κάποτε ενδεχομένω όχι. Εάν παραταθεί η κρίση, τότε το να μαθαίνουν την βιρμανική γλώσσα δεν τους εξυπηρετεί σε τίποτα. Έχοντας όμως πει αυτά τα πράγματα, η κυβέρνηση Μπαγκλαντέ αξίζει συγχαρητήρια που δέχτηκε τόσους πολλούς πρόσφυγες. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι επέτρεψαν στου πρόσφυγες αυτού να εισέλθουν στο εδαφο τους, στο έδαφο του Μπαγκλαντέ. Ορισμένα όμως από τα θέματα αυτά και το ζήτημα της εκπαίδευσης και ποια γλώσσα, σε ποια γλώσσα τα εκπαιδεύονται τα ε, νέα αυτά παιδιά και ιδίως τα κορίτσια, πρέπει να αλλάξουν. Σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική έκκληση που έγινε για ανταπόκριση στις ανάγκες των Ροχίνγκια στο Μπαγκλαντές, Υποσχέθηκαν συνολικά οι δωρητέ 950 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο 34% όμω δόθηκαν τελικά. Άρα υπάρχουν ακόμα τεράστιε ανάγκε. Και αυτό είναι ένα από τα θέματα που δεν μας επιτρέπουν να αντιδράσουμε συλλογικά, η διεθνής ανθρωπιστική κοινότητα δηλαδή, να αντιδράσει σε συλλογικό επίπεδο και να ε, βελτιώσει την κατάσταση και των γυναικών, διότι υπάρχει ένα χρηματοδοτικό κενό τεράστιο η Κομισιόν. Τους τελευταίους 12 μήνες που έχει χτυπήσει η κρίση έχει διαθέσει 65 εκατομμύρια ευρώ. Για την πλευρά του Μιανμάρ, γιατί υπάρχουν και στην Μιανμάρ. Περίπου 600.000. το, στο, στην περιφέρεια Ράκα. Δεν είχαμε δεν είχαμε, δεν είχαμε, δεν έχουμε, έχει βελτιωθεί η πρόσβαση από αυτήν του Αυγούστου 2017 και 6.000 6.000 που είναι παγιδευμένοι σε ένα είδος ε, no man's ε, αυτή λέγεται zero line ε, μεταξύ των δύο χωρών τα πρόσωπα αυτά ε, είναι εκεί κάποιο διάστημα ήδη και δεν είναι γνωστή η μοίρα τους. Τώρα, για την κατάσταση Ροχίνγκια στην πλευρά της Μιανμάρ. Οι περισσότεροι ζουν πάλι σε ανοιχτούς καταβλισμούς, αλλά όχι ακριβώς, διότι δεν έχουν ελεύθερη κυκλοφορία, ελευθερία κυκλοφορίας. Προσφέρεται βοήθεια διότι η κυβέρνηση της Μιανμάρ δεν έχει επιτρέψει την καταγραφή των προσώπων αυτών. Έκαναν μια καταγραφή όταν φτιάχτηκαν οι μεγάλοι καταβλισμοί, αλλά συνέχισαν να έρχονται άνθρωποι στους καταβλισμούς αυτούς. Τώρα για τις μερίδες που δίνονται τροφίμων κλπ. Ε, πολλοί από αυτούς δεν έχουν πρόσβαση σε, αυτές, σε αυτού του είδου τη διατροφή. Και πάλι και εκεί υπάρχουν ε, προβλήματα γενετήσια βία απέναντι στις γυναίκε και τα κορίτσια στου καταβλισμούς αυτούς και οι περισσότερε από αυτέ ζουν σε κάτι μακρόστινε παράγκες που φτιάχτηκαν πριν από 4-5 χρόνια διότι η λογική ήταν ότι ίσως χρειαστεί να διαμείνουν εκεί 6 μήνες, ένα χρόνο οι περισσότερες από αυτές έχουν ήδη αρχίσει να καταραίουν, έχουν ε, πάρει μια λοξή, μια ε, λοξή θέση και τις ενισχύουν με διάφορα δοκάρια. Σε ορισμένα από τα κορίτσια, μετά από κάποια ηλικία, όπως είπα πριν, δεν επιτρέπεται καν να βγουν από τις παράγκες αυτές. Επομένως τελικώς οι γυναίκε των Ροχίνικα και από τις δύο πλευρές του συνόρου είναι οι πιο ευάλωτε. Εμεί τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε στοχεύσει πολλά από τα έργα που κάνουμε με συνεργασία εταίρων μας στοχευμένα τα προγράμματα αυτά στην προστασία γυναικών και κοριτσιών. Όμως προφανώς αυτά τα πράγματα δεν αρκούν. Πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα και από τις δύο πλευρές για να βελτιωθεί η ζωή των γυναικών και των νεαρών κοριτσιών. Από την πλευρά τη Μιανμάρ πάντα. Α, ναι, τελειώνω, τελειώνω. Είδαμε μια ελαφρά βελτίωση της πρόσβασης, όμως εξακολουθεί να είναι πολύ χειρότερη από αυτή που ήταν πριν από ένα χρόνο. Και επειδή μιλούμε για Μιανμάρ, δεν πρέπει να ξεχνούμε και άλλη κρίση εκεί, στη, στο, στην επαρχία Κατσίν. Μόλις τον Αύγουστο αναγκάστηκαν 100.000 πρόσωπα να εγκαταλείψουν τι αιστείε τους και διαβιούν τώρα στις ίδιε άσχημες συνθήκες όπως η Ροχίνγκια στην ε, Ράκα. Θα περιοριστώ σε αυτά. Και σε ό,τι αφορά τώρα τον πληθυσμό υποδοχής, τονίζω ότι δεν πρέπει να λησμονούμε και αυτόν τον πληθυσμό ο πληθυσμό δηλαδή που υποδέχεται τους πρόσφυγε αυτούς, γιατί οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί είναι πάρα πολύ φτωχοί και χρειάζονται ενίσχυση και βοήθεια. Σα ευχαριστώ πολύ κυρία Καμινάρα, λέει η πρόεδρο, για ε, την περιγραφή της κατάστασης. Θα δώσω το λόγο τώρα στην Ισαβέλα Ντελάτρα. Ορίστε κυρία. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη και να συμπληρώσω αυτά που ήδη υπόθηκαν. Θα εστιάσω στο πολιτικό σκέλος. Να επαναλάβω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Παριεκπρόσωπος συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις μέσω της ανάπτυξης συστημάτων αντιμετώπισης της κρίσης αυτής στον Παγκλαντές αλλά και στη Μιανμάρ. Αυτό ήταν και το θέμα συζήτησης στις τελευταίες μας συναντήσεις. Τον Ιούλιο έγινε μια πολιτική διαβούλευση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μπαγκλαντές. Συζητήθηκε το θέμα αυτό. Πιο πρόσφατα έγινε μια συνάντηση ανάμεσα στην ΥΠΑΤΕ εκπρόσωπο και στον ε, Πρωθυπουργό του Μπαγκλαντές και συζητήθηκε η ανθρωπιστική κρίση των Ροχίνγκια και σε λίγες μέρες στη Σύνοδο εδώ στις Βρυξέλλες θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το θέμα. Υπάρχει σαφής πολιτική δέσμευση λοιπόν. Και έχει εγκριθεί ένα ψήφισμα στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την λογοδοσία 27 Σεπτεμβρίου ψηφίστηκε για τη δημιουργία ενός μηχανισμού λογοδοσίας βασισμένου σε αυτό. Φυσικά θα χρειαστεί καιρός να φτάσουμε σε διώξεις. Γι' αυτό θα πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στα Ηνωμένα Έθνη έτσι ώστε να εξετάσουμε και πιθανότητες χρηματοδότησης. Μετά, στην έκθεση θα γίνει αναφορά σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, μέχρι και σε γενοκτονία σε ορισμένα σημεία της Μιανμάρ. Και είναι σαμφές ότι η διεθνής κοινότητα ασκεί πιέση στη Μιανμάρ και η πίεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για να βρεθεί λύση που θα αντιμετωπίσει τα αίτια της κρίσης στην μόνο οι λύσεις που, αναφέρ, τα αίτια που αναφέρονται στην έκθεση ΑΝΑΝ θα μπορέσουν να αντιμετωπιστούν και να οδηγηθούμε σε λύσεις στην κρίση αυτή. Θα χρειαστεί επίσης να δοθεί έμφαση στην επόμενη φάση της ε, συνεργασίας και βοήθειας Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην Μιανμάρ. Η Ροχίνγκια είναι για αρκετό καιρό στο Μπαγκλαντές. Οι αρχές επίσημα δεν έχουν αναγνωρίσει ότι υπάρχει πρόβλημα. Δεν πρέπει να είμαστε και πολύ αισιόδοξοι ως προς αυτό το θέμα. Ε, κάτι θετικό ήταν και η υποδοχή της ειδική απεσταλμένης των Ηνωμένων Εθνών που θα δημιουργήσει, που θα, που θα έχει μια βάση στον επιτό, θα έχει ένα γραφείο. Και εδώ λοιπόν έχουμε επιτέλους φως στο τούνελ. Για πολλά χρόνια δεν είχαν τη δυνατότητα οι ειδικοί συγητές να πάνε στη Μιανμάρ, δεν ήταν ευπρόσδεκτοι, δεν μπορούσαν να γίνουν διερευνητικές αποστολές. Να αναφερθώ επίσης σε ένα project αξίας 50 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο στοχεύει τόσο τους πρόσφυγες αλλά και τις κοινότητες που τους υποδέχονται. Δίνεται έμφαση στην εκπαίδευση, στην επισητιστική ασφάλεια μεταξύ άλλων, η οποία είναι το μίσο που αναφέρθηκε πως υπάρχει ανάγκη βελτίωσης. Φυσικά το ποσό αυτό δεν είναι αρκετό, όμως μπορούμε να βελτιώσουμε τη χρηματοδότηση. Επίσης υπάρχουν διάφορα project μικρής κλίμακας για να αποτραπεί η ριζοσπαστικοποίηση των ε, νέων στα, στους καταβλισμούς αυτούς. Επίσης, διάφορα άλλα προγράμματα και μέτρα, τα οποία δεν αφορούν άμεσα τους ε, πρόσφυγες που βρίσκονται στους καταβλισμούς, αλλά και οι οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών, υπερμάχους ανθρώπινων δικαιωμάτων και αφορούν την καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Ίσως λοιπόν θα μπορούσαν και στο μέλλον να χρησιμοποιήσουν αυτές τις δυνατότητες για άλλους σκοπούς. Ευχαριστώ. Τώρα θα δώσω το λόγο στους ευρωβουλευτές. Πρώτα στον κύριο Γκερέρο Σαλό. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Προεδρεύουσα, και ευχαριστώ αυτούς που μας ενημέρωσαν τη διεθνή διάσωση δηλαδή την Κομισιόν και την Εξωτερική Υπηρεσία. Και τις μαρτυρίες για τα δεκτονόμενα στην περιοχή που αναφέρονται σε γενεοκτονίες και σε βία κατά γυναικών και κοριτσιών και που μας περιέγραψαν μια κατάσταση που θα μπορούσαμε να δούμε στα κοινωνικά δίκτυα ή στα ΜΜΕ αλλά εν Πρόκειται για οργανισμούς που είναι παρόντες εκεί. Το πρώτο που θα πρέπει νομίζω να λάβουμε υπόψη μας είναι ότι οι Ροχίνγκια που πήγαν στο Μπαγκλαντές αντιστοιχεί στα άτομα που έφτασαν στις ευρωπαϊκές ακτές μετά το πόλεμο στη Συρία. Θέλω να τονίσω ότι αν εμείς αντιμετωπίσαμε τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε με την άφηξη αυτών των ατόμων, τότε εύκολο, εύκολο μπορεί κανείς να φανταστεί τι σημαίνει αυτό για το Μπαγκλαντές. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο φιλοξενών πληθυσμός δεν είναι ο πλούσιος πληθυσμός της Ευρώπης, αλλά Πληθυσμό βρίσκεται στην ίδια κατάσταση φτώχειας με εκείνε τι περιοχές της Μιανμάρ. Οπότε οι εκκλησει που ακούσαμε από όλου του εισηγητέ ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε την κατάσταση που αντιμετωπίζει τον Μπαγκλαντές και να καταλάβουμε ότι είναι στρατηγική επιλογή η βοήθεια του Μπαγκλαντές για την αντιμετώπιση αυτής της ανθρωπιστικής κρίσης. Νομίζω ότι αυτό είναι κέρια σημασία για να κατανοήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα φτώχειας που αφορούν την χώρα υποδοχής και τους πληθυσμούς υποδοχής. Κατά δεύτερο λόγο, είπαμε ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε πράγματι με την παροχή τροφίμων, στέγης, η κλασική δηλαδή η ανθρωπιστική βοήθεια, να βοηθήσουν λοιπόν αυτούς τους πληθυσμούς Ροχίνγκια. Επίσης όμως είπαμε ότι θα πρέπει να δράσουμε πολιτικά και νομικά και στρατηγικός γενικότερα. Και ακούσαμε και κάποιες προτάσεις που διατυπώθηκαν. Ας πούμε να αξιοποιήσουμε τις εμπειρίες του Λιβάνου και της Ιορδανίας αμφίδρομα, ώστε δηλαδή και να πιέσουμε την Καμπότζη και την Μιανμάρ αρνητικά κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή να παγώσουμε προτιμήσεις αν δεν προχωρήσουν στα θέματα τα ανθρωπιστικά, αλλά ταυτόχρονα προς τον Παγκλαντέ με θετικό τρόπο, δίδοντάς του προτιμήσει εμπορικού ή οικονομικού τύπου, λόγω της ανάγκης που αντιμετωπίζουν με αυτό τον εκτοπισμένο πληθυσμό από τη Μιαμάρ. Κατά τρίτο λόγο, έχουμε το θέμα αυτών των δράσεων που παραβιάζουν ανθρώπινα δικαιώματα και αφορούν μορφές γενοκτονίας ή επιθέσεις κατά της σεξουαλικότητας των δικαιωμάτων των γυναικών. Όλα αυτά δεν μπορούν να μείνουν ατιμόρυτα. Και αν πράγματι η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ έχει αρχίσει να διαβλέπει τη δυνατότητα για να αποδοθούν ευθύνες νομικές, το ίδιο θα πρέπει να κάνει και Ένωση ώστε να πάμε στα διεθνή δικαστήρια σε σχέση με τη στάση της Μιαμάρ προς αυτούς τους πρόσφυγες. Όλοι ξέρετε, όσοι παρακολουθείτε τις συζητήσεις μας, ότι η Επιτροπή μας είχε ιδιαίτερη εγκύτητα με τα θέματα τα εκπαιδευτικά εν προκειμένου ενός εκατομμυρίου ατόμων. Τα άτομα αυτά που δεν ξέρουμε αν θα έχουν μέλλον ή όχι, θα πρέπει να τους προσφέρουμε ευκαιρίες εκπαίδευσης ώστε να ανταχθούν στην ενεργό ζωή και αυτό προς τον Μπαγκλαντές και σε άλλες χώρες της περιοχής. Αυτό νομίζω είναι μια στρατηγική χειρονομία, γιατί όσο πήγαμε σε καταβλισμού, νομίζω ότι όλοι από εδώ την Επιτροπή μας έχουν αντίστοιχη εμπειρία, είδαμε λοιπόν ανέκαθεν ότι οι οικογένειε θα θέλαν να λάβουν παιδεία τα παιδιά τους και ευκαιρίες. Και για την παιδεία, μάλιστα, μέσω συμφωνιών διαφόρων ειδών πετύχαμε χώρες όπως η Ορδανία, οι οποίες έθεταν φραγμούς στην εκπαίδευση μικρών παιδιών, προσφύγων, άλλαξαν τις τάσεις τους. Οπότε θα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή την εμπειρία και σε αυτή την περίπτωση. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρος. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε αργήσει 10-15 λεπτά σε σχέση με το χρονοδιαγραμμά οπότε σας παρακαλώ να είστε σύντομοι. Σεσίλια Κένια, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ και εγώ να ευχαριστήσω τους τρεις εισηγητές μας για τις πληροφορίες τους που ενισχύουν τα πιθανά μας εργαλεία ώστε να δοθεί μια λύση θα είμαι σύντομη, επειδή πολλά που θέλω να πω υπόθηκαν από τον προλαλήσαντα συνάδελφο που χαίρομαι που τα ανέφερε. Ξέρουμε ότι οι εκτοπιστέντες είναι γύρω σε 700.000 και τα θύματα 24.000. Όπως είπατε όμως, θέλουμε μια ολιστική προσέγγιση και οι λεπτομέρειες εδώ που δώσατε είναι αξιόλογες και πολιτικά αλλά και ανθρωπιστικά για οικονομική ενίσχυση. Οπότε χρειαζόμαστε καλές πρακτικές όπως στην περίπτωση του Λιβάνου και της Ιορδανίας ώστε να μεταφέρουμε αυτή την εμπειρία σε αυτή την περίπτωση για αντίστοιχε περιπτώσεις διαθρωτικής κρίσης μακροπρόθεσμης που δεν μπορούν να λυθούν άμεσα. Έχουμε τη λύση του Μπακλαντές που προτείνει την μεταφορά 100.000 ατόμων σε ένα νησί που λέγεται Μπασαντσάρ. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες λεπτομέρειες γι' αυτό. Αυτό θα είχα μόνο να ρωτήσω. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Τι ωραία που είναι η πρόεδρός μας εδώ, Λίντα Μακάβαν. Έχεις το λόγο, Λίντα. Να, α, όχι, δεν, δεν ζήτησες να λάβεις το λόγο. Καλά. Βέβαια, έχω μια ερώτηση, λέει η Λίντα Μακάβαν, όταν έφτασα ε, την ώρα που μιλούσε η Ανδρούλα. Ε, είπατε ότι τη νύχτα οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, δεν είναι πλέον παρούσες στους καταπλησμούς Αυτό συμβαίνει αλλού και είναι σύνηθες. Πρόεδρος, ωραία τότε θα ακούσουμε τις απαντήσεις και πρώτα από τον κύριο Σκίνερ. Ευχαριστώ σύντομα. Ανθρωπιστική βοήθεια και πολιτική δράση. Χαίρομαι πολύ που τα άκουσα αυτά τα πράγματα. Και αυτή είναι μακροπρόθεσμα η σωστή ε, στάση για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των Ροχίνγκια και να ενισχυθεί η αυτοδιάθεσή τους κατά κάποιο τρόπο. Χρειάζεται να ανοίξει ο χώρος αυτός, να δημιουργηθεί και περισσότερη χρηματοδότηση και για το ερώτησή σας για το νησί Μπασαντσά έχουμε όντως σημαντικές ανησυχίες να πάνε πρόσφυγες σε ένα τέτοιο νησί στον κόλπο της Βενγάλης και δεν υπάρχει αξιολόγηση των συνθήκων ακόμα και είναι αδύνατο να σχολιάσουμε για τον λόγο αυτό. Όμως θα χρειαστεί συντονισμένη και συνεκτική στάση της διεθνούς κοινότητας απέναντι ε, στην πρόταση αυτή. Για την ώρα υπάρχει μόνο θέση των ΗΕ. Εθνών, αλλά δεν υπάρχει συντονισμός της δράσης της ε, διεθνούς κοινότητας. Πολύ δύσκολο Βέβαια είναι και δύσκολο να αρνηθούμε τη λύση αυτή όταν ζητούμε να ε, μειωθούν οι πληθυσμοί των καταβλισμών. Η κυρία Καμινάρα, να απαντήσω αν μου επιτρέπετε σε ορισμένε από τις ερωτήσεις και πρώτα θα ήθελα να σας παραθέσω ένα τμήμα από την έκθεση που νομίζω ότι δίνει κανείς να καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Λέει λοιπόν ότι συνεχίζεται στην ουσία η γενοκτονία. Δεν είναι κάτι το οποίο συνέβη και τελείωσε και τώρα βλέπουμε τα αποτελέσματα. Δεν βρίσκω δυστυχώς ακριβώς ε, το σημείο αυτό στη σημειώσεις μου. Αυτό που λέει όμως είναι ότι η επίθεση κατά τον Ροχίνγκια από την πλευρά της Μιανμάρ έχει αρχίσει αλλά συνεχίζεται. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να ε, θυμούμαστε συνεχώς όταν προσπαθούμε να αποτιμήσουμε ε, το τι υφίσταται η Ροχίνγκια από την πλευρά της Μιανμάρ. Ε, για θέματα τώρα εκπαίδευσης και μέσω μακροπρόθεσμα, ένα από τα project που χρηματοδοτούμε είναι μαζί με τον IOM, όπου και κοινότητες υποδοχής και ε, πρόσφυγες συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα δενδροφύτευσης για να καταπολεμηθεί η αποψήλωση. Διότι ένα από τα προβλήματα των καταβλισμών αυτών είναι ότι αποψηλώθηκαν οι λόφοι ε, μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και τώρα ε, τα νερά της βροχής παρασύρουν το χώμα και ε, τους πνίγουν τους ανθρώπους, κάνουν πλημμύρες. Δεν είναι κάτι ακριβώς σαν εξασφάλιση απασχόλησης, πάντως τους δίνουμε κάτι να κάνουν, εξασφαλίζοντας και ταυτόχρονα μια προστασία απέναντι στις κλιματικές αλλαγές μέσω μακροπρόθεσμα. Συμφωνώ επίσης στην ανάγκη να αποδοθεί προσοχή και στις ε, κοινότητες υποδοχής. Για ένα απλό λόγο, αν δεν αποδοθεί προσοχή στην ε, κοινότητα υποδοχής που βλέπει δίπλα τους πρόσφυγες να λαμβάνουν ας πούμε μερίδες φαγητού ή πράγματα άλλα τα οποία ίδια δεν έχουν. Οι ίδιοι, οι ίδιοι οι ντόπιοι δηλαδή δεν έχουν. Ε, έστω και για λόγου πρόληψη οφείλουμε να το αντιμετωπίσουμε διότι αλλιώ πιθανά θα προκαλέσουν μια κατάσταση όπου η, η κοινότητα υποδοχή αναπτύσσει αρνητικά συναισθήματα απέναντι στους πρόσφυγες. Όταν έγινε η πρώτη εισρωή των προσφύγων, οι ντόπιε κοινότητε φάνηκαν πολύ γενναιόδορε και του ε, βάζανε στα σπίτια του. Δεν είχαν βέβαια αρκετό φαγητό να του δώσουν, αλλά ε, ε, προσπαθούσαν. μοιράζονταν το λιγοστό φαγητό του μαζί του. Αυτό πρέπει να συνεχιστεί. Να μην ανατρέψουμε αυτή την τάση με τη δική μα συμπεριφορά. Τώρα, για την γενετήσια βία. Δεν μπορεί να παραμείνει ατιμόρυτη, συμφωνώ απόλυτα και γι' αυτό άλλωστε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταβάλει προσπάθειες και κινεί όλη αυτή τη διαδικασία για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό. Και ναι, μπορούμε να διδαχτούμε από άλλες συγκρούσεις που προκαλούν μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών και τα διδάγματα αυτά να τα εφαρμόσουμε στη συγκεκριμένη κρίση. Τώρα για το νησί. Ήδη από πέρσι, όταν έγινε η μαζική μετακίνηση, η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές είπε αμέσως ότι θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει τις αναγκαίες συνθήκες ώστε να μπορέσει να μεταφέρει τις πρόσφυγες εκεί. Βέβαια, η ανθρωπιστική κοινότητα αντέδρασε, υπενθυμίζοντας ότι οι αρχές ελεύθερης κυκλοφορίας των ανθρώπων πρέπει να ληφθούν υπόψη ότι το νησί εν μέρη πλημμυρίζει από τα νερά της θάλασσας Μέχρι τώρα λοιπόν δεν έχουν μετακινηθεί άνθρωποι εκεί. Όμως η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές φτιάχνει εκεί κάποιες κατασκευές. Το επόμενο βήμα υποτίθεται θα είναι ότι θα επιτρέπεται εκπρόσωποι μη κρατικών οργανώσεων να επισκεφθούν το νησί για να δουν αν είναι κατάλληλες συνθήκες. Ελπίζουμε λοιπόν να μην δούμε μαζικές μετακινήσεις προσφύγων. Αλλά αυτή η υπόθεση του νησιού εξακολουθεί να είναι επιτάπητος. Οι αριθμοί ανθρώπων κάποτε μιλούσαν για 100.000, αλλά μιλούσαν επίσης και για άλλους αριθμούς. Είναι φυσιολογικό τη νύχτα να μην είναι κανείς. Αν δείτε τους καταβλισμούς στη Βόρεια Ράκα υπάρχει και απαγόρευση κυκλοφορίας τη νύχτα. Αν ένα παιδί, μια γυναίκα, μια, μια γυναίκα, αν γεννήσει μέσα στη νύχτα, δεν επιτρέπεται να φύγει από τον καταπλησμό. Κανεί άλλο δεν μπορεί να πάει να την βοηθήσει μέχρι να ξημερώσει. Δεν λέω λοιπόν ότι, ε, ότι είναι σύνηθε. Όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι συνήθι, δεν είναι ομαλά, αλλά είναι και η πρώτη φορά που το βλέπουμε. Από τη στιγμή που ε, δεν έχει κανείς πρόσβαση σε κάποιο τόπο, αυτό οδηγεί σε αύξηση της βίας, σε αύξηση της γενετήσιας βίας, σε αύξηση της τρομοκρατίας. Είναι πράγματι πολύ λεπτή ισορροπία να τηρήσει κανείς, δηλαδή να συνεχίσουν οι ΜΚΟ να είναι επιτόπου, να ζητούν ανάληψη δράσης, αλλά δεν μπορούν να πούν και να, μέχρι εδώ, ως εδώ και με παρέ και φεύγω. Δεν μπορούν να βάλουν κόκκινες γραμμές, όπως λένε. Ευχαριστώ. Yes, thank you. Um, just on the account... Ευχαριστώ πολύ για τη λογοδοσία. Θα ήθελα να αντιδράσω στο σχόλιο του αγαπητού Ευρωβουλευτή πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο. Νομίζω η παρουσίαση του ψηφίσματος στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ήταν σαφής. Το ψήφισμα αυτό παρουσιάστηκε από κοινού με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ε, IOC Βλέπουμε λοιπόν πως η πίεση προέρχεται από τη διεθνή κοινότητα, όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η πίεση αυτή είναι ένα από τα ισχυρότερα όπλα που διαθέτουμε προς ε, τη Μιανμάρ. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε έναν μηχανισμό για λογοδοσία, το οποίο, ο οποίος θα μας επιτρέψει τη συλλογή στοιχείων, την ενοποίησή τους και τη διατήρησή τους. Ε, μιλάμε για στοιχεία που αφορούν εγκλήματα, τα οποία διαπράχθηκαν και συνεχίζουν να διαπράττονται στη Μιανμάρ, έτσι ώστε στο μέλλον να υπάρχει δυνατότητα να ασκηθούν ποινικές διώξεις. Επίσης, ξεκίνησε μία προκαταρκτική εξέταση για τις απελάσεις Ροχίνγκια από την Μιανμάρ και η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τη δράση της Επιτροπής αυτής. Ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε να κλείσουμε το θέμα αυτό, να σας ευχαριστήσω όλους για την ανταλλαγή απόψεων και θα δώσω τώρα το λόγο στην πρόεδρό μας, Λίντα. Καλώς ήρθες. Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Okay, colleagues, my apologies. Συνάδελφοι, ζητώ συγγνώμη που δεν ήμουν εδώ από την αρχή. Το έχουμε ζήσει όλοι αυτό, τρένα που καθυστερούν. Αυτό συνέβη και σε μένα, έχασα το Eurostar και έπρεπε να περιμένω δύο ώρες στο Λονδίνο για το επόμενο. Η Μύρια έκανε εξαιρετική δουλειά ως ε, αντιπρόεδρος. Παίρναμε λοιπόν ε, στο επόμενο θέμα. Έχουμε καθυστερήσει κιόλα, γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε σύντομοι. Θα μιλήσουμε για τον σεισμό και το τσουνάμι στην Ινδονησία. Βλέπω ότι υπάρχουν 1.350 ε, επιβεβαιωμένοι νεκροί και χιλιάδες αγνοούμενοι. Έχουμε και την εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης ΕΚΟ που θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για το τι γίνεται και τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Αν δρούλα, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ, Λίντα. Πράγματι, τα νούμερα αλλάζουν συνεχώς. Επίσημα, η νεκροί χθε ήταν 1763, όμως ε, υπάρχουν αναφορές στα μέσα ενημέρωσης που μιλάνε για πάνω από 5.000 και ακόμα περισσότερους εκτοπισμένους. Έχουν αρχίσει και φτάνουν ορισμένες εικόνες από ένα χωριό όπου στην ουσία η γη γίνεται λάσπη ρευστοποίηση, κάπως έτσι το λένε. Η γη κατάπιε ένα ολόκληρο χωριό. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να υπολογίσουμε τον ακριβή αριθμό των θυμάτων. Τι κάνει εν συντομία Ευρωπαϊκή Ένωση. Κινητοποιήσαμε 1,5 εκατομμύριο ευρώ το οποίο αυτή τη στιγμή έχει ήδη χορηγηθεί. Είμαστε σε επαφή με την κυβέρνηση της Ινδονησίας η οποία έχει δηλώσει πως θα χρησιμοποιήσει τον ρυθρό Σταυρό της Ινδονησίας για ε, διάσωση και πέρα από τη δική μας χρηματοδότηση τα κράτη-μέλη έχουν διαθέσει περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ. Τι κάνουν λοιπόν τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, έχουν διαθέσει περίπου το 1 πέμπτο τη ε, διεθνού χρηματοδότηση, που ανέρχεται στα 50 εκατομμύρια. 10 λοιπόν εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε επί τόπου τον κόσμο. Επανενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός Κοπέρνικος για την αντιμετώπιση περιπτώσεων εκτάκτου ανάγκης Υπάρχουν λεπτομερείς χάρτες, έχει ενεργοποιηθεί επίσης και ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ένωση. η Δανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο ανταποκρίθηκαν στην ενεργοποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και παρέχουν στήριξη σε θέματα έλλειψης ενέργειας και στέγασης με σκηνές, με έργα συντήρηση Η Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ επίση χρηματοδοτεί εδώ και αρκετό καιρό κάποια άλλα προγράμματα και έργα, πρωτοβουλίε για μείωση του αντικτύπου καταστροφών. Το 2013 ξεκινήσαμε δουλειά σε αυτά τα project, όμως από ό,τι μας ε, πληροφορούν θα ε, μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί τα κονδύλια διαφορετικά. Θα σταματήσω όμως εδώ, δεν θα συνεχίσω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Η ετοιμότητα βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Θα δώσω όμως το λόγο στους συναδέλφους, τον Ενρίκε Γκερέρο, ο οποίος είναι ο ε, εκπρόσωπος για ανθρωπιστικά θέματα. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Ακούσαμε ότι ακόμα δεν γνωρίζουμε την πλήρη διάσταση της θεομηνίας. Δηλαδή, κάθε μέρα μαθαίνουμε περισσότερα στοιχεία για τα θύματα και το εύρος της καταστροφής. Είδα χθε εικόνες ακριβώς για το πώς μετακίνησαν τα τα ολόκληρες περιοχές, όχι μόνο με νεκρούς, αλλά και άστεγους μέσα σε μια δραματική κατάσταση σε περιοχές που ακόμα δεν είναι γνωστές και που μόνο μέσα δορυφορικών συστημάτων έχουμε μια εκτίμηση του εύρους της καταστροφής. Δεν μπορούμε λοιπόν παρά να καλέσουμε την Κομισιόν να συνεχίσει να παρακολουθεί την κρίση αυτή και να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να την αντιμετωπίσουμε. Um, Ευχαριστώ πολύ. Αν δεν έχει άλλο συνάδελφο ερώτηση, θα ήθελα και εγώ να ρωτήσω για την ετοιμότητα σε περιπτώσει καταστροφών. Έπρεπε να περιμένουμε περισσότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτόν τον τομέα. Εντάξει, κατόπιν εορτής μπορούμε να πούμε ότι ναι, θα έπρεπε να είχαμε κάνει περισσότερα. Αλλά βλέπουμε ότι υπήρχε ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης στην Ινδονησία, το οποίο χρησιμοποιήθηκε, χτύπησε κόκκινο, έδωσε σήμα, προειδοποίησε για επικείμενο τσουνάμι, οι υπολογισμοί όμως του συστήματος έπεσαν έξω. Υπήρχε λοιπόν έγκαιρη προειδοποίηση και μέσα σε μισή ώρα ή 45 λεπτά το τσουνάμι, ε, η κατάσταση αυτή επέστρεψε στο φυσιολογικό. Αυτή τη στιγμή διερευνούμε το ζήτημα. Όμως τα ευρήματα μέχρι τώρα δείχνουν ότι συνέβησαν πολλά ταυτόχρονα, πολλαπλές κρίσεις, ο σεισμός καταρχάς. Μετά, υποβρύχια δραστηριότητα, την οποία δεν μπόρεσε να αναλύσει το σύστημα που χρησιμοποιούταν. Και μετά αυτή η ρευστοποίηση του εδάφους, όπως σας είπα πριν, όπου η λάσπη κατάπια μέσα σε λίγα λεπτά ολόκληρα χωριά. Οι εικόνες είναι τρομακτικές αν τις δείτε. Σίγουρα θα μπορούσαν να είχαν γίνει περισσότερα. Εμείς στηρίζαμε την κυβέρνηση της Ινδονησίας μέχρι το 2013. Τώρα ο Ερυθρός Σταυρός έχει αναλάβει τις περισσότερες επιχειρήσεις επιτόπου. Δεν μπορούμε βέβαια να παραγνωρίζουμε το έργο του, αλλά αυτή τη στιγμή είναι πολύ νωρίς για να πούμε με ακρίβεια τι έχει συμβεί. Δεν ξέρουμε αν το μέγεθος είναι το ίδιο με την καταστροφή στην Ιαπωνία μετά το σεισμό, αλλά βλέπουμε ότι ακόμα εξελίσσεται η κατάσταση. Στις 5 και 2 το απόγευμα έγινε ο σεισμός. Υπήρξε η έγκαιρη προειδοποίηση για επικείμενο τσουνάμι. Και 20 λεπτά αργότερα το σύστημα θεώρησε πως ε, δεν θα υπάρξει τσουνάμι, οπότε επανήλθε από κόκκινο στο φυσιολογικό. Γι' αυτό και δεν ε, απεφεύχθη η τραγωδία. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Φυσικά θα μας κρατήσετε ενήμερους για τις εξελίξεις και έχετε δίκιο πώς πρέπει να εστιάσουμε στην αντιμετώπιση των καταστροφών. Και θα περιμένουμε τα ακριβή στοιχεία. Ευχαριστούμε πολύ, Ανδρούλα, που ξαναήρθατε παρά το γεγονός ότι σας καλέσαμε τελευταία στιγμή. Σας ευχαριστώ. Συνάδελφοι, μπορούμε να προχωρήσουμε στο σημείο 10, θέσπιση του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης. Είναι μια γνωμοδότηση της Επιτροπής μας, την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, ΛΥΜΠΕ. Είναι ένα νέο ταμείο που θα θεσπιστεί και θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο ταμείο ως ε, κομμάτι του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027. Προτείνεται μεγάλη αύξηση του ταμείου, 2,6 φορές μεγαλύτερη χρηματοδότηση. 10,4 δις ευρώ έχουν προταθεί. Το σκεπτικό πίσω από αυτό είναι να στηριχθούν τα κράτη-μέλη για την διενέργεια ελέγχων στα σύνορα. Η Επιτροπή Ανάπτυξης εστιάζει στις επιστροφές. Όμως, η Ellis Line, η συγγήτρια, μπορεί να μας πει περισσότερα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, προτείνεται η θέσπιση του Ταμείου Σύλλου και Μετανάστευση, το οποίο θα βοηθά τις διαδικασίες με 10,4 δισεκατομμύρια ευρώ κονδύλιο. Είναι μια σημαντική αύξηση σε σχέση με την περίοδο 2014-2020 όταν το Ταμείο είχε κονδυλέψει 6,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Καλωσορίζουμε λοιπόν αυτήν την αλλαγή, εφόσον αυτή η αλλαγή στοχεύει στην δημιουργία ενό καλύτερου και πιο αποτελεσματικού συστήματο ασύλου και μετανάστευση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματο Ασύλου. Η πρόταση αυτή θα επιτρέψει στι τρίτε χώρε να συνδεθούν με το Ταμείο αυτό, θα ενισχύσει τι δραστηριότητε Ευρωπαϊκή Ένωση εξωτερικά. Είναι επομένω αναγκαίο για την Επιτροπή Ανάπτυξη να θέσει ξεκάθαρες ασφαλιστικές ε, δικλίδες και να διασφαλίσει πώς οι δραστηριότητες θα αναφέρονται ρητά. Το άρθρο 5 της πρότασης της Επιτροπής δεν αναφέρει συγκεκριμένα τα είδη συνεργασίας που θα επιτρέπονται στο πλαίσιο του Ταμείου αυτού και δεν ε, αναφέρεται λοιπόν και ο πιθανός αντίκτυπος στις τρίτες χώρες. Η συνεργασία με τι τρίτε χώρε στο υφιστάμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο περιορίζεται στι εσωτερικέ υποθέσει και συγκεκριμένα στην νόμιμη μετανάστευση, τι ε, επιστροφέ και την επανεισδοχή. Πρέπει να αποφύγουμε από σταθεροποίηση των τρίτων χωρών, χρησιμοποιώντας αυτή την πολύ στενόμυαλη προσέγγιση και δίνοντα προτεραιότητα στην διαχείριση της μετανάστευσης. Η συνεργασία με τις τρίτες χώρες θα πρέπει να βασίζεται σε μια μηβαία προσέγγιση και όχι σε μονόπλευρη πρόσπιση των συμφερόντων της Ένωσης και της ασφάλειας των συνόρων. Η πρόταση δίνει υπερβολική έμφαση στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην πρόθεσή της να αυξηθούν οι επιστροφές και πανεσδοχές. Τα κριτήρια που έχουν προταθεί για την χρηματοδότηση σε εθνικά προγράμματα έχουν να κάνουν ως εξής. Το 40% της χρηματοδότησης, ανάλογα με τους ε, δείκτες, ε, θα διατίθεται στις επιστροφές ε, παράτυπων μεταναστών. Αυτό θα έχει καταστροφικές συνέπειες σε θέματα ασύλου, νόμης, μετανάστευσης και ενσωμάτωσης και θα δημιουργήσει κίνητρα σε κράτη-μέλη για να εφαρμόσουν αποφάσεις επιστροφής χωρίς να λάβουν υπόψη τους κινδύνους για όσους επιστρέφουν και ε, για τις χώρες προέλευσης. Προτείνουμε λοιπόν να εξισορροπηθεί η χρηματοδότηση. Πώς? έτσι ώστε να διοχετεύεται ως επιτοπλίστων στην διαχείριση του ασύλου και του συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη μετανάστευση μέσω νομίμων οδών. Ίσως το σχέδιο γνωμοδότησης θα έχετε διαβάσει ότι προτείνουμε να διατεθεί 40% για το άσυλο, 40% για την νόμιμη μετανάστευση και την ένταξη και 20% στην αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και στις επιστροφές. Θέλουμε να δώσουμε έμφαση στην ανάπτυξη έτσι ώστε οι επιστροφές να μην είναι μόνο αποτελεσματικές και, ένα, και με διάρκεια, αλλά και βιώσιμες τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και τις χώρες προέλευσης. Χρειάζεται μία εκτίμηση της και εξελόγηση της κατάστασης και της ικανότητας απορρόφησης σε τοπικό επίπεδο. Επίσης, να ε, αναλυθεί ο αντίκτυπος στις ε, τρίτες χώρες και να εξεταστούν τρόποι αντιμετώπισης της ε, ευάλωτης αυτής κατάστασης στην οποία θα περιέλθουν. Θα πρέπει να δημοσιοποιούνται τα στοιχεία επιστροφών έτσι ώστε να υπόκειται σε πλήρη έλεγχο από το Κοινοβούλιο και την κοινωνία των πολιτών και τις οργανώσεις της. Προσβλέπω στη συνεργασία με όλους τους και ηγητές και τους συναδέλφους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ελή, ξεκάθαρα ήταν. Και ως ομιλητές μέχρι τώρα έχω τη μοίρια. Όχι. Ο κ. Χολβένη πρώτα από το ΕΛΚ. Ναι, με τιμά που είμαι πρώτος. Μόνο σήμερα το απόγευμα είχαμε την ευκαιρία να το κοιτάξουμε, οπότε στο προκαταβολικά, συγγνώμη αν κάνω κάποια λάθη, αλλά με ενδιαφέρει πραγματικά πολύ το σχέδιο κειμένου της Έλλη. Και οι επικρίσεις δεν αφορούν το άτομό σου, αλλά το περιεχόμενο και θα γυρίσω στη μητρική μου γλωσσά. Ουγγρικά θα μιλήσω λοιπόν. Θα ήθελα λοιπόν να πω τα εξή. Εδώ έχουμε ένα φιλοσοφικό ζήτημα. Σε τι επικεντρωνόμαστε τον Ιούλιο το Συμβούλιο αποφάσισε την ενίσχυση δράσεων στο τοπικό επίπεδο. Αυτή ήταν η απόφαση του Συμβουλίου. Και οι τροπολογίες στα σημεία 3 και 9 νομίζω ότι κάνουν πιο αδύναμη την πρόταση της Κομισιόν. Καταλαβαίνω ότι θα μπορούσαμε να αλλάξουμε τα ποσοστά και καταλαβαίνω τους λόγους για τους οποίους γίνεται αυτό. Υπάρχει όμως κάτι το σημαντικό. Η παράνομη μετανάστευση θα πρέπει να εξαλειφθεί και θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες για αυτό το στόχο, για να το πετύχουμε. Επαναειστοχές. Αυτό δεν είναι στην ευρωπαϊκή κουλτούρα. Θεωρείται ως κάτι βίο, κάτι ομό, κάτι απαράδεκτο κάτι το οποίο είναι αδιανόητο. Ναι, το παραδέχομαι ότι δεν είναι εύκολο να το φανταστεί κανείς αυτό. Γι' αυτό ακριβώς θεωρώ το 3 ότι είναι προβληματικό το σημείο. Γιατί όχι μόνο εμποδίζει τις προσπάθειες που γίνονται, αλλά στην πράξη για αυτά τα άτομα καθίσταται αδύνατο να γίνουν οι και νομίζω ότι δεν είναι προσυμφέρον Και υπάρχει και άλλη μια παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω, κάπως προσωπική αυτή. Πήγα στην Αφρική, πήγα στη Μέση Ανατολή. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τους ντόπιου πληθυσμού, αυτούς που φεύγουν από τις χώρες τους, τι κινήτρα έχουν. Νομίζω ότι είμαστε ανεύθυνοι αν εμείς ενθαρρύνουμε τον κόσμο να φύγει από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Θεωρώ ότι με το σχέδιο αυτό του κειμένου, με τρόπο ανεύθυνο, τους ενθαρρύνουμε να φύγουν από τα σπίτια τους και στην ουσία να καταστήσουν αδύνατη την επιστροφή τους. Τελευταία παρατήρηση. Η διεθνής κοινότητα είναι υπεύθυνη για τα άτομα τα οποία είναι εκτοπισμένα με τη βία ή εθελοντικά και νομίζω ότι είναι τελικά προς το συμφέρον όλων να προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε αυτά τα άτομα όσο πιο κοντά γίνεται στο σπίτι τους. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να τονιστεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Ελένη Θεοχάρους, παρακαλώ. Ελένη. Πρόεδρε, για να είμαι ειλικρινής, τώρα είδα το κείμενο. Έχω κάποιες παρατηρήσεις να κάνω ε, και ε, νομίζω αρκετά ε, ε, αρκετές τροπολογίες. Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία ε, για μας είναι η επιστροφή των ετούντων πολιτικού άσυλο στις χώρες που θα τους δεχθούν πίσω να είναι sustainable, να είναι βιώσιμη, να μην είναι και πάλι εκτεθειμένοι σε κινδύνους ε, που δεν θα τους επιτρέπουν να παραμείνουν εκεί ή που θα τους οδηγήσουν και πάλι στην ε, παράνομη ε, μετανάστευση. Οπωσδήποτε είναι δύσκολο να στέλνουμε τον καθένα στην χώρα από την οποία προέρχεται ε, και οι συμφωνίες επανεισδοχής νομίζω ότι θα είναι μια κατευθυντήρια γραμμή για αυτό το ζήτημα. Άρα θα πρέπει να δούμε ξανά όλες τις συμφωνίες επανεισδοχής που έχουν υπογραφεί. Αυτά για την ώρα και θα τα ξαναπούμε. Thank you um, Πρόεδρος, ε, ευχαριστώ πολύ. Μία βρήκε από τους φιλελευθέρους. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για την εισήγηση. Νομίζω ότι είναι σωστό που έχουμε την εισήγηση αυτή για το Ταμείο Προσφύγων και Μετανάστευσης και πολύ σωστά το Ταμείο καλύπτει τις δαπάνες αυτές για την κοινή πολιτική μετανάστευσης και μεταναστευτικού και προσφυγικού. Πρέπει να υπάρχουν ορισμένε προϋποθέσεις για την εφαρμογή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Και αν υπάρχουν δράσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να μπαίνουν όρια σε αυτές. Και αυτές να υπακούν στους γενικότερους στόχους του Ταμείου. Να μην υπάρχει επικάλυψη με άλλες δράσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από άλλα ταμεία. Η δε Έλλης τα έχει λάβει αυτά υπόψη. Στην τροπολογία της μόνο 6 για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. υποστηρίζει την εθελοντική επιστροφή και το κείμενο τη Κομισιόν. Και εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικό να υποστηριχτούν αυτές. Όμως, στο Ταμείο θα πρέπει να μπει και ένα στοιχείο ευελιξίας, ώστε να μπορούμε να αναπτύξουμε αυτό το θεσμό των ε, εθελοντικών επιστροφών. Εάν ένα πρόσωπο έχει λάβει μια αρνητική απόφαση, το έχει δηλαδή κοινοποιηθεί μια αρνητική απόφαση, θα πρέπει το Ταμείο να καλύπτει την επιστροφή και βέβαια και σε περιπτώσεις όπου δεν είναι θελοντική η επιστροφή αλλά συνεπάγεται κόστος. Το Ταμείο χρηματοδοτεί λοιπόν τις επιστροφές αυτές Στην πράξη όμως πρέπει να στοχεύει στην πρώτη φάση της ένταξης δηλαδή των μεταναστών. Ε, πάντως εγώ θα υποστηρίξω την πρόταση της Ellis Line που μιλεί για το μερίδιο του 44% να μπει για θέματα επιστροφής Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Κιένγκε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την Έλλη και για αυτή την πρόταση. Το ταμείο αυτό είναι πολύ σημαντικό για να προσεγγίσουμε το θέμα της μετανάστευσης όχι ως κάτι το οποίο μόνο, αλλά ως κάτι το οποίο θα πρέπει να το μισθεί με μέσω μακροπρόθεσμες λύσεις. Και αυτό θα εξαρτηθεί από τον τρόπο με τον οποίο εμεί θα προσφέρουμε λύσει με το Ταμείο αυτό. Καταρχά έχουμε το θέμα σεβασμού του δικαιώματος ασύλου και γι' αυτό θα πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά την ε, αρχή της μη επαναεισδοχής, να δούμε τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις πολιτικές μετανάστευση και ασύλου της Ένωσης για την επανασδοχή. Εγώ επιμένω πολύ στο θέμα της αξιοπρέπειας των ατόμων. Αν θα πρέπει να επιστρέψουν αυτά τα άτομα, θα πρέπει να είναι σεβαστή η αξιοπρέπειά τους. Και ένα άλλο σημείο που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ως πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτό που αφορά την ε, νόμιμη μετανάστευση και την εσωμάτωση. Αυτό είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που κατά την άποψή μου πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση μέσω και τοπικών πολιτικών να πετύχουμε την ενσωμάτωση και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας σε όλη την επικράτεια και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επικράτεια. Οπότε θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αποκλείσουμε ή να εξαιρέσουμε θεσμούς και κυβερνήσεις που δεν θέλουν να προωθήσουν πολιτικές ενσωμάτωσης. Τα πιο σημαντικά είναι αυτά. Αλλά το κυριότερο θα έλεγα είναι ακριβώς η ενσωμάτωση και τα νόμιμα μέσα για την επίτευξη της. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει η πρόεδρος Μακάβαν. Δεν βλέπω άλλα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που να ζητεί το λόγο. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Καζεύσκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών. Ε, μπορείτε να κλείσετε το μικρόφωνο σας, ε, κυρία Θεοχάρους. Ευχαριστούμε. Ε, DG Home, λοιπόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για όλες ε, τις τοποθετήσεις των αξιοτήμων μελών σας και για το ενδιαφέρον που δείχνετε στις προτάσεις που κάναμε τον Ιούνιο. Πράγματι, υπάρχει ανάγκη σημαντικών συνεργειών συμπληρωματικοτήτων και συνοχής μεταξύ του παρόντος μηχανισμού που κατευθύνεται κυρίως στις χώρες μέλη και των χρηματοδοτικών μηχανισμών που στοχεύουν σε στόχους περισσότερο ανάπτυξης. Έχουμε προβλέψει μια εξωτερική διάσταση του Ταμείου και στα τρία σκέλη στόχων για το άσυλο, προστασία για νομική, συγγνώμη, για ένομη μετανάστευση, ένταξη και για επανεισδοχή. Εκεί υπάρχουν παντού πτυχές εξωτερικής πολιτικής και περιλαμβάνονται, μάλλον μεταφράζονται σε στόχους που καθορίζονται σαφώς στο τμήμα των στόχων, δηλαδή στο παράρτημα 2, όπου λέμε καθαρά ποια είναι η ανάγκη και η σκοπιμότητα συνεργασίας με τρίτες χώρες και προβλέπουμε εξ αρχής τις ανάγκες αυτές και τις σαφείς προτεραιότητες. Τώρα το πώς θα γίνει. Υπάρχουν τρόποι, modalities, για την καθιέρωση της συνεργασίας σε μια βάση επιτούτο, ad hoc, emergency assistance ας πούμε και βέβαια και πιο μακροπρόθεσμη δράση συνεργασίας. Θέλω να τονίσω λοιπόν ότι οι μηχανισμοί αυτοί είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, τονίζουμε τη σημασία των συμφερόντων των χωρών μελών για τη συνεργασία τους, για να δουν οι δράσεις τους να υποστηρίζονται από το Ταμείο. Έχουμε προβλέψει και μια thematic facility, που νομίζουμε ότι είναι καλός μηχανισμός για την κατανομή σταδιακά των πόρων. Αυτό θα εξαρτηθεί από τις προτεραιότητες, ανάγκες και κατάσταση. Θέλουμε δηλαδή, έχουμε προτείνει ποσοστά κατανομών για άσυλο, νόμιμη μετανάστευση, επανα, επανεισδοχή, ποσοστά τα οποία θα κατανεμούνται στις χώρες μέλη. Όμως, θέλω να σας επισημάνω τον ε, σημαντικό μηχανισμό ευελιξίας της Thematic Facility. Μπορούμε ε, να διαθέτουμε υψηλότερα ή χαμηλότερα κονδύλια ανάλογα με τις προτεραιότητες κατά τη διάρκεια της ε, διαχείρισης εφαρμογής του Ταμείου μέχρι το 2027. Ο μηχανισμός θα επιτρέπει λοιπόν ευελιξία και προσαρμογή και από την πολιτική σκοπιά. Είναι βέβαια σημαντικό να δοθούν προτεραιότητες σε διεθνή προγράμματα και σε ένα πρόγραμμα εργασίας της Thematic Facility Θέλω όμως να τονίσω και την πτυχή διακυβέρνησης, διαδικασία διακυβέρνησης για να επιτύχουμε συνέργειες στα πλαίσια των δράσεών μας. Δηλαδή εδώ υπάρχει διπηρεσιακή συνεργασία για να έχουμε τις αναγκαίες πληροφορίες, για να κατευθύνουμε τη διαδικασία σταδιακά. Θα χρειαστούμε αντιπροσωπείες. Αυτό που είναι σημαντικό όμως, θα χρειαστούμε μάλλον α, αναθέσεις εντολών να δούμε τα δεδομένα και να δούμε και τα αποτελέσματα των δράσεων που υποστηρίζει χρηματοδοτικά το Ταμείο μας. Σας ευχαριστώ. Η Έλλη Σλάιν τώρα πάλι. Επιθυμώ να ευχαριστήσω όλους και όλους για τα σχόλιά τους. Είμαι βεβαία ότι θα έχουμε χρόνο τις επόμενες εβδομάδες να τα συζητήσουμε. Λυπούμε που καθυστέρησε κάπως. Υπήρχε ένα τεχνικό πρόβλημα. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα λάβαμε τη γνωμοδότηση και αντιλαμβάνεστε αυτή έπρεπε και να αναθεωρηθεί και από κάποιες υπηρεσίες ή να επανεξεταστεί. Τις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε χρόνο να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες. Ήθελα ιδιαιτέρως να διαβεβαιώσω τον συνάδελφό μου Τζόρτζ για το γεγονός ότι ο παρόν κανονισμός δεν έχει επίπτωση στις, στην, στο θέμα της επανεισδοχής ή των επιστροφών γενικότερα. Πρόκειται για νέο ταμείο το οποίο πριν στόχευε την μετανάστευση και άσυλο και τώρα κατά κάποιο τρόπο διευρύνεται ώστε να περιλάβει και την εξωτερική διάσταση επομένω και τις επιστροφές. Δεν το αμφισβητούμε καν στη γνωμοδότησή μας. Αυτό που κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε από τη σκοπιά τη ανάπτυξη εφόσον πρόκειται μόνο για γνωμοδότηση και αυτή θα συζητηθεί στην Επιτροπή Θεμελιωδών Ελευθεριών. Να, ληφθεί ιδιαίτερα, ε, να ληφθεί υπόψη μάλλον η ιδιαίτερη κατάσταση των αναπτυσσόμενων χωρών όταν θα λαμβάνονται αποφάσεις για επιστροφές και θα χρησιμοποιείται αυτό ο διαθέσιμο τώρα πλέον χρηματοδοτικός μηχανισμό Θεωρείται ίσως είστε ίσως κάπως υπεραισιόδοξος όταν θεωρείτε ότι οι μετανάστες θα διαβάσουν πρώτα τον κανονισμό του MFF για να δουν αν αξίζει τον κόπο να φύγουν στις πατρίδες τους ή όχι. Είμαι βέβαιος ότι έχουν άλλους λόγους για να αποφασίσουν τελικώς να εγκαταλείψουν τις χώρες τους και όχι το πώς θα κάνουμε εμείς την κατανομή των κονδυλίων μεταξύ ασύλου, νόμιμης μετανάστευσης και επιστροφών. Δεν ακολουθώ δηλαδή καμιά ιδιαίτερη ιδεολογική προσέγγιση για την σύνταξη των τροπολογιών μου. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι η πτυχή της ανάπτυξης να λαμβάνεται υπόψη στη χρηματοδότηση του Ταμείου. Συμφωνώ απολύτως με την Ελένη σε ό,τι αφορά την ανάγκη διατήρησης της βιωσιμότητας. Θα τα δείτε αυτά και στις τροπολογίες μου. Και βεβαίως και με το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων που θύμισε ο συνάδελφος του Άλτε και η Σεσίλ Κιένγκε. Και τι άλλο, τώρα δεν βλέπω τίποτα άλλο μια στιγμή ε, διαβάζω τα, τις σημειώσεις που έχω κάνει για τα σχόλιά σας. Ναι, θα συζητήσουμε επίσης και τα ποσοστά. Έχουμε εμπειρία και δει την εμπειρία ότι όταν μπαίνουν στο ίδιο καλάθι, χρηματοδοτικό καλάθι, διάφορες προτεραιότητες, πρέπει να εξισορροπηθούν. Πρέπει δηλαδή να φροντίσουμε να μην δημιουργήσουμε λάθος κίνητρα προς μια κατεύθυνση που μπορεί να επιφέρει ζημία σε άλλες προτεραιότητες. Χρειάζεται να διασφαλίσουμε ότι οι χώρες μέλη θα μπορούν να εργάζονται αποτελεσματικά για το σύστημα ασύλου μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργώντας νόμιμες εναλλακτικέ επιλογές. Αν θέλουμε να δούμε και νόμιμη μετανάστευση δηλαδή. Να εξισορροπήσουμε λοιπόν τις χρηματοδοτήσεις αυτές των χωρών μελών, αλλά και προς τα έξω με τρίτες χώρε. Και όλοι όσοι ασχολούνται με τον τομέα και ιδίω εκείνοι που ασχολούνται με τις εθελοντικές επιστροφές μας είπαν ότι είναι θεμελιώδε να λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση επιτόπου και η ικανότητα απορρόφησης. Δεν θέλουμε δηλαδή να επιστραφούν κάποιοι και μετά να προσπαθήσουν ξανά με επικίνδυνο τρόπο να επανέλθουν εδώ σε μας. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και αναμένουμε ενδιαφέρον πραγματικά τη συνεργασία μαζί σας. Το τελευταίο σχόλιο που θα κάνω είναι ότι επειδή έχουμε βάλει σε ένα μηχανισμό διαφορετικούς στόχους, αγαπητή Λίντα, τα έχουμε επιτώσει πολλές φορές, πόσο δύσκολο είναι για μας να διασφαλίσουμε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο του Ευρωκοινοβουλίου, διότι είμαστε σε μια κατάσταση οριακή, δηλαδή είμαστε πάνω στα όρια με άλλα, με ε, ταμεία. Και με το καταπιστευματικό ταμείο για την Αφρική. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε μια βεβαιότητα, να μην υπάρχει αμφισημία και να διασφαλίσουμε ότι οι στόχοι και τα πράγματα που θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το νέο ταμείο είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα διατυπωμένα μέσα στο κείμενο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Λίντα Μακάβανα. Ευχαριστώ πολύ. Όπως είπες, έχει, υπάρχει χρόνος να τα συζητήσουμε. Έχουμε δηλαδή μέχρι τις 29 Δεκάτου το μεσημέρι για την κατάθεση τροπολογιών και η ψηφοφορία θα γίνει στις 3.12 του. Άρα δεν χρειάζεται μεγάλη βιασύνη, υπάρχει χρόνος. Ευχαριστώ λοιπόν και πάλι την αγαπητή Έλλη και τους υπολείπους και την εκπροσώπηση της DigiHome. Να έρθουμε τώρα στο υπαριθμό 11. Το πρόγραμμα δηλαδή του ε, εθελοντικού σώματος της Ένωσης άλλο ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο θα ενταχθεί στο νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Εκεί εμείς συντάσσουμε γνωμοδότηση ε, για την αρμόδια της ουσίας Επιτροπή Πολιτισμού. Όμως εμείς έχουμε αποκλειστική αρμοδιότητα για το θέμα του προγράμματος Solidarity Core. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να συγχωνεύσει τα προγράμματα και να συγχωνεύσουν επομένως το εθελοντικό ε, σώμα των, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με άλλο πρόγραμμα το European Solidarity Corps που είναι πρόγραμμα για τους νέους και εγκρίθηκε φέτος το καλοκαίρι από ορισμένες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Εδώ λοιπόν εμείς είμαστε συναρμόδιοι με την ε, Επιτροπή Πολιτισμού. Έχουμε παρουσία στην Επιτροπή μας σήμερα της ενδιάμεσης αξιολόγησης της σχετικής πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και νομίζω η ιδέα είναι να ακούσουμε πρώτα την παρουσίαση της Midterm Evaluation πριν να αρχίσουμε την συζήτηση και την πρόταση πριν να κάνουμε τη συζήτηση. Να ακούσουμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενδιάμεση πανεξέταση και μετά θα δούμε γιατί γίνεται η προσπάθεια συγχώνευσης. Χαίρομαι πάντως διότι έχουμε την κυρία Μικέλε Μισελ Σόιντροβα από την ε, Συναρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Ε, να αρχίσουμε τότε λοιπόν. Ακούγοντας την εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης ΕΚΟ της ε, Κομισιόν, η οποία θα παρουσιάσει την αξιολόγηση της νέας προτάσεως. DG Education and Culture. Θα μας εξηγήσετε σίγουρα ποιος ε, λαμβάνει το λόγο, θα μας συστηθείτε. Ε, δεν έχω το όνομά σας. Ευχαριστώ πολύ. Έμπα Μούσαρ από την Γενική Διεύθυνση Εκονομάζομαι. Είμαι υπεύθυνη για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Η Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ διαχειρίζεται την ε, πρωτοβουλία εθελοντών τη Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και την αξιολόγηση του προγράμματο. Συγγνώμη, λέει η Συζητάμε χωρί το σχέδιο γνωμοδότηση. Είναι πρώτη συζήτηση μόνο για να συλλέξουμε πληροφορίε. Θα πρέπει να το πω στην αρχή. Συγγνώμη που σα διάκοψα. Συνεχίστε. Θα κάνω λοιπόν μία σύνοψη, ακριβώς διότι δεν έχετε χρόνο. Και φυσικά υπάρχουν πολλέ λεπτομέρειε. Καλό θα ήταν να είχαμε μια ολόκληρη ώρα στη διάθεσή μα για λεπτομερή παρουσίαση. Η αξιολόγηση λοιπόν βρήκε ότι είναι πολύ σημαντική για τα κράτη-μέλη, όμως η, η πρωτοβουλία αυτή, η εφαρμογή της κυλοποίησή της όμως ε, έχει ελλείψει στην αποτελεσματικότητα ακριβώς διότι η πρωτοβουλία αυτή δεν χρησιμοποιείται αρκετά από τις διάφορες μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Παρέχεται κάθε χρόνο χρηματοδότηση στα, στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις για να χρησιμοποιήσουν εθελοντές. Πολύ χαμηλά λοιπόν τα επίπεδα της ανάληψης πρωτοβουλίας της χρήσης. Τώρα έχουμε φτάσει στον βασικό κανονισμό σε κατά εξουσιοδότηση και εκτελεστικό κανονισμό, οι οποίοι θα αναφέρονται με πολλές λεπτομέρειες ε, στις ε, επιμέρους διατάξεις. Λοιπόν, το 2005 πρώτο χρησιμοποιήθηκε, θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε 350 εθελοντές, καταλήξαμε στο τέλος να χρησιμοποιήσουμε μόνο 44, Στην επόμενη χρονιά από 350 τα λήξαμε να χρησιμοποιούμε τους 160. Το 2017 θέλαμε να ανεβάσουμε τα νούμερα αυτά γιατί η πρωτοβουλία είχε καθιερωθεί πλέον. Θέλαμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε πάνω από 500 εθελοντές και καταφέραμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο 175. Φέτος μειώσαμε το στόχο, ζητήσαμε λιγότερα για να χρησιμοποιήσουμε μόνο 367 εθελοντές. Τώρα όμως τα στοιχεία αυτά αφορούν την περίοδο 2005 μέχρι το πρώτο μισό του 2017 και όπως καταλαβαίνετε η βάση δεν είναι αρκετά μεγάλη. Αυτή η σύγκριση λοιπόν αποτελεσματικότητας δεν ήταν ικανοποιητική. Βρήκαμε επιπλέον ότι ο σχεδιασμός του προγράμματος είναι αρκετά περίπλοκος και τα πρότυπα για την ε, διαχείριση των εθελοντών είναι δύσκολα. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις πρέπει να περάσουν μία αρκετά δύσκολη διαδικασία, γραφειοκρατική επίπονη, μέχρι να φτάσουν σε σημείο να μπορούν να χρησιμοποιήσουν εθελοντές. Ο εκτελεστικός κανονισμός, για παράδειγμα, αναφέρει πως οι θέσεις πρέπει να δημοσιεύονται τέσσερις εβδομάδες νωρίτερα, Ύστερα πρέπει να διοργανώνεται κατάρτιση που θα διαρκεί δύο εβδομάδες προτού φτάσουν στο σημείο να να εφαρμόσουν και να χρησιμοποιήσουν το σύστημα. Είναι λοιπόν δύσκολη διαδικασία, περίπλοκη, χρονοβόρα. Αναλύσαμε επίσης θέματα εφαρμογής, άλλη γενική διεύθυνση, DGEAC. Εκεί είχαμε καλύτερα αποτελέσματα, όμως πρέπει να μειωθούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια, σχετικά με την διαχείριση των εθελοντών που επιβαρύνουν και το επιτόπιο προσωπικό. Μετά, ένα ακόμα έβριμα ήταν ότι το πρόγραμμα αυτό δεν είναι αρκετά γνωστό. Χρειάζεται λοιπόν να εντείνουμε τις προσπάθειες για ενημέρωση. Σε γενικές γραμμές, η ένταξη στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης μπορεί να βοηθήσει για να αντιμετωπιστούν ορισμένες από αυτές τις ελλείψεις. Είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα και μπορούμε να εποφεληθούμε από αυτό. Χρειάζεται βέβαια να γίνει πρόθεση, να χρησιμοποιήσουμε την Ευρωπαϊκή Θελοντική Υπηρεσία που προϋπήρχε έτσι ώστε το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης να πάει ακόμα παραπέρα. Επίσης, τι άλλο είδαμε, ότι υπάρχει σύγχυση. Οι Ευρωπαίοι εθελοντές δεν ξέρουν πού να απευθυνθούν, πού να δηλώσουν εθελοντική συμμετοχή. Υπάρχει επίσης και πρόβλημα στην διαδικασία αίτησης, γι' αυτό λοιπόν προτείνουμε τη δημιουργία μιας μονοαπευθυντικής θηρίδας όπου θα μπορούν να προσφεύγουν οι εθελοντές και επίσης τη συγχώνευση κάποιων υπηρεσιών όπως για παράδειγμα κατάρτιση, ασφάλιση, πρόθεση, πληροφορική έτσι ώστε να εξοικονομήσουμε πόρους. Αυτά ως προς την ενδιάμεση αξιολόγηση. Θα χαρώ πολύ να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ωραία. Θα ακούσουμε την παρουσίαση και του νέου μέσου από την Γενική Διεύθυνση Καλ... Καλύτερα να τα ακούσουμε και τα δύο και μετά να περάσουμε σε ερωτήσεις από τους ευρωβουλευτές. Η αξιολόγηση δεν είναι αρκετά θετική. δεν κατάφερε το project αυτό να προσελκύσει μη κυβερνητικέ οργανώσεις... να προσελκύσει εθελοντέ. Ίσως λοιπόν θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεδομένης της εμπειρίας και των μη θετικών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, να μας πει τι μπορεί να γίνει για να αλλάξει, πώς μπορεί να τροποποιηθεί για να βελτιωθεί το πρόγραμμα. Να δούμε ποιος είναι ο στόχος του προγράμματος, έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μια νέα πρόταση. Κύριε Φράντσα από εκεί διεύθυνση εκπαίδευσης και πολιτισμού. Όπως είπατε, με τη νέα πρόταση προσπαθούμε να λάβουμε υπόψη μας όλες τις συστάσεις από την ενδιέμεση εξολόγηση των προγραμμάτων εθελοντισμού. Παρουσιάσαμε την νομική βάση, η οποία είναι αρκετά απλή και επικεντρωθήκαμε σε δύο πτυχές. Καταρχάς, η ποιότητα των δραστηριοτήτων. Δεύτερον, η περιληπτικότητα και επί τη ευκαιρία στην υπηρεσία εθελοντισμού έχουμε την εμπειρία ότι ένας από τους τρεις συμμετέχοντες είναι νέοι με λιγότερες ευκαιρίες. Οπότε αυτό είναι και ένα μάθημα για την ανθρωπιστική βοήθεια. Όταν μιλάμε λοιπόν για ενσωμάτωση, μιλάμε για δύο βασικές ε, διαστάσεις. Αποτελεσματικότητα και αποτελέσματα. Αυτά πώς θα προσεγγίζουμε. Νομίζω ότι ένα από τα κέρδη της ενσωμάτωσης το ανέφερε η Κατρίνα. Δηλαδή, έχουμε μια κοινή ομπρέλα για όλα τα προγράμματα, έχουμε μια κοινή επωνυμία για λόγους επικοινωνίας, αλλά και διαφάνειας και ορατότητας και το τωρινό εθελοντικό σώμα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει γύρω στους 80.000 νέους που εξέφρασαν ενδιαφέρον εθελοντικά να συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες στην Ευρώπη και βεβαίω με την ολοκλήρωση του κεφαλαίου της ανθρωπιστικής βοήθειας το οποίο είναι συγκεκριμένο κεφάλαιο στην πρόταση τότε η ορατότητα θα διευρυνθεί και θα επεκταθεί δηλαδή και σε αυτό το κεφάλαιο της ανθρωπιστικής βοήθειας. Μπορούμε να βασιστούμε στους αποτελεσματικού μηχανισμούς εφαρμογής που ήταν επαδοσματική τα 25 χρόνια ζωής αυτής της υπηρεσίας και στις Βρυξέλλες και στις διάφορες χώρες. Έχουμε διάφορα εργαλεία με τα οποία είμαστε βέβαιοι ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε και εξοικονομήσεις. Είναι αυτονόητο ότι υπάρχουν κάποια χωριστά χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων ανθρωπιστικής βοήθειας και βεβαίως αυτά θα ληφθούν υπόψη δεόντως, παραδείγματο χάρη μέσω συγκεκριμένων μορφών εκπαίδευση των εθελοντικών, δηλαδή που θα είναι των εθελοντών που θα είναι δραστήριοι στην ανθρωπιστική βοήθεια. Και συνοψίζοντας, μάθαμε από τις συστάσεις των εμπειρογνωμόνων, προτείναμε ένα ενιαίο αποτελεσματικό κανονισμό που διασφαλίζει την ποιότητα, την περιληπτικότητα και όλες οι δραστηριότητες βρίσκονται εκεί ακριβώς. Δηλαδή βάσει αυτών των αρχών που είπαμε προηγουμένως, δηλαδή περιληπτικότητα, ο μικροσκοπικός χαρακτήρας κτλ. Αυτό από μένα και με εδώ να ακούσω σχόλια και προτάσεις σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Λέκη Πρόεδρος. Τώρα, να ρωτήσω την Ελένη Ελένη, να δώσω το λόγο πρώτα στην κυρία Σοτρόβα. Συμφωνείς? Κυρία Σοντρόβα, παρακαλώ. Πείτε μα την άποψη τη Επιτροπή Πολιτισμού. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για το λόγο και την πρόσκληση. Χαίρομαι που μπορώ να συμμετάσχω σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων με εσάς εκτιμώ αυτή την ε, ανθρωπιστική δραστηριότητα που είναι βέβαια αρμοδιότητα της δικής σας Επιτροπής και άκουσα με ενδιαφέρον την αποτίμηση του προγράμματος της Ένωσης βλέποντας βέβαια κάποια αδύναμα στοιχεία σε αυτά τα προγράμματα παροχής βοήθειας. Βλέπουμε λοιπόν αυτά τα προγράμματα να παρουσιάζουν και πλεονεκτήματα αλλά και ενδεχόμενου κινδύνου. Οπότε θα ήταν καλό να το γνωρίζουμε αυτό. Τα πλεονεκτήματα είναι η ορατότητα, η προσβασιμότητα, η αλληλεγγύη του σώματος αυτού που θα δώσει περισσότερη ορατότητα και ευκαιρίες στο σώμα δίνοντας ή μάλλον προκαλώντας, δημιουργώντας αυτό το one-stop shop και ένα σήμα Ευρωπαϊκού Θελοντικού Σώματος και ελπίζουμε να είναι εύκολο οι συμμετέχοντες οργανισμοί να προσφέρουν θέσεις και να βρουν τους κατάλληλους υποψηφίους και για τους υποψηφίους του ίδιου θα έπρεπε να είναι πιο εύκολο να βρουν περισσότερες ευκαιρίες μέσω ενός ενιαίου πόρταλ. Συμφωνώ με τους εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης και άλλους συναδέλφους ότι υπάρχει αυτό το μεγάλο πλεονέκτημα ενός κοινού ενιαίου προγράμματος. Αφετέρου υπάρχουν όμως και κάποια άλλα στοιχεία που θα πρέπει να δούμε, ας πούμε περιορισμός ε, ηλικιακός 30 χρονών και αυτό ισχύει και για την ανθρωπιστική βοήθεια. Προσωπικά είμαι υπέρ. Εξάλλου το εθελοντικό σώμα αφορά νέους ανθρώπους και η ηλικία, το όριο ηλικία θα πρέπει να αφορά όλες τις δραστηριότητες του σώματος αυτού. Επιπλέον, Σύμφωνα με πληροφορίες που έχω, το 14% των συμμετεχόντων στα προγράμματα ήταν άνω των 30. Ίσως οι εκπρόσωποι της ε, Κομισιόν να θέλουν να το σχολιάσουν αυτό. Οι άνω των 30 θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στις ανθρωπιστικές δραστηριότητες, όχι όμως στο πλαίσιο του εθελοντικού σώματος. Και από ό,τι καταλαβαίνω από κάποια προοπτική, από κάποια σκοπιά, οι ανθρωπιστικές δραστηριότητες λόγω του χαρακτήρα τους απαιτούν περισσότερη οριμότητα, επειδή ακριβώς αντιμετωπίζουν μεγαλύτερους κινδύνους. Και γι' αυτό ακριβώς θα ήθελα να σεβαστώ βέβαια την θέση τη δική σας και την γνωμοδότηση που υιοθετήσατε στην Επιτροπή σας. Ήδη έχω υποβάλει το σχέδιο έκθεσης και θα το συζητήσουμε εμείς την Τετάρτη. Προτείνω διάφορες οριζόντιε αλλαγές που θα έχουν αντίκτυπο και στην ανθρωπιστική βοήθεια. Καταρχάς αποφάσισα να επαναεισαγάγω κάποια σημεία τα οποία ήταν αντικείμενο συμφωνίας στον τριμερή διάλογο στον πρώτο του Εθελοντικού Σώματος, του Ευρωπαϊκού, και αυτό έχει να κάνει με κάποιου ορισμούς, καταρχάς. Κατά δεύτερο λόγο θα ήθελα να είπα να εισαγάγω μία ενδεικτική κατανομή των κοντιλίων ανάλογα με τι δραστηριότητε. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό ώστε να διασφαλίσουμε το ότι ο θελικός χαρακτήρας αποτελεί τον πυρήνα του προγράμματο. Και στον τριμερή διάλογο είχαμε μία έκκληση για τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να έχουμε μια ενδεικτική κατανομή ακριβώς των κονδυλίων σε σχέση με τις ε, δραστηριότητε αυτές. 19% στα εθελοντικά, 10% για την κατάρτιση και την εκπαίδευση και νομίζω ήταν καλό κλίδα κατανομή αυτό. Θα ήθελα να το τηρήσουμε αυτό, λαμβάνοντα ταυτόχρονα υπόψη και την ολοκλήρωση τη συμμετοχή της ευρωπαϊκής βοήθειας. Δηλαδή ενδεικτικά 86% θα αφορά τις ε, δράσεις εθελοντισμού και αλληλεγγύης και τα προγράμματα εθελοντισμού. 8% θα αφορά την απασχόληση και την εκπαίδευση, 6% ανθρωπιστική βοήθεια. Το ενδεικτικό αυτό 6% αντιπροσωπεύει περισσότερο από ό,τι, από έχουμε στον προπολογισμό της Ένωσης αυτή τη στιγμή. 147,9 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή και μας επιτρέπει να τηρήσουμε στόχους σε σχέση με τους συμμετέχοντες. Προτείνω επίσης και διάφορα μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ορατότητα του προγράμματος. Είναι φιλόδοξη η πρόταση της Κομισιόν, όπως ξέρετε 350 ευκαιρίες μαζί με την ανθρωπιστική βοήθεια, οπότε θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει επαρκές ενδιαφέρον και, στους, και μεταξύ των συμμετεχόντων και μεταξύ των εθελοντών. Γι' αυτό ακριβώς προτείνω οι συμμετέχοντες να έχουν τη δυνατότητα να γίνουν πρεσβευτές του προγράμματος. Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να προωθείται δυναμικά σε επικοινωνικό επίπεδο, μέσω κοινωνικών δικτύων κτλ. Να φτάσει σε αποβακρισμένες περιοχές και το διοικητικό βάρος σε σχέση με την ε, κατανομή επίσης θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί ιδιαίτερα για τις ε, και Αυτό θα πρέπει να το δούμε και ένα έδρας δραστηριότητα. Δηλαδή, τα προπετούμενα αναδραστηριότητα ποικίλουν άλλο στην ανθρωπιστική, άλλο σε άλλε δραστηριότητε και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μα. Και εκτό από αυτό, προτείνω διάφορε άλλε αλλαγέ, οι οποίε δεν έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ανθρωπιστική βοήθεια, όμω θα μπορούσαν να βελτιώσουν τις προϋποθέσεις ή τις συνθήκες Παραδείγματο χάρη να τονίσω την ενσωμάτωση, το στόχο της ενσωμάτωσης, ώστε να έχουμε περισσότερη προσβασιμότητα για άτομα που έχουν λιγότερες ευκαιρίες. Επίσης, διευκρίνησα τον ορισμό του εθελοντή και επανεσήγαγα τον ορισμό της αλληλέγγυας δραστηριότητα. Στις 10 Οκτώβρη, λοιπόν, θα τα παρουσιάσω όλα αυτά, λοιπόν, και είστε πρόσδεκτοι να παραστείτε κατά διάρκεια της συζήτησης και ελπίζω να έχουμε μια καλή συνεργασία με την εισηγήτρια της ε, γνωμοδότησης. Και προσβλέπω στις περαιτέρω συζητήσεις μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, Ελένη, Thank you, Chair. Despite... Κυρία Θεοχάρους, παρά το γεγονός ότι το νομικό πλαίσιο και το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού για το πρόγραμμα του European Solidarity Corps ξεκινούν από την πρόταση της πρώην Επιτρόπου Γεωργίευα που ήταν, είχε το χαρτοφυλάκιο της ανθρωπιστικής βοήθειας στην πρόταση που είχε κάνει τότε για τη δημιουργία μιας ανθρωπιστικής ε, δύναμης ειδικών καθηκόντων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Παρ' όλα αυτά λοιπόν ε, σήμερα ε, στοχεύουμε σε ένα άλλο πράγμα και για το λόγο αυτό να μου επιτρέψετε να έρθω σε ορισμένα θέματα και να θέσω κάποιες ερωτήσεις που έχω τώρα. Όσον αφορά το σκέλος ε, του Ευρωπαϊκού Ανθρωπιστικού Εθελοντισμού, μέχρι το τέλος του 2018 αναπτύχθηκαν μόνο 206 εθελοντέ σε 28 χώρε μέλη. Από το 2015. Χαμηλό αριθμό. Με την συμπερίληψη αυτού του σκέλους στο European Solidarity Core μπορούν να αναπτυχθούν συνέργειες που να δίνουν την ευκαιρία να αυξηθεί η ορατότητα αυτού του ανθρωπιστικού προγράμματος. Εδώ μπαίνει το ερώτημα. Γιατί ο αριθμός αυτός υπήρξε τόσο μικρός, τόσο χαμηλό μέχρι τώρα. Εγώ έχω μια απάντηση. Λόγω του γεγονότος ήταν πολύ δύσκολο για όλες τις θελοντικές οργανώσεις της Ένωσης να καταγραφούν στους αρμόδιους οργανισμούς. Για παράδειγμα, στο ΕΚΟ, έχοντας υπόψη ότι υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων που εργάζονται όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι το πρόβλημα αυτό θα λυθεί όμω με την προβλεπόμενη διαδικασία. Τώρα κάποια άλλα πράγματα που με απασχολούν είναι η αποτελεσματικότητα του προγράμματος του European Solidarity Corps που πρέπει να στρέφεται σε συγκεκριμένους στόχους και συνοχή και να αποτελεί μέρος αυτό της νομικής βάσης. <clears throat> Επίσης, πρέπει να γίνεται αναφορά στους ε, στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Εδώ, στο πρόγραμμα αναφέρεται μόνο στο περιβάλλον. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, όμως, για την ανθρωπιστική βοήθεια σε φυσικές καταστροφές και θεομηνείς. Όμως, πρέπει να γίνεται αναφορά και σε δραστηριότητες των διαφόρων προγραμμάτων και συνοχή τους με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Προβλέπονται λιγότερες λεπτομέρειες από τον κανονισμό που έχει διατυπωθεί. Εμείς θα θέλαμε το σχετικό κεφάλαιο να είναι πιο συγκεκριμένο. Να αυξηθεί η ορατότητα του European Solidarity Corps και οι ευκαιρίες που προσφέρει σε νεαρούς Ευρωπαίους μέσω των κοινωνικών μέσων και με μια εκστρατεία ε, ενημέρωσης. Έχω και μια ερώτηση σχετικά με το όριο ηλικία που θέσατε προηγουμένως. Διότι στο παρελθόν όλοι οι εθελοντές στην Ευρώπη είχαν την ηλικία που έχει τώρα ο Μπερνάρ Κουσνέρ. Ίσως λίγο νεότεροι. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ανθρώπους με ηλικία άνω των 30 ετών από το να συμμετέχουν στο πρόγραμμα και μπορεί να έχουν και τη δυνατότητα να προσφέρουν υπηρεσίες στη βάση εκπαίδευση που έχουν. Πρέπει να το ξανασυζητήσουμε λοιπόν. Τώρα, υψηλή ποιότητα εκπαίδευση για του Ευρωπαίου εθελοντέ για ανθρωπιστική βοήθεια. Έχοντα υπόψη τι ανάγκε των νέων ανθρώπων στα διάφορα στρώματα της κοινωνίας, αλλά και τις επιτόπου ανάγκε για την προσφορά ανθρωπιστικής βοήθεια, τι ιδιαιτερότητε της ανθρωπιστικής βοήθειας και τι ιδιαιτερότητε των αναπτυσσόμενων χωρών. Θα επεκτείνουμε το πρόγραμμα και για υπερπόντια εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και την γειτονία τους. Σημαντική έμφαση στην ε, αποφυγή κοινωνικού αποκλεισμού υπέρ ευάλωτων ομάδων, προσφορά εκπαίδευσης για μη ε, κερδοσκοπικούς λόγους και έχω εδώ τώρα και μια άλλη ανησυχία σχετικά. Δεν θέλουμε δηλαδή να δημιουργήσουμε 100.000 νέες θέσεις απασχόλησης γιατί αλλιώς δεν θα μιλούμε για εθελοντικό σώμα. Για το λόγο αυτό πρέπει να μιλήσουμε λίγο παραπάνω. Τώρα, συμπεραίνοντας, για να εμφυσίσουμε στους νεαρούς Ευρωπαίους το πνεύμα του εθελοντισμού και να αναπτύξουν πνεύμα πρωτοβουλίας και να αναπτύξουν έργα για τις ντόπιε κοινωνίες τους, πρέπει να τους προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες, χωρίς διάκριση, με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες και στο ευάλωτο των τοπικών κοινοτήτων και να τους φέρουμε πιο κοντά στην επίτευξη μιας βιώσιμης ανάπτυξης και στην απαλήψη της φτώχειας. Η δική μου εμπειρία, κυρία Πρόεδρε, μου λέει ότι επί του παρόντος μόνο νεαροί δάσκαλοι και δασκάλες και κοινωνικοί λειτουργοί ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν δεν βλέπουμε νοσηλευτές, νοσηλεύτριες, μέες, γιατρούς να έρθουν να συμμετάσχουν. Αυτό λοιπόν είναι ένα σημείο όπου πρέπει να δουλέψουμε πολύ σκληρά για να του προσευχήσουμε και αυτού. Αναμένω με ενδιαφέρον τώρα τα σχόλιά σας και σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ Ελένη. Έχω κάποιους και οδησίτες. Σιόνφελτ, Γκερέρο, Άλλος κανείς επιθυμεί. Να λάβει το λόγο. Γιατί έχουμε και άλλο ένα θέμα. Σα έχω γράψει κύριε Σιόνφελτ. Δίνω το λόγο στον Σιόνφελτ λοιπόν. Παρακαλώ να είστε σύντομες, κάθετο σύντομοι, για να μην καθυστερήσουμε περισσότερο. Έχουμε άλλη μια έκθεση. E, e, e, Είναι αλήθεια ότι θα έχουμε ένα κανονισμό αλλά πριν να έχουμε το κειμένο νομοδότηση, είναι δύσκολο να πούμε κάτι συγκεκριμένο. Τώρα ξεκινήσαμε μια πρώτη συζήτηση με ανταλλαγή απόψεων, οπότε μπορούμε να συζητήσουμε έτσι γενικά και να εκφραστούμε, να τοποθετηθούμε γενικά. Εγώ νομίζω ότι όταν έχουμε μία νέα λύση που δεν είναι κάτι το απολύτως νέο, αλλά προέρχεται από υπάρχουσες πρακτικές, νομίζω το πιο σημαντικό είναι να κάνουμε μια καλή ανάλυση των δραστηριοτήτων που είχαμε μέχρι τώρα. Αν γνωρίζουμε και το ακούσαμε στην συζήτηση, αν γνωρίζουμε λοιπόν ότι η αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων μέχρι τώρα ήταν κάπως αμφίβολη, τότε νομίζω ότι αυτό αποτελεί ένα συναγερμό, ένα κόδωνα που μας προειδοποιεί σε σχέση με τα αποτελέσματα που θέλουμε να πετύχουμε. Γιατί νομίζω ότι δεν ασχοληθήκαν όλοι με την μελέτη αποτελεσματικότητα μέχρι τώρα. Γιατί αν τη είχαν όλοι κοιτάξει όλοι προσεκτικά, τότε θα μπορούσαμε ε, να κάνουμε και τα ίδια σφάλματα χωρίς πρόοδο. Και αυτό ακριβώς το λόγο θα ήθελα κυρίω να επικεντρωθούμε στι αναλύσει που έχουν γίνει, να τι μελετήσουμε στι αναλύσει που έχουν γίνει, να δούμε τα αποτελέσματα για να πάρουμε μια απάντηση στο ερώτημα. Γιατί δεν ήταν τόσο αποτελεσματικά όλα αυτά, γιατί ας πούμε το ενδιαφέρον των ατόμων, τα άτομα για τα οποία συζητάμε εδώ, οι νέοι ας πούμε, γιατί ναι δεν έδειξαν τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Όταν λοιπόν έχουμε την απάντηση στο ερώτημα αυτό το γιατί, τότε θα μπορούσαμε να βρούμε καλύτερες λύσεις ακριβώς για να αποφύγουμε τα λάθη του παρελθόντος. Πρώτο αυτό. Δεύτερο, εγώ διερωτώ με τι θέλουμε να πετύχουμε. Όχι τόσο εμείς, αλλά η Επιτροπή. Αλλά τέλο πάντων, α το πούμε στον πληθυντικό. Θέλουμε όλοι μας εδώ να δημιουργήσουμε μία δομή αποτελεσματική, τέλο πάντων δυναμική, η οποία στις διάφορες χώρες και εκεί που θα είναι απαραίτητο θα διαθέτει την ανθρωπιστική βοήθεια σε πιο υψηλό επίπεδο. Στην Ευρώπη λοιπόν θέλουμε να δημιουργήσουμε μία δομή, ή ένα σύστημα που θα είναι αποτελεσματικά ή θέλουμε αντίθετα να έχουμε κάποιες λύσεις μέσα των οποίων και ζητώ συγγνώμη έτσι που εκφράζομαι με αυτόν τον τρόπο λύσεις οι οποίες τέλος πάντων στην ουσία θα ανακυκλώσουν κόσμο. Είπε ο πρόεδρος Γιούνκερ ότι μέχρι το 2020 θα πρέπει να έχουμε 100.000 άτομα και μέχρι το τέλο του προγράμματο 405.000 ε, άτομα. Αλλά νομίζω στα προγράμματα δεν έχει σημασία η ποσότητα, η ποιότητα. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για βοήθεια προ άλλου συνανθρώπου. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε μια αποτελεσματική δομή ή θέλουμε να έχουμε κάτι το οποίο απλά και μόνο θα συνοδεύεται από ωραίε στατιστικές ιδιαίτερα όσον αφορά τον αριθμό των συμμετεχόντων. Μετά έχουμε και άλλα ερωτήματα που έχουν να κάνουν με τη γραφειοκρατία, α πούμε να θυμηθούμε ότι όταν έχουμε να κάνουμε μια εμπορική επαγγελματική δραστηριότητα, όταν υπάρχουν γραφειοκρατικοί τέλο πάντων φράγμα και εμπόδια, τότε ο κόσμος θέλει για διαφορούς λόγους να ξεπεράσει αυτά τα εμπόδια. Αντίθετα, όταν έχουμε μια εθελοντικού τύπου δραστηριότητα, η οποία δεν είναι αμοιβόμενη, όσο πιο πολλή γραφειοκρατία υπάρχει, τόσο περισσότερα εμπόδια υπάρχουν. Αν θέλει κάποιο δηλαδή να βοηθήσει, θέλει να κάνει μια εθελοντική δραστηριότητα κτλ. Όταν βλέπει ο κόσμος ότι υπάρχει τέλο πάντων ένα πάκο χαρτιά τα οποία θα πρέπει να συμπληρώσει και περίπλοκες διαδικασίες κτλ. Το βεβαίω χάνουν ενδιαφέρον και κίνητρο. Και αυτό ακριβώ το λόγο το σύστημα δεν λειτουργήσε τόσο σωστά, τόσο καλά μέχρι τώρα. Τώρα το να ενώσουμε το Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντισμού και την Υπηρεσία για τους Εθελοντές, να τα ενώσουμε όλα αυτά, θα μπορούσε να έχει ένα μόνο αποτέλεσμα. Ότι εντάξει, το τσάι θα είναι πιο γλυκό παιδί, θα ανακατεύουμε τη ζάχαρη αλλά θα είναι δύσκολο να γίνει μόνο με το ανακάτεμα πιο γλυκό το τσάι, έτσι, να το πω έτσι μεταφορικά. Οπότε, καταρχάς, θα πρέπει εμείς να επικεντρωθούμε στην ανάλυση αυτή που ανέφερα προηγουμένως για να συνάξουμε τα σωστά συμπεράσματα, για να μην επαναλάβουμε τα σφάλματα του παρελθόντος και να κοιτάξουμε προς το μέλλον. Και ένα τελευταίο σχόλιο, Πρόεδρε, για το όριο ηλικία. Είναι σημαντικό αυτό. Μιλάμε για στατιστικέ και αποτελεσματικότητα. Αν θέλουμε να πετύχουμε στατιστικά αποτελέσματα, α βάλουμε οποιαδήποτε ηλικία θέλουμε. Αν θέλουμε όμω να είμαστε αποτελεσματικοί, αν κάποιο θέλει να βοηθήσει, τότε θα πρέπει να απορρίπτουμε άτομα με εμπειρία. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αφιερώσει ώρες, μήνες και χρόνια από τη ζωή τους βοηθώντας τους συνανθρώπους. Οπότε δεν μπορούμε να τους αποκλείσουμε αυτούς τους ανθρώπους επειδή ας πούμε είναι πάνω άνω των 30. Αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε. Ευχαριστώ. Ο Ενρίκη, ευχαριστώ. Ενρίκη, σύντομα. Ναι, είναι πολύ σύντομα. Πράγματι, μέχρι να έχουμε συγκεκριμένη πρόταση στα χέρια μας, που θα υποβάλει η Επιτροπή Πολιτισμού, σε λίγες μέρες δηλαδή, είναι δύσκολο μέχρι τότε να έχουμε ξεκάθαρη θέση για κάποια συγκεκριμένα ζητήματα. Να κάνω δύο-τρία γενικά όμως σχόλια. Καταρχάς πιστεύω ότι όταν ο πρόεδρος της Κομισιόν, ο κ. Γιούνκερ, παρουσίασε το θέμα αυτό στην κατάσταση της Ένωσης το 2016 είχαμε αυτή την ιδέα κιν, κινητοποίησης κυρίως της νεολαίας όχι μόνο των νέων, της νεολαίας γενικότερα της Ευρώπης για μια δραστηριότητα συνεργασίας και εθελοντισμού με οργανωμένες μορφές εθελοντισμού στην κάθε χώρα ώστε να δώσουμε μια υφή, μια σφραγίδα ευρωπαϊκής αυτής της εθελοντικές δραστηριότητες. Αυτό αποτελούσε ένα κίνητρο. Κινητοποιούσε κόσμο. Όπως το Εράσμος δηλαδή, κάτι το οποίο κινητοποιεί νέους, κυρίως από την Ευρώπη, προς όφελος των συνανθρώπων. Και είναι αλήθεια τα στοιχεία που ακούσαμε σήμερα είναι μάλλον απεσιόδοξα. Αν δηλαδή κινητοποίησα μόνο 500 άτομα και τελικά πετύχαμε τα 175, αν το διαιρέσουμε αυτό με ε, τις 27 χώρες μέλη, το λέω αυτό υπέρ της Πρόεδρο, έτσι, τότε το, ο τελικός αριθμός είναι πραγματικά γελίος. Θα μπορούσε αυτό τώρα να αλλάξει με την ενσωμάτωση, το συνδυασμό των δύο αυτών σωμάτων που κάνουν θελοντική δουλειά. Μακάρι, μακάρι. Πάντως, από την σκοπιά της Κομισιόν Ανάπτυξης και τη δική μου την προσωπική για τα ανθρωπιστικά θέματα, αυτά που ακούσαμε είναι θετικά για την ανθρωπιστική βοήθεια. Δηλαδή, υπό την έννοια ότι οι δραστηριότητες κατάρτισης και τα προσόντα που θα πρέπει να έχει ένας εθελοντής για τα ανθρωπιστικά, όλα αυτά θα ληφθούν υπόψη όταν θα διαρθρωθεί, θα συγκροτηθεί ας πούμε αυτό το εθελοντικό σώμα. Έχω και κάποιες σοβαρές αμφιβολίες και εγώ για το όριο ηλικία των 30 ετών. Για διάφορους λόγους. Σε συγκεκριμένες ανθρωπιστικές κρίσεις το να είναι κανείς κάτω το 30 είναι απαραίτητα θετικό. Δεν είναι και τόσο θετικό. Γιατί πολλές φορές αυτές οι κρίσεις θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από συγκροτημένα άτομα με δυνατότητα να ασκήσουν κάποιο έλεγχο, με εμπειρία που χρειάζεται. Υπάρχουν λοιπόν διάφορα απαραίτητα στοιχεία που ιδιαίτερα όσον αφορά την ιδιαιτερότητα των ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων δεν συντείνουν στο να μειώσουμε την ηλικία, το όριο ηλικίας, γιατί υπάρχουν και άλλες πτυχές του εθελοντισμού που βεβαίως θα πρέπει να κινητοποιούν νέους και μάλιστα πολύ νέους. Όμως, όμως δεν, δεν θα έκλεινα αυτό, δεν θα το απέκλεια μάλλον αυτό το στοιχείο, ιδιαίτερα στην ανθρωπιστική βοήθεια. Ευχαριστώ. Να προσθέσω κι εγώ κάτι πριν δώσω το λόγο στην συγκεκριά. Νομίζω ότι ο Ενρίκε έχει δίκιο. Να αναρωτηθούμε ποιος είναι ο στόχος αυτού του προγράμματος, γιατί έχω αμφιβολίες Δηλαδή δεν θέλουμε να το κάνουμε. Φαίνεται ότι θέλουμε να το κάνουμε τέλο πάντων ένα πρόγραμμα νέων ώστε να αποκτήσουν εμπειρία. Δεν είναι αυτό το σωστό μήνυμα που θα έπρεπε να στείλουμε σε φτωχέ χώρε στον πλανήτη. Πήγαμε στην Κάνα την εβδομάδα. Η Αφρική, α πούμε, έχει εκατοντάδε χιλιάδε νέων ικανών ατόμων που μπορούν κάλλιστα να εργαστούν και θα μπορούσαν να αποφεληθούν από τι ευκαιρίε και την εκπαίδευση στι χώρε του. Οπότε ε, δεν είναι σωστό να στείλουμε του δικού μας νέου. Και στην ανθρωπιστική βοήθεια, στην ουσία, έχουμε να κάνουμε με άτομα που είναι έμπειροι. Γιατροί, νοσοκόμες, που μπορούν να βοηθήσουν αυτέ τις χώρες. Όχι να βοηθήσουμε αυτού που αναζητούν μια πρώτη εργασιακή έτσι, εμπειρία. Οπότε για το θέμα της ηλικία είναι δύσκολο πραγματικά όπως είπε και ο Ντρίκε, πολλοί ας πούμε που είναι μεγαλύτεροι μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικοί στην διαχείριση ανθρωπιστικών καταστάσεων. Ίσως λοιπόν εδώ ανακατεύουμε τα πράγματα. Δηλαδή ένα πράγμα για τους νέους, κάτι σαν το Εράσμου, στη στιγμή που θέλουμε κάτι διαφορετικό. Δεν έχουμε άλλο χρόνο σήμερα για συζήτηση, δεν θα δώσω το λόγο στην Κομισιόν, θα δώσω το λόγο μόνο στην Ελένη για να κλείσει στο κάλος. Αλλά θα πρέπει να το σκεφτούμε περισσότερο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς όσους συνεισέφεραν. Θα εξετάσω με μεγάλη προσοχή τις προτάσεις και θα επανέλθω. Να αναφερθώ σε τρία σημεία. Καταρχάς, δεν υπήρχε χαμηλό ενδιαφέρον μέχρι τώρα. Ήταν όμως δύσκολο οι νέοι να βρουν χρηματοδότηση. έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση σε μια ανθρωπιστική οργάνωση, να καταρτιστούν για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν στο πεδίο αργότερα. Είχαν δείξει όμως μεγάλο ενθουσιασμό συμμετοχής και συμφωνώ με τον κύριο Γκέρερο Σαλόμ εδώ όταν κάποιος θα χρησιμοποιηθεί σε πεδίο, θα πρέπει να είναι αρκετά όριμος. Και να μην αποτελεί μόνο ο ενθουσιασμός κίνητρο. Μιλάμε για το πώς να σώσει ζωές σε ορισμένες περιπτώσεις. Έπειτα. Το λέω σε όλους μας πρέπει να αποφύγουμε τη δημιουργία επαγγελματικού στρατού εθελοντών. Δεν θέλουμε επαγγελματίε εθελοντές. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα περιμένουμε λοιπόν την έκθεσή σας και τη συνεργασία με τους συναδέλφους στην ε, άλλη Περνάμε τώρα στο σημείο 12 το οποίο αφορά πάλι ένα νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό το νέο Πουδουπού. Ίντερεγ, Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, έχει να κάνει με διασυνοριακή συνεργασία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εξωτερική διάσταση, όμως που, περιλαμβάνει τις χώρες εταίρους, υπερπόντια εδάφη και χώρες και η Ελένη Θεοχάρου είναι η συγκίτρια και για αυτό το θέμα. Έχετε πολλά να πείτε σήμερα. Έχουμε μόνο 10 λεπτά γι' αυτό. Σας παρακαλώ να είστε σύντομοι. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, είχα δύσκολη μέρα σήμερα, είναι αλήθεια. Στόχος της ε, πρωτοβουλίας Interreg είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, κρατών σε τρίτη τρίτων χωρών ή υπερποντίων εδαφών. Αναμένεται η πρόταση αυτή κανονισμού για την περίοδο 2021-2027 να απλουστεύσει τη συνεργασία πέρα από τα σύνορα της Ένωσης. Παράλληλα, τα μελλοντικά χρηματοδοτικά μέσα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τα υπερπόντια εδάφη και χώρες έχουν στόχο να δημιουργήσουν σαφείς κανόνες έτσι ώστε να μεταφερθεί στο Interreg μέρος της χρηματοδότησης, καθώς δεν είναι νομικά εφικτό να δημιουργηθεί ένα ε, ταμείο εντός συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συγκεκριμένοι στόχοι αφορούν την καλύτερη διακυβέρνηση και περισσότερη ασφάλεια στην Ευρώπη. Η πρόταση αυτή εναρμονίζεται επίσης με τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, δηλαδή ε, πιο έξυπνη και πράσινη ανάπτυξη και οικονομία και Ευρώπη κοντά στους πολίτες. Καλωσορίζουμε με την πρόταση της Επιτροπής, θεωρούμε όμως ότι θα πρέπει να φαίνονται καλύτερα οι στόχοι της συνεργασίας. Οι προτάσεις μας επομένως εστιάζουν στα ακόλουθα. Όλα τα συστατικά στοιχεία του Ίντερεγκ θα συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και την απαλυφή της φτώχειας, όπως αναφέρεται ρητά στο άρθρο 108 της Συνθήκης της Λισαβόνας. Επίτευξη συνοχής σε όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές είναι κρίσιμη για τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Η στρατηγική για κάθε ένα από τα προγράμματα του Ίντερεκ θα πρέπει να δείχνει πώς το πρόγραμμα αυτό θα συνεισφέρει στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, όπως αυτοί αναφέρονται στην Ατζέντα 2030. Διασφάλιση ότι οι τρίτες χώρες, τα υπερπόντια εδάφη και χώρες θα, συμμετέχουν στο Ίντερεγ και οι ιδιαιτερότητες τους θα λαμβάνονται υπόψη. κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού των προγραμμάτων αυτών. Ο στόχος θα είναι η προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των χωρών και εδαφών αυτών και η σύσφυξη των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των χωρών αυτών και, στην, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς ε, ευημερία των χωρών αυτών. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει συνεισφορά στους ε, στόχους για το κλίμα στο πλαίσιο των διεθνών συμφωνιών όπως η COP21. Η διάσταση του φύλου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται επίσης σε όλα τα στατικά στοιχεία του Ίντερεγ, όπως και η απαλήφη της φτώχειας, η χρηστή διακυβέρνηση, η μείωση των ε, κινδύνων από καταστροφές και διαχείριση συνόρων, μετανάστευση και ασφάλεια μεταξύ άλλων. Προώθηση θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και μη κρατικών φορέων, πρόθεση της χρηστής διακυβέρνησης και καταπολέμηση της διαφθοράς. Κύριε Πρόεδρε, αναμένω σχόλια και σκέψεις τόσο από εσά όσο και από τους συναδέλφους. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ο κύριος Τσέλερ θα ήθελε το λόγο ως σκιώδης συζητητής και η Σεσίλ Κιέγγε. Δεν έχουμε χρόνο όμω, μην το ξεχνάτε. Στην ε, Περιφερειακή Επιτροπή μόλις συζητήσαμε το θέμα αυτό. Ενίσχυση δηλαδή των στατικών Interreg. Διότι στα πλαίσια του Interreg έχουμε μια πραγματική βάση για να συνεργαστούν διαμεθοριακά διάφορες περιφέρειες αλλά και θεσμοί. Ενώ μέχρι τώρα τα προγράμματα Interreg συνήθως είχαν μια, έναν εσωτερικό προσανατολισμό, δηλαδή μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι έχει έρθει ο καιρός πια να ξεκινήσει μάλιστα από τη δική μας Επιτροπή να δοθεί το μήνυμα ότι πρέπει να δραστηριοποιηθούν και διαμεθοριακά προς περιφέρειες εκτός Ευρώπης. Γι' αυτό όμως χρειαζόμαστε οπωσδήποτε την υποστήριξη και της Επιτροπής Αναπτύξεως με την έννοια ότι τα κονδύλια για τα προγράμματα Interreg δεν θα πρέπει να περικοπούν όπως προτείνει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θα πρέπει να διατηρηθούν το λιγότερο στο επίπεδο της τρέχουσας προγραμματικής περίοδου, ώστε το εργαλείο αυτό της εδαφικής συνεργασίας να αποδώσει και, στη, και στην ε, ε, διαπεριφερειακή. Ναι, ακόμα καλύτερα να ενισχυθούν τα κονδύλια. Εν πάση περιπτώσει χρειάζεται οπωσδήποτε διατήρηση των κονδυλίων και αν είναι δυνατόν να συνδεθούν και με την αναπτυξιακή συνεργασία ώστε και οι περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι θεσμοί οι οποίοι λειτουργούν στη βάση του Ίντερεκ να ενισχύσουν τη συνεργασία αυτή, να ενταχθούν ενισχυμένα στη συνεργασία αυτή. Αυτό θα αποδώσει θετικά αποτελέσματα. Δεν πρέπει να αφήσουμε την αναπτυξιακή συνεργασία μονάχα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή μόνο στι χώρε μέλη. Σα ευχαριστώ. Δύο λεπτά. Σε Κιέντια, σε παρακαλώ, μην ξεπεράσει τα δύο λεπτά. Λίντα, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την συνάδελφο Ελένη. Να υπογραμμίσω, όπως είπε και η συγκήτρια μας, ότι η Επιτροπή μας θα πρέπει να διασφαλίσει μια απλή πρόσβαση στην ενεργό δράση και σε τρίτες χώρες και στις υπερπόδιες χώρες στα πλαίσια του Interreg. Η δουλειά της συναδέλφου είναι ένα θαυμάσιο σημείο κίνηση και μπορούσα να εκτιμήσω πολλές από τις ε, προτάσεις της Ρέτζη. Νομίζω ότι θα συνεργαστούμε όλοι ώστε να συμπληρώσουμε το κείμενο γιατί το Interreg είναι από τα καλύτερα προγράμματα της Ένωσης ε, όπως το Erasmus Sin και αποτελεί μια καλή ευκαιρία για να αξιοποιήσουμε ακριβώς το αίσθημα ευρωπαϊκής υπηκότητας δίνοντας, προσφέροντας ε, στους πολίτες τρόπους συνάντησης ευρωπαϊκούς, ενισχύοντας βεβαίως την τοπικότητα και τη δυνατότητα χάραξης ε, προγραμμάτων που θα πρέπει να παραμείνει δική μας αρμοδιότητα και κυρίως όταν στις χώρες ε, μέλη βλέπουν να υπάρχει ένα αντίθετο ρεύμα με τα προγράμματα της κοινωνίας των πολιτών. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε την συνεργατική συνεργασία και προσωπικά Νομίζω ότι εμείς ως μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να προσέχουμε ώστε τα προγράμματα που αναπτύσσει το Ίντερεγ μέσω των εξωτερικών ταμείων χρηματοδότησης να είναι ε, να τηρούν μάλλον τις κατευθυντήριες γραμμές και θα πρέπει να δίδεται στην κοινωνία των πολιτών μια προστευμένη πρόσβαση σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για το μέλλον της Ένωσης και τους στόχους όπως βιωσμή ανάπτυξη, εξαλειψή στοχείας, καταπλέμιση ε, ε, κλιματικής αλλαγής, δηλαδή η Ατζέντα Θεματολόγιο 2030. Η πρόταση επικεντρώνεται στην προστασία των μειονοτήτων υπό όλες τις μορφές. Το Interreg στην Ένωση, στις χώρες εταίρους και στις χώρες της Ένωσης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τα πιο ευάλωτα άτομα και τις μειονότητες. Οπότε, χάρη στην συγγήτρια, θεωρώ θα κάνουμε μια πολύ καλή δουλειά. Ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελένη, έχετε ένα λεπτό αν θέλετε να ολοκληρώσετε. Δυστυχώ δεν υπάρχει χρόνο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λυπάμαι πολύ. Η διερμηνία θα σταματήσει στις 7 ακριβώ. Θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Ωραία, έτσι κι αλλιώ θα επανέλθουμε. 26 Οκτωβρίου η προθεσμία για τροπολογίε στι 12 το μεσημέρι. Συγγνώμη, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που δεν ε, λάβατε το λόγο. Θα ήθελα να ενημερώσω τους συναδέλφους ότι η επόμενη συνεδρίαση αύριο στις 9 το πρωί στο κτίριο 2Q2 θα έχουμε δημόσια ακρόαση και στη συνέχεια ψηφοφορία για το βραβείο Ζαχάροφ. Αύριο πρωί λοιπόν στην αίθουσα 2Q2. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστούμε τους διερμηνείς.